guten Morgen, liebe Καλημέρα συνάδελφε. Είναι πολλά τα έργα έξω από το Κοινοβούλιο και γι' αυτό λοιπόν και εγώ αλλά και άλλοι συνάδελφοι καθυστερήσαμε κάπως μία καθυστέρηση μικρή στα πλαίσια του Ακαδημαϊκού Τετάρτου βέβαια. Ας ε, ξεκινήσουμε όμως λοιπόν την συνεδρίαση της Επιτροπής Ελέγχου του Προπολογισμού. Θα ήθελα να σας καλωσορίσω όλους τρίτη φορά θα συναντιόμαστε αυτή την εβδομάδα. Να σας ρωτήσω αν συμφωνείτε και με την ημερήσια διάταξη. Δεν βλέπω να υπάρχει κάποια επιθυμία να γίνει κάποια αλλαγή. Εγκρίνεται λοιπόν η ημερήσια διάταξη. Και περνάμε λοιπόν στο 2 της ημερήσιας διάταξης. Να σας επισημάνω ότι είναι δημόσια η σημερινή μας συνεδρίαση. Μεταδίδεται στο διαδίκτυο. Και έχετε μπροστά σας και τις γλώσσες στις οποίες μπορείτε να παρακολουθήσετε τη συνεδρίαση για την ψηφοφορία. Αναβλήθηκε. Θα τοποθετηθώ ως προς αυτό αργότερα. Να σας πω ότι στις 7 Νοεμβρίου από τις 15 και 50 έως τις 16 και 10 σήμερα δηλαδή θα έχουμε συντακτική συνεδρίαση μια συνεδρίαση με την Επιτροπή Προϋπολογισμού Αυτά λοιπόν είναι τα σημεία τα οποία ήθελα να σας αναφέρω. Και έτσι μπορούμε να περάσουμε στο 3 της ημερήσιας διάταξης, στην ακρόαση των υποψήφιων μελών του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου. Και θα ήθελα καταρχάς να καλωσορίσω τον υποψήφιο που προτείνεται από τις ε, ελληνικές αρχές, ε, τον κύριο Νικόλα Μιλιώνη. Καλωσορίσατε στην ε, Επιτροπή μας. Σας αποστήλαμε ένα ερωτηματολόγιο και θα σας παρακαλούσα τώρα λοιπόν να κάνετε την πρώτη σας παρέμβαση πρωτού περάσουμε στη συζήτηση. Καλώς ορίσατε, έχετε το λόγο. Uh, good morning, uh, Mr. President. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα τοποθετηθώ στα αγγλικά, στις ερωτήσεις σας, στη συνέχεια, στα ελληνικά, τη μητρική μου γλώσσα. Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε, μέλη της Επιτροπής της, του ελέγχου του προπολογισμού. Ιδιαίτερη τιμή που αισθάνομαι, βρίσκομαι οποίο σα σήμερα, ελπίζοντα ότι θα δώσετε θετική γνώμη για την, το διορισμό μου ω μέλου του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου. Η θετική σα γνώμη θα επιβιώσει την ε, πίστη σας ε, στην ανεξαρτησία και τις επαγγελματικέ μου ικανότητες και θα αποτελέσει την απαρχή ενός θεσμικού διαλόγου και συνεργασίας. Προέρχομαι από μια μικρή πόλη της Δυτικής Ελλάδας, γεωργική οικογένεια, η οποία με ανέθρεψε με τις αξίες της ε, εντιμότητας, της επιμέλειας και της ταπεινοφροσύνης. Ε, ολοκλήρωσα τις σπουδές μου, ε, το σχολείο δηλαδή, στην πατρίδα μου και σπούδασα νομική στο Πανεπιστήμιο των Αθηνών με υποτροφία. Στη συνέχεια πέρασα τις εξετάσεις της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και ε, έγινα μέλος του ελεγκτικού συνεδρίου της πατρίδας μου ως δικαστής. Είχα την καλή τύχη δε να ε, μελετήσω ιδιαίτερως το δημόσιο δίκαιο και τις, ε, τα, δημοσιονομικά και, και απόδοση λογαριασμών στο Πανεπιστήμιο του Παρισιού, όπου επίσης παρακολούθησα μια σειρά διασκέψεων του Γαλλικού Ελεκτικού Συνεδρίου, του Κοντεκόντ, όπου και αργότερα εργάστηκα ως ε, βοηθός. Αυτές οι εμπειρίες μου λοιπόν με βοηθούν ιδιαίτερα να αντιλαμβάνομαι πόσο σημαντική είναι η διεθνή συνεργασία. Μου προσφέρουν επίσης ε, βάση έρευνας για τη θεωρία του ε, δημόσιου οικονομικού δικαίου. Η εμπειρία μου επίσης από την εκπαίδευση μου επέτρεψε να προσφέρω βοήθεια ως μέλος σε επιτροπές για το σχεδιασμό του ε, συστήματος δημοσιονομικού ελέγχου στην πατρίδα μου. Ταυτόχρονα καλλιέργησα τα ενδιαφέροντά μου στην ζωγραφική και τη λογοτεχνία. Δραστηριότητες οι οποίες μου δίνουν τη δυνατότητα, την ικανότητα, την επιστήμη μου, το επάγγελμά μου να τα δω μέσα από ένα πιο ανθρώπινο πρίσμα και να καταλαβαίνω τα προβλήματα της κοινωνίας και της ε, αγωνίας του ανθρώπου πίσω από τα νούμερα, τις στατιστικές και τα γραφήματα. Έχω πλήρη πεποίθηση ότι το Ευρωπαϊκό Ελεκτικό Συνέδριο η δημοσιονομική δηλαδή συνείδηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορεί να φέρει τη δική του επίδραση και με τα μέσα και τα, με μέσω του μηνύματος που αποστέλει. Οι ευθύνε που αναλαμβάνει, η μέθοδη του δημοσιονομικού ελέγχου οι εκθέσεις και οι γνωμοδοτήσεις που αφορούν την εκτέλεση του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού είναι αποτελεσματικά μέσα για τη ασφάλιση των δημοσίων οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με τους ελέγχους του το Ευρωπαϊκό Ελεκτικό Συνέδριο δίνει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ανεξάρτητη, αντικειμενική και αξιόπιστη πληροφόρηση που του επιτρέπει να εξετάζει την ε, εκτέλεση του ευρωπαϊκού ε, προϋπολογισμού. Έτσι λοιπόν είναι θεσμικός εταίρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου το Ελεκτικό Συνέδριο δίνει πολύτιμη συνδρομή ως προς τη, με τη διαδικασία της απαλλαγής, επιβεβαιώνοντας ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εκτελέσει όπως οφείλει τις δημοσιονομικές της ευθύνες. Ως μέλλον μέλος του Ευρωπαϊκού Ελεκτικού Συνεδρίου, όπως ελπίζω, θα καταβάλω κάθε δυνατή προσπάθεια να εξασφαλίσω πως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Επιτροπή ενημερώνονται για, τις, για τα ευρήματα και οι Επιτροπή σα ενημερώνονται για τα ευρήματα του ελεγκτικού συνεδρίου μέσα σε ένα διάλογο επικοδομητικό και σε πνεύμα ανοιχτή αντιπαράθεσης, ανοιχτή συνεργασίας. Γνωρίζω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το ένα σκέλος τη Μοσυνομική Αρχής αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στη συνεργασία με το ελεκτικό συνέδριο και ιδιαίτερα την εφαρμογή και τη αξιολόγηση των δημοσιονομικών επιδόσεων των δραστηριοτήτων τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίση, γνωρίζω ότι συνεχίζονται οι προσπάθειέ σα για να συμβάλλετε με νέε ιδέε και καλύτερη οργάνωση και λειτουργία του Ευρωπαϊκού Ελεκτικού Συνεδρίου. Βρίσκομαι λοιπόν ενώπιον σα με έναν ευρύ ορίζοντα μπροστά μου που θα μου επιτρέψει πιστεύω να εφαρμόσω οτιδήποτε έχω μελετήσει, γράψει, διδάξει και συλλέξιους εμπειρία όλα αυτά τα χρόνια. Εάν μου δώσετε την ε, θετική σας νομοδότηση για το διορισμό μου θα εργαστώ ε, με επιμέλεια για να συμβάλλω σε συνεργασία με τους συναδέλφους μου και φυσικά μαζί σας στη βελτίωση του θεσμικού ρόλου του ελεκτικού συνεδρίου ως τον οφθαλμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την εκτέλεση του Ευρωπαϊκού Προϋπολογισμού, την προστασία των μεσονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή όλων ημών. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ πολύ για την εξέταση της υποψηφιότητά μου. Ευχαριστώ κύριε Μιλιώνη. κύριε και κύριοι, θα παρακαλέσω τώρα να λάβετε εσείς το λόγο για να διατυπώσετε τις ερωτήσεις σας για την προτινόμενη υποψηφιότητα στον κύριο Μιλιώνη. Η συγγήτρια παρακαλώ, κυρία Γιάννα Ζέντερ. Sí, Λυπάμαι που καθυστέρησα. Είχε πάρα πολλή κίνηση. Και ξέρετε, έχουμε πολλές δραστηριότητε πάντα ως πολιτική. Θα ήθελα να καλωσορίσω τον κύριο Μιλιώνη ως υποψήφιο για το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο. Θα ήθελα να του διευκρινίσω ότι το βιογραφικό του είναι πάρα πολύ ε, ενδιαφέρον και εντυπωσιακό. Και σίγουρα έχει πάρα πολλές ικανότητες να προσφέρει. Θα εξετάζουμε λοιπόν πάντα ποιες είναι οι εμπειρίες των υποψηφίων στα εθνικά τους πλαίσια. Και γι' αυτό δεν θα σας προκαλέσει έκπληξη το σας ε, ρωτώ το εξής. Ε, τα τελευταία χρόνια στο ελληνικό ελεγκτικό συνέδριο βλέπω ότι συμμετείχατε και θα ξέρετε ασφαλώς ότι η Ελλάδα ε, αντιμετωπίζει ιδιαίτερες συνθήκες τα τελευταία χρόνια. Αυτό ισχύει και για την Ισπανία, ξέρετε. Η γενική κρίση που πλήττει την Ευρώπη έχει πλήξει ιδιαίτερο στα δημοσιονομικά της Ελλάδας και την σχέση μεταξύ δαπανών και εσόδων στη χώρα σας. Γι' αυτό λοιπόν ερωτώ. Οι σημαντικές αποφάσεις ε, τις οποίες ε, έχετε λάβει ως μέλος του Ελληνικού Ελεκτικού Συνεδρίου. Πείτε μας ήταν η συνδρομή σας στο ελληνικό ελεγκτικό συνέδριο χρήσιμη, ωφέλιμη για να αντιμετωπιστούν τα ζητήματα αυτά σε ό,τι αφορά τα προβλήματα των ελληνικών δημοσιονομικών. Πώς συμβάλλατε εσείς. Για το σημείο 8 τώρα η επόμενη ερώτηση. Μιλάτε για ένα μακρύ κατάλογο σε ό,τι αφορά τις ε, δημόσιες υπηρεσίες και αυτά που θα πρέπει να συμβάλλουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Γι' αυτό λοιπόν σας ερωτώ. Θεωρείτε ότι από πλευράς δημοσιονομικών το θέμα είναι να διαμορφωθεί μια πιο αποδοτική κατάσταση που να εξυπηρετεί καλύτερα το σκοπό της. Αυτό είναι ενδιαφέρον. Αυτό αποτελεί ένα από τα βασικά στοιχεία της δραστηριότητά σας. Παρακαλώ αναπτύξτε το αυτό. Και πολύ ε, ενδιαφέρουσα η δημοσίευση για το ε, τρόπο που γίνεται ο έλεγχος από πλευράς του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου. Ένα κείμενο του 1998 και ένα κείμενο του 2012 όπου αναφέρεται οι εγγυήσει που προβλέπονται από τον κανονισμό σε ό,τι αφορά το Ευρωπαϊκό Ελεκτικό Συνέδριο. Αυτό είναι πολύ ενδιαφέροντα και σε ό,τι αφορά τον Όλαφ. Θα ήθελα να ακούσω πιο πολλά για αυτό το θέμα. Ευχαριστώ. Άλλε ερωτήσει υπάρχουν, παρακαλώ. Όχι προ το παρόν. Α ακούσουμε τότε την απάντηση. Όχι, ο κύριο Μπελσίτη. Ο κύριο Μίλτερ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και εγώ ήθελα να πω ότι είναι πολύ εντυπωσιακό το βιογραφικό σας. Έχω μια ερώτηση πάντως. Στην Ελλάδα για χρόνια υπήρξε πρόβλημα στον έλεγχο των γεωργικών επιδοτήσεων. Ενώ ήταν το σύστημα στηριγμένο στις πληρωμές ανά εκτάριο, στην επιφάνεια δηλαδή της γεωργικής ε, γης, δεν υπήρχε εκτιματολόγιο. Πώς μπορείτε λοιπόν να κάνετε επαλήθευση όταν δεν υπάρχει επαρκέ σύστημα εκτιματολογίου. Μπορείτε να μας πείτε ποια είναι η κατάσταση τώρα και αν έχει βελτιωθεί. Και επίσης πώς βλέπετε εσείς ως το ψήφιο μέλος αυτή την κατάσταση. Σας ευχαριστώ, ο συνάδελφος Βοντή και μετά ο κύριος Μπαλτσίτης. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εκ μέρου τη ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματο, θα ήθελα και εγώ να σα καλωσορίσω κύριε Μιλιώνη. Να σα ευχαριστήσω για τι διευκρινήσει που μα δώσατε. Για είναι μέλο κανεί του Ελεκτικού Συνεδρίου, του Ευρωπαϊκού Ελεκτικού Συνεδρίου, θα πρέπει να πληρεί δύο όρους. Πρώτον, να έχει επαρκή γνώση προς το δημοσιονομικό έλεγχο και δεύτερον, να πληρεί κανόνες δεοντολογίας και κυρίως ανεξαρτησίας. Στα τεχνικό σκέλος έχετε ένα εντυπωσιακό φάκελο υποβάλλει, έχετε πολύ ε, μεγάλη εμπειρία ως δημοσιονομικός ελεγκτής. Νομίζω ότι ικανοποιούν τα όσα βλέπουμε, τους όρους που ζητεί η Επιτροπή του Ελέγχου του Προϋπολογισμού, αλλά όσον αφορά τους ελέγχους, ε, τους δημόσιου, τους μεσονομικούς ελέγχους στην Ελλάδα, αυτό ήταν και μέλος του ελεγκτικού συνεδρίου εκεί, έχουμε δει πολλές διαρροές στον τύπο που λένε ότι ήταν ε, φαρκιδευμένοι αυτοί οι λογαριασμοί που παρουσίαζαν οι ελληνικές αρχές. Ε, εσείς ως μέλος του ελεγκτικού συνεδρίου έχετε δει ένα τέτοιο φαινόμενο, έχετε διαπιστώσει αλλίωση λογαριασμών, είχατε τη δυνατότητα με τεχνικό τρόπο από την τεχνογνωσία και την εξειδίκευση σας να πείτε, να διαπιστώσετε αν ήταν εσφαλμένοι λογαριασμοί ή όχι. Γιατί ε, μαθαίνουμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε στηριχθεί σε στατιστικές και όχι σε ε, λογαριασμούς, ε, απόδοση λογαριασμών από το, ευρωπαϊκό, από το ελληνικό δημόσιο, γιατί ακριβώς εκεί υπήρχε το πρόβλημα. Τι έχετε να μας πείτε γι' αυτό. Και η δεύτερη ερώτηση που έχει να κάνει με την ανεξαρτησία σας. Δίνετε το ιστορικό σας, το βιογραφικό σας, εξηγείτε ότι έχετε διδαχθεί, έχετε ανατραφεί με τις αρχές της ε, ταπεινοφροσύνης και θα ήθελα να ρωτήσω αν αισθάνεστε πραγματικά ανεξάρτητος έναντι της ελληνικής κυβερνήσεως, γιατί ως μέλος του ελεγκτικού συνεδρίου θα χρειαστεί να λάβετε θέσεις οι οποίες μπορεί να φέρουν σε δύσκολη θέση στην κυβερνήση αυτή. Ε, πώς μπορείτε λοιπόν να, να μας καθησυχάσετε, να μας διαβεβαιώσετε ότι άπαξ και διοριστείτε θα είσαστε το όντι ανεξάρτητος έναντι της ελληνικής κυβερνήσεως. Ευχαριστώ. ευχαριστώ κύριε Μπαλτσίτη. είναι επόμενο. Ευχαριστώ πρόεδρε. Αγαπητέ κύριε υποψήφια, η δική μου ερώτηση είναι κάπως διαφορετική από αυτές των συναδέλφων. Οι εμπειρίες σας και τα επαγγελματικά σας προσόντα δεν επιτρέπουν οποιοδήποτε περιθώριο αμφιβολίας. Κάθε υποψήφιος εξαρτάται από την εθνική κυβέρνηση σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό. Είναι αναπόφευκτο. Ε, ρωτώ λοιπόν κάτι διαφορετικό. Γιατί προσπαθείτε να γίνετε μέλος του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου. Η μεγαλυτερο βαθμο ειναι αναποφευκτο εκεί είναι τεχνικής φύσεως και δεν θα είσαστε σε θέση να εκπληρώσετε τις προσωπικές σας φιλοδοξίες. Μιλάμε για υψηλόβαθμες θέσεις. Είχατε πολύ υψηλόβαθμες θέσεις σε εθνικό επίπεδο. Τελευταίος, ο κ. Σταυρακάκης. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Μιλιώνη, σας καλωσορίζω και εγώ με τη σειρά μου στην Επιτροπή μας. Ε, έχω διαβάσει στη ζωή μου, λόγω της επιστημονικής μου ιδιότητας, πάρα πολλά βιογραφικά και ειλικρινά σας λέω ότι απόλαυσα το βιογραφικό σας διαβάζοντα το με πολύ μεγάλη προσοχή όσον αφορά τις σπουδέ σα, την επαγγελματική πείρα, την διδακτική εμπειρία που έχετε και γενικά όλη σας την δραστηριότητα στο ελληνικό Ελεκτρικό συνέδριο. Ε, πραγματικά πιστεύω ότι είστε ο σωστό άνθρωπο στη σωστή θέση. Πείτε μου όμως, σας παρακαλώ, πόσο πραγματικά ανεξάρτητος και δίκαιος θα είστε όσον αφορά την χώρα μας και ιδιαίτερα σε ευαίσθητους τομείς που κατά καιρού σχεδόν κάθε χρόνο το, η ετήσια έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεκτικού Συνεδρίου ε, στον τομέα της πολιτικής συνοχής, στην περιφερειακή ανάπτυξη, τα ποσοστά λάθους στη χώρα μας είναι σχετικά υψηλά. Σας ευχαριστώ και, και πάλι σας καλωσορίζω. Σας ευχαριστώ. Ακούσαμε διάφορες ερωτήσεις. Κύριε Μιλιών, έχετε το λόγο για να απαντήσετε. στην... Ε, ευχαριστώ πολύ για τις ερωτήσεις, ευχαριστώ πολύ για τα καλά σας λόγια. Ε, στην πρώτη ερώτηση της κυρίας εισηγήτριας, της κυρίας Αγιάλα Σέντερ, ε, κατά πόσον συνέβαλα σε αυτά τα οποία λέγω σε ό,τι αφορά τις αλλαγές που έγιναν στο ελληνικό ελεγκτικό συνέδριο, θα αρχίσω από το εύκολο σε ό,τι αφορά τα έσοδα, πραγματικά εκεί η δουλειά μου ήταν τυπική, διότι όλοι γνώριζαν την ανάγκη δημιουργίας ενός θεσμικού πλαισίου για να υπάρξει δυνατότητα ε, εισρωών στον προϋπολογισμό. Γιατί πράγματι ο προϋπολογισμός σε ό,τι αφορά αυτό το ζήτημα ήταν χολός. Δεν λειτουργούσε σωστά. Το δύσκολο ήταν σε ό,τι αφορά τον περιορισμό του προληπτικού ελέγχου. Εμείς είμαστε οι τελευταίοι, όχι ίσως οι τελευταίοι, οι τελευταίοι στην Ευρώπη που κάνουμε προληπτικό έλεγχο των δαπανών. Είναι μια ε, παρμοδιότητα περίπου 150 ετών. Το ελεγκτικό συνέδριο θεσπίστηκε, στηρίχτηκε στον προληπτικό έλεγχο αφήνοντας κατά μέρος τους κατασταλτικούς ελέγχους και λοιπά και τους ελέγχους διαχείρισης στηρίχθηκε εκεί γιατί καταλάβαινε πως υπάρχει ένα πρόβλημα στην ελληνική δημόσια διοίκηση, ε, πρόβλημα δομικό. Λοιπόν, και γι' αυτό θεωρούσε πως ο προληπτικό, η προληπτική έλεγχη είναι ε, η σοβαρή έλεγχη που θα μπορούσε να κάνει σε μια χώρα σαν την Ελλάδα. Μέσα στην κρίση όμως ε, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο μας υπέδειξε πως πρέπει να περιοριστούν οι έλεγχοι αυτοί. Όμως υπήρχε σχετική συνταγματική διάταξη η οποία μας το απαγόρευε. Εκεί η συμβολή μου πραγματικά τόσο στο, στη φάση της κατάρτισης του νόμου, του νόμου του 2010, όσο <coughs> και στην έκδοση του Προεδρικού Διατάγματος ήταν πραγματικά δύσκολη. Να, γιατί ε, μιλάμε πως έπρεπε να ε, αντιλήψεις πολλών ετών. Ε, σε ό,τι αφορά τα έσοδα, απάντησα, προσπάθησα να απαντήσω και σε ό,τι αφορά τα έσοδα, όπως είπατε, και σε ό,τι αφορά τις δαπάνες. Ε, πραγματικά, στο σημείο 8 μιλάμε για την αποδοτικότητα. Ε, η αν, δεν υπάρχει δημόσια... αν δεν υπάρχει απόδοση, αν δεν υπάρχουν στόχοι να τεθούν και να ελοποιηθούν, δεν μπορούμε να μετρήσουμε για απόδοση. Στην Ελλάδα έχουμε... είχαμε... είχαμε το πρόβλημα αυτό μέχρι τη δεκαετία του 90 ε, δεν ξέραμε τι είναι αποδοτικότητα, δεν ήμασταν οι μόνοι βέβαια, αλλά οι άλλοι δυστυχώς για μας προχώρησαν πάρα πολύ γρήγορα. Εμείς μείναμε πίσω, σε παλαιωμένες αντιλήψεις. Λοιπόν, στην αποδοτικότητα άρχισε πρώτα να γίνεται «evaluation de politique publique», όπως λένε οι Γάλλοι. Άρχισαν δηλαδή πρώτα η δημόσια, η δημόσια διοίκηση να υιοθετεί ε, τουλάχιστον στα χαρτιά, στο νόμο, το ζήτημα της αξιολόγησης. Δεν το προχώρησε. Σε ό,τι αφορά την, ε, την, το performance audit μετά, δηλαδή το να κάνουμε αξιο, ε, έλεγχο επί των αξιολογήσεων που κάνει ο διατάκτης, που κάνει η διοίκηση, ε, ήρθε τώρα τελευταία το 10 και μάλιστα με, το, ε, με καθυπόδειξη του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Ε, σε ό,τι αφορά τα κείμενα του 98, αν θυμάμαι καλά, είναι που λέει για το European Style of Audit και του 12 είναι για ε, τον έλεγχο ε, της, αυτό που λένε οι Γάλλοι ε, ε nouvelle gouvernance, η νέα, διακυβέρνηση. Η νέα διακυβέρνηση. Πραγματικά το, το κείμενο του 1998 ήταν ένα κείμενο που απηχούσε την εμπειρία μου στο Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο. Σήμερα βέβαια μοιάζει υπαρχιωμένο, διότι το Ελεγκτικό Συνέδριο στις αρμοδιότητες του ανοίχτηκε πάρα πολύ, εισήγαγε καινούργια πράγματα, εισήγαγε και εφάρμοσε σε μεγάλη έκταση το performance audit που τότε δεν ήταν, ήταν στα σπάργανα ακόμη. Ε, σε ό,τι αφορά το, το κείμενο του 12, αυτό ε, είναι ένα κείμενο που απηχεί την εισαγωγή και στην Ελλάδα του performance audit, την, ε, των αξιολογήσεων των δημόσιων πολιτικών κλπ. Ε, στην δεύτερη ε, ερώτηση για τις γεωργικές δαπάνες ε, πραγματικά στην Ελλάδα το ζήτημα των γεωργικών επιδοτήσεων είναι ένα πρόβλημα με πληγές παλαιές και σύγχρονες. Παλαιές διότι οι γεωργικές επιδοτήσεις είχαν εκ μέρους ε, του, της Ευρωπαϊκής Ένωσης είχαν τύχει μια κακής διαχείρισης σε μεγάλη έκταση, σε μεγάλη έκταση, τα σκάνδαλα ήταν τρομακτικά. Ε, απ' την άλλη, όντως, δεν υπάρχει αυτή η δομή δηλαδή το κτηματολόγιο. Το κτηματολόγιο ξέρετε πως κάποια στιγμή πάλι με, ε, στις αρχές του 2000, στα μέσα της δεκαετίας του 2000, ε, είχε προχωρήσει αλλά πάλι έπεσε σε σκάνδαλα ε, με την κτηματολόγιο, μια ανώνυμη εταιρεία με το όνομα κτηματολόγιο και σταμάτησε. Τώρα το πράγμα έχει προχωρήσει, τυχαίνει επειδή προείδρευα σε μια σε ένα, σχηματισμό του ελεγκτικού συνεδρίου που εκεί περνούσαν τα σχέδια των συμβάσεων, ε, σχέδια συμβάσεων δημοσίων υπηρεσιών, έτυχε να περάσουμε και του, ε, το σχέδιο συμβάσεως, τα επιμέρους σχέδια συμβάσεων για το, για το κτηματολόγιο. Ε, ελπίζω τα πράγματα, ε, εμείς τουλάχιστον προχωρήσαμε το πράγμα και το κτηματολόγιο. Βέβαια, επειδή στο κτηματολόγιο τα συμφέροντα των ιδιωτών είναι πολύ ισχυρά, κυρίως των τοπογράφων και των επιχειρήσεων αυτών, ε, τώρα τα πράγματα είναι στα διοικητικά δικαστήρια. Υπάρχει ένα έντονο, μια έντονη ε, ε πώς το διάσταση απόψεων και έφτασε στα δικαστήρια. Ε, σε ό,τι αφορά την, τις, ε, ερωτήσεις του κυρίου Οντί. Ε, ευχαριστώ πολύ για το καταρχάς για τα καλά λόγια. Ε, πραγματικά σε ό,τι αφορά την δεοντολογία και την ε, ανεξαρτησία μου ε, βέβαια υπάρχει το τυπικό γεγονός πως είμαι δικαστής και τυπικός είμαι ανεξάρτητος. Το ζήτημα της ε, του ουσιαστικού μέρους αυτού είναι ζήτημα το οποίο είναι η φήμη που έχει κανείς στο δικαστήριό του και κατά πόσον μπορεί να τα βάλει πέρα με αποφάσεις της κυβέρνησης. Όπως θα είδατε στο βιογραφικό μου έτυχε να είμαι πρόεδρος, ε, σε, ε, όχι πρόεδρος, προείδρευα σαν αρχαιότερος σύμβουλος σε ένα τμήμα που είχε πολύ σημαντικές υποθέσεις με πρώην υπουργού, ε, πολύ ισχυρούς σχεδόν πρωθυπουργούς κάποια στιγμή της χώρας μου και με άλλους υπουργούς και, τώρα και με πολύ δυνατούς δημοσιογράφους μπόρεσα και τα έφερα εις πέρας. Η φήμη μου υπάρχει στο, στο ελληνικό ελεγκτικό συνέδριο ε, για την ανεξαρτησία μου. Ε, σε κάθε περίπτωση το ελεγκτικό συνέδριο επειδή είναι μια θεσμική αντιπολίτευση όπως λέει η, η θεωρία. είμαστε θεσμικός αντιπολιτευόμενη την κυβέρνηση. Είναι το, το σύνταγμα μας το λέει και η φύση της δουλειά μας. Είμαστε εκ των πραγμάτων ανεξάρτητοι. Όχι πως δεν γίνονται απόπειρε για να φαλκιδευτεί αυτή η ανεξαρτησία. Το ζήτημα είναι δικό μας, κατά πόσον αυτό εμείς το κάνουμε τρόπο ζωής στην ανεξαρτησία μας. Ε, για την φαλκίδευση των λογαριασμών που είπατε, θα σας πω ένα παράδειγμα. Πραγματικά έχουν φτάσει ε, στα, και στον τύπο έχει φτάσει πως ε, ε, πολλοί λογαριασμοί ενώ καταλαβαίναμε πως υπήρχαν αποδείξεις πια πως, δηλαδή στον κατασταλτικό έλεγχο βλέπαμε πως υπήρχε, υπήρχε διαφθορά υπήρχαν κοινοτικέ δαπάνες που ο αρμόδιος διαχειριστής έβαζε και τους συγγενείς του μέσα. Λοιπόν, εκεί επειδή αυτές οι υποθέσεις είχαν περάσει από τον προληπτικό έλεγχο, γιατί σας είπα πως εμείς έχουμε και ένα άλλο είδος ελέγχου, λίγο παλαιωμένο, αλλά τουλάχιστον αποδοτικό προς το παρόν, ε, και επειδή επρόκειτο για μια αντίληψη, για μια νομολογία 150 ετών, πως αν περάσει από τον προληπτικό έλεγχο δεν μπορεί να ελεγχθεί στον κατασταλτικό, να όμως που βρέθηκε στον κατασταλτικό έλεγχο η, η διαφθορά. Εκεί προσπαθήσαμε να ανατρέψουμε μια νομολογία 150 ετών και το καταφέραμε και το καταφέραμε. Αυτό το μπαράζ το διαρρήξαμε. Ε, στην ερώτηση γιατί πραγματικά θέλω να γίνω. Ε, ε, θα εννοείται βέβαια γιατί έχω και τις άλλες παράλληλες αρμοδιότητες. Πάντα τις είχα αυτές. Ε, αυτές πάντα νομίζω πως μου γονιμοποιούσαν τη σκέψη οι άλλες. ξέρω πως είναι ένα πολύ σημαντικό, ε, ένα σημαντικό λειτουργήμα αυτό του μέλους του ελληνικού συνεδρίου. Αλλά θεωρώ πως πάντα θα βλέπω τις εκθέσεις μου, πάντα θα διαβάζω τη λογοτεχνία μου. Το βράδυ πριν κοιμηθώ έτσι κάνω και τώρα εξάλλου. Ε, δεν είναι ζήτημα. Ε, για ποιο λόγο, επειδή είναι ζητήματα τεχνικής φύσης, ε, λοιπόν αυτά τα ζητήματα τεχνικής φύσης χρειάζονται κάποια, δροσιά. Νομίζω αλλιώς <laughs> αποξηραίνεται κανείς. Ε, γιατί θέλω να γίνω, ε, ξέρετε αυτό, γιατί θέλω να γίνω μέλος του ελεγκτικού συνεδρίου. Διότι όταν ήμουν πριν, 20 χρόνια έτυχε να, να είχα την τύχη ε, να, να, να πάω για λίγο, για δύο χρόνια, ε, στο, στο καμπινέ του Έλληνα μέλους. Λοιπόν, αυτή η συμπάθεια έγινε έρωτας με τα χρόνια και ε, είμαι μπροστά σας για να εκπληρωθεί ο έρωτας αυτός. Ε, για τον κύριο Σταυρακάκη ε, και πάλι ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια κύριε Σταυρακάκη ε, όντως η, η, η ετήσια έκθεση του ελεγκτικού συνεδρίου μας στοχοθετεί πολλές φορές. Δεν είμαστε οι μόνοι, ίσως είμαστε οι πιο αδύναμοι να αντικρούσουμε τις κατηγορίες. Δεν, δεν αντιλέγω πως έχουμε μέτωπα ανοιχτά πάρα πολλά πάρα πολλά και με το σαν, σαν εθνική ε, κυβέρνηση, δηλαδή σαν διαχείριση δηλαδή εθνική και με το ελληνικό ελεγκτικό συνέδριο και με το ευρωπαϊκό ελεγκτικό συνέδριο. Θα πρέπει να μάθουμε με τα λάθη μας, να τα θεραπεύσουμε τα λάθη μας. Ευχαριστώ πολύ. Ja, vielen Dank. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Μιλιώνη. Και τώρα η κυρία Γκρέσλε θα θέσει τα επόμενα ερωτήματα. Σα Σας ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να μιλήσω εξ ονόματός μου. Έχω ένα πρόβλημα με την υποψηφιότητά σας κύριε Μιλιώνη, δεν σας γνωρίζω, αλλά με ανησυχεί ιδιαίτερα γιατί ήσασταν πρόεδρος του Εκτικού Συνεδρίου, ε, σε όλες τις αποφάσεις που λήφθησαν και τελικά αποδείχθησαν λαθασμένες, ε, ήσασταν μαζί κι εσείς. Δεν ξέρω λοιπόν την, πώς να σας εκτιμήσω ως ε, άτομο προσωπικότητα, γιατί εδώ είμαστε υπεύθυνοι ενώπιον του Ευρωπαίου πολίτη, του Ευρωπαίου Ευρωλογόμενου. Θέλω να βγω και να πω στον Ευρωπαίο πολίτη ότι εμείς δεν κάναμε λάθη. Και πείτε μου, σε ό,τι αφορά τα προβλήματα των ελληνικών δημοσιονομικών. Τι κάνατε εσείς. Ε, ήμασταν ε, δύο φορές επισκεφτήκαμε με την Επιτροπή μας το 2007 και το 2010 ε, την Ελλάδα στο follow-up και το 2010 για τις αγροτικές δαπάνες. Δεν ξέρω κατά πόσο κάποιος από τους συναδέλφους ήταν και αυτός μαζί. Το 2007 λοιπόν επισκεφτήκαμε και το 2010 το Ελληνικό Ελεκτικό Συνέδριο και είδαμε λοιπόν τι γινόταν. Ήσασταν κι εσείς μια φορά νομίζω εκεί και είδαμε ότι ήταν απρόθυμο να διδραματίσει το ρόλο του. Έχω λοιπόν ένα πρόβλημα. Ένα μέλος του ε, ελεγκτικού συνεδρίου της Ελλάδας προτείνεται εδώ ως υποψήφιος. Γι' αυτό λοιπόν πείτε μας, εσείς προσωπικά τι κάνατε για την κατάσταση με τα προβλήματα ε, που είχε η Ελλάδα και τα δημοσιονομικά. Είχαμε τόσες πολλές ε, προβλήματα σε ό,τι αφορά τα πραγματικά χρέη. Δεν θέλω να σας ε, δώσω την εντύπωση τη λανθασμένη, αλλά το θέμα της Ελλάδας είναι πολύ σημαντικό για μας, γιατί σε κάθε κρατος μέλος διδραματίζει μεγάλο ρόλο βλέποντας την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη και πόσο υποφέρει, πόσο επιβαρύνεται από το γεγονός ότι επιτρέψαμε πάρα πολλά πράγματα το 2010 στην δεύτερη επίσκεψη στην Ελλάδα μου δόθηκε καλή εντύπωση, πρέπει να ομολογήσω. Και όπου εκεί να πηγαίνουμε, βλέπουμε άτομα τα οποία έχουν αναλάβει τα καθήκοντα του τρει-τέσσερι εβδομάδε και μα λένε ότι α, δεν φταίμε εμεί, ήταν οι προκάτοχοι. Και μετά από πέντε χρόνια και πάλι ξαναεπισκεπτόμαστε τη χώρα και πάλι μα λένε ότι α, έφταιγαν οι προηγούμενοι, αλλά εμεί θα τα πάμε καλύτερα. Ξέρετε, συμμετέχω πάρα πολύ καιρό σε αυτό το παιχνίδι. Το ξέρω καλά. Θέλω πιο πολύ αξιοπιστία. Θέλω πιο πολύ εγκυρότητα. Σας παρακαλώ πείστε με, Κοίταξα και τους δείκτες για τη διαφάνεια και για την διαφθορά. Η Ελλάδα είναι στην θέση 94 με τον Τζιμπουτί, την Σουαζιλάνδη. Εσείς πώς έχετε ζήσει στο λειτουργήμά σας τη διαφθορά. Γιατί βλέπω ότι έχετε ασκήσει και άλλα, άλλα αξιώματα πέρα από το λεκτικό συνέδριο. Ερωτώ λοιπόν, γιατί δεν προσπαθήσατε να αποτρέψετε αυτήν την καταστροφή ή τι κάνατε, εν πάση περίπτωση για να αποτραπεί η καταστροφή. Σας ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Κύριε Μιλιώνη, θα θέλατε ίσως να απαντήσετε κατευθείαν. Ε, θα ήθελα να απαντήσω στις ε, ερωτήσεις σας Ω εξή Καταρχάς, δεν είμαι πρόεδρος, απλώς προείδευσα λόγω αρχαιότητος σε ένα τμήμα. Ε, πρόεδρος είναι άλλος. Εγώ είμαι σύμβουλος, ένας από τους πολλούς συμβούλους. Ε, πραγματικά, το τι κάναμε για την κρίση του ελεγκτικού συνεδρίου, για την κρίση της, ε, ε Ελλάδος σε αυτό το διάστημα μετά το 2010, είναι κάτι It was, Αναφέρθηκε, στα χαρτιά. Ε, το τι κάναμε ήταν ένα μεγάλο πρόβλημα. Ίσως να μην κάναμε τίποτα γιατί δεν μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα. Ο ελεγκτικό, θεσμός, γιατί εμείς είχαμε περιοριστεί, μας είχαν περιορίσει στον έλεγχο νομιμότητας και κανονικότητας των δαπανών, σε προληπτικό και κατασταλτικό. Δεν είχαμε τη δυνατότητα να κάνουμε ελέγχους επιδόσεων. Δεν είχαμε την, την δυνατότητα εκ του νόμου. Δεν φταίμε εμείς γι' αυτό. Κάποια στιγμή που επιχειρήσαμε να δώσουμε ένα άνοιγμα στην έννοια της, ε, του ελέγχου και να συμπεριλάβουμε και τον έλεγχο του performance audit, μας το, μας το απαγόρευσε. Δεν μας, ε, το Υπουργείο Οικονομικών ήρθαμε σε σύγκρουση. Λέει αυτό έχετε, με αυτό μπορείτε να κάνετε τη δουλειά σας. Πραγματικά στην Ελλάδα το μεγάλο ζήτημα είναι ο έλεγχος της αξιοπιστίας. Δεν, το, δεν αντιλέγει κανείς. Ο έλεγχος της, του, της εγκυρότητας των στοιχείων. Μας κατηγόρησαν πως, ακόμη πως μπήκαμε και στην, Ευρω... και στην με φαλκιδευμένα στοιχεία. Δεν ξέρω κατά πόσο αληθεύει αυτό. Είναι μια κατηγορία η οποία πλανάται. Σε εμά αυτή τη στιγμή μα κατηγορούν στην Ελλάδα πω ω ελεγκτικό θεσμό, ω ελεγκτικό συνέδριο δεν κάναμε τίποτα. Αλλά δεν μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα. Πιστέψτε με, ήμασταν πολύ περιορισμένοι. Πολύ περιορισμένοι. Στην Ελλάδα, ξέρετε, δεν υπήρχε η έννοια του εσωτερικού ελέγχου. Κάτι το οποίο εσεί θεωρείτε αυτονόητο, για μα εισήχθη το 2010 Συνεπώς, φανταστείτε πως εμείς στις εκλογές του 2009 πήγαμε στις εκλογές του 2009 με ένα, με ένα ε, χρέος λίγο παραπάνω από τα κριτήρια του Μάστριχ. Και μετά τις εκλογές εμφανίστηκε από την Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία εννέα μονάδες πιο πάνω. Πού είναι η εγκυρότητα την οποία, την οποία έχετε δίκιο και εξανίσταστε και αντιδράτε. Μετά από λίγο έρχεται η Κομισιόν και μας λέει «Πω, δεν είναι ξέρω εγώ, 10, 12, είναι 13 και 14». Καταλαβαίνετε πως εμείς χαθήκαμε, βρεθήκαμε σε μια κατάσταση. Από τη μία πλευρά εμείς ήμασταν ανίκανοι και κακώς μας τύπτει η κοινωνία και εσείς και η ελληνική κοινωνία και η ευρωπαϊκή, πως δεν κάναμε καλά τη δουλειά μας, αλλά απ' την άλλη είμαστε σε μια κατάσταση που δεν μπορούσαμε να αντιδράσουμε. Γιατί η διαφορά πραγματικά δεν είναι ε, επειδή τυχαίνει να, να είχα ασχοληθεί και με τη διαφθορά σε κάποια, ε, κάποια αρθρογραφία μου και παρατηρώ αυτού του δείκτε διαφθορά, δεν με κολακεύει καθόλου ω Έλληνα να είμαι μαζί με το τσιμπουτί. Δεν με κολακεύει καθόλου. Ξέρετε και εγώ, σα το ομολογώ, πω κάποια στιγμή, επειδή ήμουν πρόεδρο σε ένα ε, ε, κλιμάκιο, σε ένα, ένα σχηματισμό για τον, για τον έλεγχο, τον προσυμβατικό έλεγχο των σχεδίων συμβάσεων, και ήταν, ήρθε κάποιος ε, επιχειρηματίας και μου είπε σας παρακαλώ αν θέλετε προχωρήστε λίγο την υπόθεσή μου εντάξει του λέω πολλές, πολλές είναι εδώ αφού βιάζεστε θα το κάνω και μετά ήρθε να μου δώσει χρήματα τρόμαξα, με είδε ευγενικό και νόμισε πως αυτός είναι χειραγωγούμενος μετά μόλις κατάλαβα περί τίνος πρόκειται του λέω σας παρακαλώ μην ανοίξετε αυτό το πράγμα μην ανοίξετε την τσάντα σα γιατί θα καλέσω τον αστυνομικό από την, από την είσοδο. Καταλαβαίνετε πόσα αυτό που θεώρησε αυτονόητο για μένα, να το κάνει σε μένα που ήμουν δικαστή, πού το, που το είχε κάνει. Η διαφθορά είναι κάτι το οποίο δυστυχώ ανθεί στη χώρα μου, όπως και οι πορτοκαλιές. Δυστυχώ. Ελπίζω να σας έπεισα με την απάντησή μου. Ευχαριστώ πολύ. Στο σημείο αυτό θα ευχαριστήσω. Θα ζητήσω κάτι ακόμη από τον κύριο Μιλιώνη. Θα επιμείνω, διότι υπάρχει μια ερώτηση. Ακόμη. Κατά βάση. Τώρα, η Ελλάδα είναι 30 χρόνια μέλο Ευρωπαϊκή. 40 μέλο Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αν καταλαβαίνω αυτό που μα λέτε, γι' αυτό και επιμένω με την ερώτησή μου. Μα λέτε ότι το ελληνικό Ελεκτικό συνεδρίο για νομικούς, πραγματικούς όρους δεν ήταν η θέση να προβεί στον έλεγχο του, ελληνικού, του προπολογισμού του ελληνικού κράτους κατά τρόπον ώστε ε, ε, σφαλμένες χρήσεις ή εγγραφές και προβλήματα όπως αυτά που διαπιστώνονται τώρα με την Τρόικα να διαπιστωθούν από το ελεγκτικό συνέδριο της Ελλάδας. Δηλαδή το ελληνικό ελεγκτικό συνέδριο, αν καταλαβαίνω σωστά αυτό που μας λέτε, για, για λόγους πραγματικούς, πρακτικούς ή νομικούς, δεν μπορούσε να κάνει σωστό δημοσιονομικό έλεγχο του ελληνικού προπολογισμού. Εάν αυτό ισχύει, το ερώτημα για μένα είναι το εξή. Η Ελλάδα ως κράτος μέλος θα πρέπει να έχει στο μέλλον να λαμβάνει ευρωπαϊκά κονδύλια. Πώς βλέπετε εσείς αυτό με τον προβληματισμό. Ε, πράγματι κύριε Πρόεδρε, η Ελλάδα είναι πολλά χρόνια, είναι από το 81 μέλος της, ε, των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων τότε και της Ευρωπαϊκής Ένωσης βέβαια μεταγενεστέρως. Ε, το ελεγκτικό συνέδριο, ποια είναι η σχέση τώρα του ελεγκτικού συνεδρίου με όλο αυτό. Πραγματικά το ελεγκτικό συνέδριο για λόγους νομικούς, για λόγους πραγματικούς, είχε περιορισμένες αρμοδιότητες. Έμεινε σε, έναν νομικισμό, δηλαδή σε μια, έναν τρόπο περιορισμού με διατάξεις. Δεν μπορούσε να έχει έναν πραγματισμό και να ξεπεράσει αυτές τις, ε, αυτού, αυτά αυτούς τους περιορισμούς. Ε, όμως, την άλλη δεν πρέπει να το αδικούμε και πάρα πολύ διότι στην ετήσια έκθεση και στην έκθεση του απολογισμού του κράτους που ε, υποβάλλει στην Βουλή το ελεγκτικό συνέδριο έκανε παρατηρήσεις αλλά έκανε παρατηρήσεις οι οποίες ε, ήταν εις ότα μη ακουόντων διότι ε, και το όλο σύστημα ήταν χολό και τι εννοώ οι εκθέσεις οι οποίες υποβάλλονταν, υποβάλλονταν στον πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων χωρίς να συζητηθούν περαιτέρω. Ε, τώρα τελευταία εισάγονται στην Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου της Ελληνικής Βουλής. Σημαίνει πως δεν υπήρχε και η θεσμική συγκρότηση όχι μόνο του Ελληνικού Ελεγκτικού Συνεδρίου και από την άλλη της Βουλής για να δεχθεί, για να ακούσει σοβαρά τις παρατηρήσεις του ελεγκτικού συνεδρίου και να τις υιοθετήσει. Αυτά γράφονταν και ξαναγράφονταν στις αιτήσεις εκθέσεις και τη μία χρονιά και την άλλη χωρίς να βρούμε ανταπόκριση. Ε, πραγματικά τώρα με την Τρόικα σε αυτή την κατάσταση που βρισκόμαστε ε, έχετε δίκιο να λέτε για το ζήτημα το τόσα χρόνια τι κάνατε με τις κοινοτικές, με τις δαπάνες. Πραγματικά ε, η, η κατάχρηση αυτή των κοινοτικών δαπανών είχε φτάσει σε τέτοια σημεία μέχρι σαν εκδότου ε, το πώς γίνονταν η κατάχρηση αυτών των χρημάτων. Ε, ίσως φταίνε πολύ, ίσως να φταίει το όλο σύστημα όπως ήταν διαρθρωμένο από την αρχή που δίνονταν οι ε, κοινοτικές ε, ενισχύσεις χωρίς να έχει ελεγχθεί προηγουμένως αν υπάρχει σύστημα εσωτερικού ελέγχου σε κάποια χώρα και ε, προκειμένου στη χώρα μου. Και αυτά τα χρήματα έφευγαν ως, ως ο πίθος των Δαναίδων. Έριχνε το νερό και έφευγε από κάτω. Ήταν δηλαδή μια κατάσταση πολύ δυσάρεστη και έχετε δίκιο να εξανίσταστε και να ε, αμφισβητείται ακόμη και την δυνατότητα της χώρας μου να ε, παίρνει τέτοιες ε, κοινωτικά χρήματα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Οντή, μετά η κυρία Γκρέστσλε. Αυτές οι ακροάσεις γίνονται όλο και πιο συναρπαστικές τελικά. Δεν σκόπευα να διατυπώσω το ίδιο ερώτημα για τα κατά ταμεία, αλλά προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στρεφόμενος, δεδομένου ότι δεν γνωρίζω καλά τα κεφάλαια των διαπραγματεύσεων για την ένταξη των κρατών μελών, αλλά πιστεύω ότι για την ένταξη ενός κρατου μέλους στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχει κάποιο κεφάλαιο προς τις διοικητικές δομές για το δημοσιονομικό έλεγχο και άρα η προσχώρηση ενός κράτους μέλους έγινε την εποχή εκείνη χωρίς επαλήθευση ότι το εθνικό θεσμικό όργανο ελέγχου δεν είχε τον έλεγχο στον προπολογισμό. Άρα ε, θα πρέπει να δούμε πώς υλοποιείται. ε, να γνωρίζουμε ότι έχει γίνει ο σωστός δημοσιονομικός έλεγχος. Πώς λοιπόν μπορεί να συνέβη κάτι τέτοιο και πώς μπορεί να μην έχουν ξεκινήσει ανάλογες διαδικασίες αν δεν υπήρχε ανεξαρτησία. Ευχαριστώ πολύ κυρία Γκρέσλε. Θα ήθελα να μας πείτε δύο λόγια. Καταρχάς σας ευχαριστώ για τις απαντήσεις σας, σας ευχαριστώ για τη δέσμευση που κρύβεται πίσω από αυτές. Ξέρω ότι για εσάς είναι δύσκολη η κατάσταση και πιστέψτε μας και για μας είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση. Εγώ ήμουν στις δύο επισκέψεις στην Ελλάδα. Στην πρώτη επίσκεψη ο λόγος ήταν ότι η Ελλάδα δεν είχε εφαρμόσει το Άγιαξ το 2007 παρά το γεγονός ότι υπήρχε αυτή η προϋπόθεση από το 97 για να, πάρει, ε, να παίρνει πόρους. Δηλαδή, επί 10 χρόνια και πλέον έπαιρνε χρήματα η, η Ελλάδα χωρίς να έχει χωρίς να πληρούνται οι, οι, οι κατάλληλοι όροι. Και η κυρία Φίσερ Μπέλ νομίζω το έχει επισημάνει αυτό. Ε, βοήθησε η επίσκεψή μας. Και είπαμε ότι κοιτάξτε, εάν σε δύο έτη δεν πληρούνται οι παρετόροι, τελείωσε. Το 2010 το ποσοστό σφάλματος είχαμε διαπιστώσει ήταν στο 3,5%, 4%, περίπου 3,5%. Το 2010 στην όλη αυτή η κατάσταση διαπιστώσαμε κάτι ενδιαφέρον. Μιλήσαμε και με τα άτομα τα υπεύθυνα για τα διευθυντικά ταμεία. Μας είπαν ότι όλα πήγαιναν καλά και τότε Φύγαμε από τις συνομιλίες και στο δείπνο διάβασα την εφημερίδα Le Monde. Μία συνέντευξη συμπεριλαμβανόταν με τον Υπουργό Οικονομίας και ανέφερε ότι, κοιτάξτε, τα χρήματα για τα ελευθερωτικά ταμεία τα σπαταλήσαμε, τα κατασπαταλήσαμε για πισίνες και αυτοκίνητα. Υπό ποια μορφή λοιπόν το ελεκτικό συνέδριο φρόντισε για τα μέσα αυτά, για τα ελευθερωτικά ταμεία, για τα αγροτικά τους αγροτικούς πόρους και έχω μία ανησυχία, μην την πάρετε προσωπικά γιατί δεν σας γνωρίζω προσωπικά, δεν σας έχω ξαναγνωρίσει. Νομίζω σε μία επίσκεψη ήταν και εσείς μαζί, αλλά εν πάση περιπτώσει. Η Ελλάδα παίρνει πλέον ένα 95% συγχρηματοδότηση. Δηλαδή ουσιαστικά υπάρχει και επιβράβευση. Εσείς πώς θεωρείτε αυτή την συγχρηματοδότηση. Γιατί για πολλά έργα δεν έχουμε εκθέσεις ε, και οι εκθέσεις της Τρόικας και οι εκθέσεις της Task Force είναι πολύ ενδιαφέρουσες γιατί ακριβώς μιλούν για τα έργα αυτά. Εγώ ανησυχώ ότι η ευθύνη της Ελλάδας θα είναι ακόμα πιο μικρή λόγω της συγχρηματοδότησης. Μήπως επιδεινώνεται η κατάσταση. Και γι' αυτό η δική σας θέση είναι πάρα πολύ σημαντική, γιατί σε καμία περίπτωση δεν θα μπορέσουμε να ανοιχτούμε ο Έλληνας υποψήφιος, το, ελληνικό, το μέλος από πλευράς της Ελλάδας, να προσπαθήσει να συγκαλύψει τέτοιες καταστάσεις. Ευχαριστώ. Uh, Ευχαριστώ. Ένα τελευταίο μέλος θέλει να κάνει μια ερώτηση και νομίζω θα πρέπει να ολοκληρώσουμε τότε την ε, ακροασία. Ο κύριος Επίνγκ. Ε, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εγώ έχω μία ερώτηση να κάνω, επειδή βλέπω στο βιογραφικό ότι ο υποψήφιος το 95-96 ε, εργαζόταν ε, ως επιτετραμένος για το ελληνικό ελεκτικό συνέδριο και τότε ήταν ο κύριος Νικολάου Κολόπου ήταν το άτομο αυτό το υπεύθυνο από πλευράς του ελληνικού συνεδρίου. Yes. Okay. Go ahead, please. Δεν παρακαλώ, λέει ο Ε, δεν ξέρω αν θυμάμαι λάθος. Ε, δούλευα για τον Επιτροπό Κάλλας στην υπηρεσία του το 2003 μέχρι το 2007. Ακούστηκε ένας whistleblower που μας ε, είπε ότι κάποια μέλη του ελληνικού ελεκτικού συνεδρίου και μας μίλησε για ένα μέλος το οποίο συνήθιζε τα μέλη της υπηρεσίας τους να τις δίνουν ένα τμήμα του μισθού τους. Το γνωρίζετε αυτό, γνωρίζετε να υπήρξε κάτι τέτοιο. One question, uh, θέλεις να κάνεις ε, την ερώτησή σου πριν την απάντηση ή μετά την απάντηση του κυρίου Μιλιώνη. Μετά, μετά την απάντηση. Κύριε Μιλιονί. Ε, πράγματι ε, κύριε Οντή, ε, το ζήτημα των ε, διοικητικών δομών στην Ελλάδα είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Το είπαμε και το ξαναλέμε, δεν υπάρχουν εσωτερικοί έλεγχοι. Αυτό είναι το μεγάλο ζήτημα. Το μεγάλο ζήτημα και μπορεί να έρχονται χρήματα ή μπορεί να έρχονταν χρήματα μέχρι πρώτη. Τώρα αναγκαζόμαστε να κάνουμε εμβαλωματικές λύσεις, αλλά προσπαθούμε να κάνουμε λύσεις έρχονταν και έφευγαν όπως από το πιθάρι, από τον πίθο των Δαναίδων όπως σας είπα. Αυτό είναι ένα μεγάλο, μια μεγάλη αλήθεια, δεν θέλει κανείς να την κρύψει, την ξέρουμε. Την ξέρουμε, ξέρουμε τα προβλήματά μας. Ε, σε ό,τι αφορά βέβαια για τα διαρθρωτικά ταμεία και με τις πισίνες και τα αυτοκίνητα, ε, εμείς, ε, κυρία Γκρέσλε, έχουμε, σαν ελεγκτικό συνέδριο, έχουμε μια αρμοδιότητα να κάνουμε έλεγχο, όχι πρωτογενή, δευτερογενή, στα συγχρηματοδοτούμενα, ε, τον πρωτογενή έλεγχο τον κάνει το Υπουργείο Οικονομικών. Υπάρχει μια ε, Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου, η οποία ε, ελέγχει τα συγχρηματοδοτούμενα και κατόπιν έρχονται σε εμά ακολουθώντας την, δικαστική οδό. Εκεί πραγματικά συμμετείχα, συμμετείχα και καταλόγησα, δηλαδή ζήτησα χρήματα πίσω πάρα πολλά. Ίσως να ήμουν και αυστηρός, περισσότερο από το κανονικό. Ε, το ξέρω πως ε, τα ζητήματα αυτά τα, ε, με, τα, μεγάλα ε, δομικά συστημικά προβλήματα της Ελλάδος ενδεχομένως να οδηγήσουν να, μειωθεί η, ελληνική συνεισφορά και να αυξηθεί. Αλλά αυτό είναι ζήτημα το οποίο είναι πολιτικό υποθέτω. Αλλά εμείς τη δουλειά μας προσπαθούμε να την κάνουμε. για το Άλλο ζήτημα για τον κύριο Αντρουτσόπουλο ή, τον, ή την κυρία Νικολάου. Δεν έχω ακούσει κάτι τέτοιο. Εγώ ήμουνα μέλος, ε, βοηθός, ατασέ του αείμνηστου του Αντρουτσόπουλου έχει πεθάνει ο άνθρωπος αυτός τώρα, ε, με την κυρία Νικολάου πραγματικά έχει ακουστεί, δεν ξέρω αυτό τώρα αν είναι αληθινό ή δεν το ξέρω αυτό για τον μισθό. Ξέρω όμως πως είχε άλλα προβλήματα και είχε φτάσει σε σημείο μέχρι και το δικαστήριο για να, της στερηθεί, να, να αποστερηθεί την σύνταξή της. Ε, αυτά ξέρω για την κυρία Νικολάου, δεν την ξέρω την κυρία, εγώ είχα φύγει, αλλά μιλάμε για την... Ο, άλλος, ο, ανθρωπόπουλος ήταν ένα τίμιο άνθρωπος, σοβαρό, δεν ανήκε βέβαια, ήταν από άλλο, ήταν νομικό, απολύτω νομικό, το νομικό συμβούλιο του κράτου. Ευχαριστώ πολύ. Σα ευχαριστώ πολύ. Και τώρα η συγκέντρια κυρία Γιάννα Σάντερ, παρακαλώ. Κύριε Μιλιώνη δεν είστε εσείς υπεύθυνο για όλα τα οικονομικά και κοινωνικά θέματα και τις σχετικές δομές, αλλά σας θέτουμε ερωτήσεις ε, και καλείστε να δώσετε απαντήσεις να είστε ε, υπεύθυνο όλων των ε, δράσεων των κυβερνήσεων από την ένταξη της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι αλήθεια πάντως ότι η κατάσταση του ελεκτικού συνεδρίου στην Ελλάδα είναι ε, θεμελιώδης σημασίας και για το μέλλον ε, της συνεργασίας των διαφόρων εθνικών ελεκτικών συνεδρίων. Γιατί θα πρέπει να ισχύουν κάποιες ε, διατάξεις και κάποια εναρμόνιση όπως αναφέρεται πολύ σωστά στη σελίδα 15 της εκθεσής σας. Οπότε το 2010, τη στιγμή που μπορούμε να πούμε ότι θεσπίζεται ο νόμος ώστε το ελεκτικό συνέδριο να μπορεί να στέλνει τις εκθέσεις του στο, στην Βουλή των Ελλήνων γιατί λέτε κι εσείς ότι η συνεργασία αυτή είναι σημαντική για την σωστή διαχείριση και τον έλεγχο των λογαριασμών. Θα ήθελα να υπενθυμίσω στους συναδέλφους ότι δεν θα πρέπει μαζί με τα ξερά να κλαίμε, να κλαίμε και τα χλωρά. Ο κύριος ε, Μιλιώνης έδωσε πραγματικά μάχη και έκανε ό,τι μπορούσε σε ένα λεκτικό συνέδριο που ήταν ήδη προβληματικό. Αλλά όπως είπε ο κύριος Σοντή, Πολύ συχνά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν ξεκίνησε η διαδικασία επιβολή κυρώσεων ούτε κατά τη Ελλάδα, ούτε κατά τη δική μου πατρίδα Ισπανία, αλλά ούτε κατά τη Γαλλία, ούτε και κατά τη Γερμανία. Όταν αθετήθηκαν οι υποχρεώσεις τους, αυτές που είχαν αναλάβει δηλαδή στο Συμβούλιο του Άμστερνταμ. Θα πρέπει λοιπόν να είμαστε συνεπείς και να εφαρμόζουμε τον ίδιο κανόνα σε όλους, όχι μερικές φορές να εφαρμόζουμε καλύτερα τον ένα κανόνα σε ορισμένους και χειρότερα σε άλλους. Και εμεί παρακολουθήσαμε εκ του σύνεγγυ στην κατάσταση στην Ελλάδα, αλλά σίγουρα ο κύριο Μιλιώνη δεν είναι ο υπεύθυνο, ο υπέτειο για την κατάσταση στην Ελλάδα, Απλώ είναι υπεύθυνο γιατί επισήμανε, ανέδειξε ουσιαστικά ε, τις ανεπάρκειες του ελεκτικού συνεδρίου της Ελλάδας, στο οποίο συμμετείχε. Και από την στιγμή που ανέλαβε τα καθήκοντά του, συνέβαλε στη βελτίωση του συστήματος. Δεν θα ήθελα λοιπόν να, μετατρέψουμε σε αποδιοπομπαίο τράγο έναν υποψήφιο που συνέβαλε στη βελτίωση της κατάστασης θα πρέπει να υιοθετήσουμε και μια διαλεκτική μέθοδο και θα πρέπει να έχουμε άμεσο και ειλικρινή διάλογο μεταξύ μας. Εγώ πιστεύω ότι συγκεντρώνεται και βαθύτατες και έγκυρες γνώσεις ε, για την κατάσταση και μάλιστα εσείς στυλιτεύσατε, αναδείξατε και στυλιτεύσατε τις ανεπάρκειες αυτές που εντοπίσατε στη χώρα σας. Και πιστεύω ότι θα μπορέσετε και εσείς να συμβάλλετε και να μας βοηθήσετε ώστε να αποφύγουμε και το ελεγκτικό συνέδριο της Ελλάδας που στο μέλλον θα συνεργαστεί με το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο αλλά και όλα τα συστήματα ελέγχου των ε, Ευρωπαϊκών Ταμείων και της χρήσης των Ευρωπαϊκών Κονδυλίων τα οποία αξιοποιεί, λαμβάνει και αξιοποιεί η Ελλάδα θα εξασφαλίζεται σημαντικός έλεγχος ε, για την διαχείρισή τους και στη περίπτωση που εγκρίνουμε την υποψηφιότητά σας για να είστε ο επόμενος Έλληνας μέλος του Ελεκτικού Συνεδρίου, με τι συγκεκριμένες δράσεις πιστεύετε ότι θα μπορούσαμε να βελτιώσουμε ε, την κατάσταση και να διορθώσουμε αυτές τις ε, κρεμότητες που υπάρχουν και τα μεγάλα ερωτηματικά σε ό,τι αφορά τη χρηστή, ε, το χρηστό έλεγχο τον, ε, ευρωπαϊκό λογαριασμό, τον ελληνικό λογαριασμό σε ό,τι αφορά τη χρήση και την αξιοποίηση των ευρωπαϊκών κονδύλιων. Σε περίπτωση λοιπόν που διοριστείτε πώς θα συμβάλλετε ώστε να εξασφαλίσουμε όλη αυτή τη διαφάνεια που χρειαζόμαστε για την κατάσταση των λογαριασμών της Ελλάδας, τι μηχανισμούς έχετε για να μας βοηθήσετε για κάτι που είναι θεμελιώδες και για τη χώρα σας αλλά και για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα παρακαλώ το λόγο να λάβει ο κύριος Μιλιώνης. Σας και παρήγορο ε, λόγο, ε, όμως πραγματικά αισθάνομαι υπεύθυνο για αυτά που συμβαίνουν στη χώρα μου, γιατί όπως έλεγε και ο Νίκος Καζαντζάκης, κάτι να μην πάει καλά στην κοινωνία, υπεύθυνο είμαι εγώ. Ε, αν ε, λάβω την ε, ε, ευνοϊκή σας γνώμη, τη συγκατάθεσή σας για, την, για το διορισμό μου, Καταρχάς, σε ό,τι αφορά την, τη σχέση μου με το ελληνικό ελεγκτικό συνέδριο, θα είναι ο ρόλος μου περιορισμένος. Θα είναι ένας ρόλος ο οποίος θα στηρίζεται κυρίως σε προσωπικούς και, σε, και λιγότερο σε, θεσμικούς, σε θεσμικές δυνατότητες. αν από τη θέση την οποία ενδεχομένως να έχω μέλος του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου έχω την δυνατότητα να επηρεάσω το, το, Προεδρείο του Ελληνικού, Ελεκτικού, του, του Ελληνικού Ελεγκτικού Συνεδρίου να μεταβάλει όπως και πράγματι θέλει και στην πραγματικότητα άρχισε να μεταβάλει τους, τις δομές του Ελληνικού Ελεγκτικού Συνεδρίου θα το κάνω με μεγάλη μου χαρά. Κυρίως εκείνο που έχει σημασία στην Ελλάδα είναι να φύγουμε από τον νομικισμό, δηλαδή από τον εγκλισμό μας στις νομικές ε, διατάξεις και να περάσουμε σε έναν πραγματισμό. Ε, να γίνουμε πιο εμπειριστές αντί να είμαστε να κολλάμε στο πνεύμα του νόμου. Αυτό θα γίνει μέσω του ελέγχου επιδόσεων. Και πραγματικά στην Ελλάδα το νομικό, το πλαίσιο υπάρχει και υπάρχει και η επιθυμία να αρχίσουμε ελέγχους επιδόσεων, performance audit. Σε ό,τι αφορά βέβαια τις ε, δικές μας ε, την επαφή μου με, το, με την Επιτροπή σας θα είναι ζήτημα, είναι ζήτημα ε, πλέον είναι θεσμικό. Ε, ε, το, το, ελεγκτικό συνέδριο της, το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο είναι κομμάτι από εσά. Έγινε με δικιά σας πρωτοβουλία και συνεπώς οι σχέσεις μας πρέπει να είναι εξαιρετικές και τακτικές και ειλικρινείς. Αυτά έχω να πω. Ευχαριστώ πολύ. Ja, vielen Dank. Wir danken Ευχαριστούμε κύριε Μιλιώνη για, την, ε, για τις απαντήσεις που δώσατε στις ερωτήσεις μας. Έτσι μπορούμε να ολοκληρώσουμε την ακρόαση του κύριου Μιλιώνη. Σας ευχαριστούμε πολύ και στο επανειδέν. Ευχαριστώ και εγώ. Καλή σας μέρα.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 Κυρίε äh, Κυρίες και κύριοι, σε αυτή τη φάση θα ήθελα να καλωσορίσω την υποψήφιο της ε, Γαλλίας, την κυρία Ντανιέλ Λαμάρκ. Καλώς ορίσατε. Θα θέλαμε να ακούσουμε την παρέμβασή σας. Καλώς ορίσατε κυρία Λαμάρκ. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι Ευρωβουλευτέ, σας ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνετε ε, να έρθω εδώ και χαίρομαι και αισθάνομαι ιδιαίτερη τιμή για την ακρόαση αυτή στην Επιτροπή σας. Όπως διαβάσατε και από το βιογραφικό μου, ε, η σταδιοδρομία μου αφιερώθηκε κυρίως στον έλεγχο των ε, δημοσίων οικονομικών στα πλαίσια του Γαλλικού Ελεκτικού Συνεδρίου και μάλιστα είχα την τύχη να ασχοληθώ με όλες τις πτυχές ε, του ελέγχου και στις αστικές και ποινικέ διαδικασίες και την αξιολόγηση των δημοσίων οικονομικών που μετά με τη συστηματική αναθεώρηση του 2008 έχει ε, ενταχθεί στις ε, αρμοδιότητες του Ελεκτικού Συνεδρίου και στην υπηρεσία του Κοινοβουλίου. 15 χρόνια είχα τέτοια εμπειρία στο Ελεκτικό Συνέδριο και ήμουνα και ε, πρόεδρο σε δύο περιφερειακά ελεκτικά συνέδρια, στη Μαρσαλία και στην Άλπα Κονταζούρ στην Εκτή και ε, στην διάρκεια της αντιδρομίας μου είχα διάφορες δραστηριότητες ε, σε κρατικές υπηρεσίες και μάλιστα τα μέλη του Ελεκτικού Συνεδρίου της Γαλλίας ε, συμμετέχουν σε διάφορες επιτροπές ή προεδρεύουν σε συμβούλια γιατί γνωρίζουν τα γρανάζια του κράτους και έχουν φυσικά και την φήμη της αμεροληψίας. Οπότε στις διάφορες δραστηριότητες που συμμετείχα. Συμμετείχα και στο Διοικητικό Συμβούλιο μιας μεγάλης σχολής για κατάρτιση στο τομέα της υγείας. Συμμετείχα στο Επιστημονικό Συμβούλιο Αξιολόγησης της ε, Κρατικής Πολιτικής και σε, διάφορες, ε, σε διάφορα συνέδρια, κριτικές επιτροπές, σεμινάρια και το καθεξής. Σε όλες τις ευθύνες που άσκησα στα, παράλληλα με, με την ιδιότητά μου ως μέλος του Γαλλικού Ελεκτικού Συνεδρίου, έλαβα, έμαθα και διδάχθηκα πολλά. Επίσης, ε, ως μέλος του Περιφερειακού Ελεκτικού Συνεδρίου, ε, είδα όλες τις φάσεις του ελέγχου, από τον προγραμματισμό έως τις ε, σχέσεις με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Προγραμματισμό σημαίνει επιλογή των οργανισμών και των θεμάτων, για τα οποία είναι πιο χρήσιμο και σημαντικό να εργαστεί κανείς, ανέβρεση του καλύτερου συνδυασμού μεταξύ της στρατηγικής ελέγχου και των περιορισμένων μέσων που διαθέτουμε και επίσης ε, παρακολούθηση όλων των βασικών σημείων του ελέγχου, καθορισμός του σχεδίου ελέγχου, επιλογή των καλύτερων μεθόδων για τα πιο ε, καλά αποτελέσματα, επιθεώρηση του ελέγχου, διαχείριση και σχηματισμό σύνθεση των ε, μονάδων και τηρήση των χρονοδιαγραμμάτων και υποβολή ποιοτικών εκθέσεων, προκειμένου να εξασφαλιστεί η αυστηρότητα ε, και η αποτελεσματικότητα του έργου και η βελτίωση η αναβάθμιση της ποιότητάς του. Και πιστεύω ότι με αυτή την εμπειρία θα μπορέσω να ασκήσω και τα καθήκοντά μου ως μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινικού Συνεδρίου, αν με ε, εγκρίνεται. Καθ' όλη τη διάρκεια της σταδιοδρομίας μου ε, ήμουν υπέρ των διεθνών επαφών γιατί πιστεύω ότι μαθαίνουμε πολλά από τους άλλους και όσο ήμουν επικεφαλής ε, της Διεθνούς Υπηρεσίας, ε, του Συμβουλίου, Σχέσεων του Συμβουλίου, είχα επαφές με συναδέλφους ε, από ελεκτικά όργανα της Ένωσης, προκειμένου να βελτιωθεί η συνεργασία μεταξύ των Εθνικών Φορέων Ελέγχου και του Ευρωπαϊκού Ελεκτικού Συνεδρίου. Επίσης, είχα αναλάβει τις σχέσεις του Ελεκτικού Συνεδρίου με διάφορες φορείς, εντός και και με τις 45 φορείς ε, του γαλόφωνο, των γαλόφωνων χωρών. Και θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό να συσφίξουμε τι σχέση μεταξύ των θεσμικών οργάνων, ώστε να βοηθήσουμε τους πιο ευάλωτους ε, να εμπεδώσουν την ανεξαρτησία τους και να μπορέσουν να διαδραματίσουν πιο αποτελεσματικά το ρόλο στη χώρα τους. Είναι σημαντικό ο ρόλο τη Ευρωπαϊκή Ένωση μέσα αυτών των αντιπροσωπιών. Καθ' όλη τη διάρκεια τη διαδρομία μου είχα στενέ σχέσει και με τον πανεπιστημιακό κόσμο, με δημοσιεύσει, ε, με σεμινάρια και διαλέξεις και πιστεύω ότι μπορούμε να ασχοληθούμε με το δίκαιο, με, τις, με την οικονομία, τις κοινωνικές επιστήμες. Όλα αυτά είναι χρήσιμες πτυχές για την καλύτερη αντίληψη ε, και κατανόηση της κατάστασης. Θα ήθελα τώρα να, επιμείνω σε, να, επιμείνω σε ένα σημαντικό θέμα ε, το οποίο σας είναι ιδιαίτερα προσφυλές, ε, το θέμα της ανεξαρτησίας. Ήμουν ανεξάρτητο μέλος ανέκαθεν και θεωρώ ότι η ανεξαρτησία βρίσκεται στο επίκεντρο της ε, δεοντολογίας ε, του επαγγέλματός μου. Και μάλιστα με το, τη μονιμότητα που έχουμε, έχουμε ένα είδος προστασίας, οπότε ε, εξασφαλίζεται η αμεροληψία και η ιδιαιτερότητα μας. Όλες οι παρατηρήσεις μας είναι ε, δημόσιες και απευθύνονται στον Ευρωπαίο πολίτη. Πιστεύω ακράδαντα στην ανεξαρτησία και όχι μόνο για κανονιστικούς και θεσμικούς λόγους. Είναι μια πρακτική, μια ανατροπή και μια κουλτούρα που θα πρέπει συνεχώς να ενισχύουμε. Για να είναι κανείς ε, όντως ανεξάρτητος θα πρέπει να μην υπόκειται ούτε σε προκαταλήψεις, ούτε σε ιδέες προκαθορισμένες, ούτε να άγεται και να θέλετε από την κρατούσα γνώμη της, ε, διάφορης ε, στιγμής. Γι' αυτό είναι σημαντική και η κατάρτιση, η εκπαίδευση και οτιδήποτε μας βοηθά να προοδεύσουμε στην πρακτική μας, στην ενίσχυση των μεθόδων μας και στην καλύτερη επαφή με τον εταίρο μας και των ε, Φυσικά ανεξαρτησία χτίζεται με τις ανταλλαγές και όχι με μια ισοστρέφεια. Φυσικά και το Ευρωπαϊκό Ελεκτικό Συνέδριο θα πρέπει να, εργάζεται, να συνεργάζεται στενά με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το να λαμβάνει υπόψη τον προγραμματισμό του, ώστε ο έλεγχος αυτός να ανταποκρίνεται στις προσδοκίες των Ευρωπαίων πολιτών. Αν με τιμήσετε με την εμπιστοσύνη σας. Θα αναλαμβάνω τη δέσμευση να έχω στενές επαφές με την Επιτροπή σας ως μέλος του Ευρωπαϊκού Ελεκτικού Συνεδρίου και θα είμαι στη διάθεσή σας και θα σας ακούω με ιδιαίτερη προσοχή. Ευχαριστώ. Ε, Ευχαριστώ πολύ, κύριε Λαμάρκ. Και τώρα μπορεί να γίνει συζήτηση. Καλύτερα η ερωτήτα από ακρίσεις και ρωτώ ποιος θέλει να ξεκινήσει. Η συγγήτρια πρώτα. Κυρία Γιάννα Σάντερ. Ευχαριστώ. Καλώς ήρθατε στην Επιτροπή μας, κυρία Λαμάρκ. Είστε υποψήφια των Γαλλικών Αρχών για το Ευρωπαϊκό Ελεκτικό Συνέδριο. Χαίρομαι ιδιαίτερω γιατί η κυβέρνησή σα έλαβε υπόψη τι συστάσει τη επιτροπή Ελέγχου προπολογισμού, προσπαθώντα να επανισορροπήσει την εκπροσώπηση των δύο φύλων στο Γαλλικό Ελεκτικό Συνέδριο. Και από τι πέντε υποψηφίου που έχουμε σήμερα ε, είστε εσεί η μόνη γυναίκα υποψήφια και χαίρομαι για το γεγονό. ότι υπάρχει έστω και μία γυναίκα υποψήφια για τη θέση του μέλους του Ευρωπαϊκού Ελεκτικού Συνεδρίου και αν ευοδοθεί η υποψηφιότητά σας θα εξασφαλιστεί κάπως μεγαλύτερη ισορροπία σε ένα θεσμικό όργανο ώστε να ανταποκρίνεται περισσότερο στην εικόνα και της κοινωνίας. Το βιογραφικό σας ε, είναι πολύ εντυπωσιακό. Αυτό με ενδιαφέρει, που με ενδιαφέρει περισσότερο είναι η εμπειρία σας στο Γαλλικό Ελεκτικό Συνέδριο. Είστε μάλιστα και πρόεδρος ε, ενός τμήματος που για μας είναι πολύ ενδιαφέρον και στο μέλλον αυτό μας ενδιαφέρει, να δούμε πώς ε, οι υποψήφοι των εθνικών αρχών μπορούν να βοηθήσουν καλύτερα την ε, λειτουργία του ελεγκτικού συνεδρίου. Η... Ήταν... Είναι πολύ εντυπωσιακή βέβαια η δραστηριότητά σας ό,τι αφορά την καταπολέμηση της ε, διαφθοράς και της δωροδοκίας. Η... Και σίγουρα ε, ήταν τόσο εντυπωσιακή δραστηριότητα που θα λείψετε πολύ από, τις, από τα περιφερειακά ελεκτικά συνέδρια της Μασαλίας και της περιοχής Ροδανούα, ε, ε, Ροδανόα, Άλπαιων και Κιανισακτής γιατί ήταν πραγματικά πολύ σημαντικό το έργο σας. Εσείς με την πλούσια πείρα που έχετε από την εμπειρία σας και την δραστηριότητά σας πώς μπορείτε να μας βοηθήσετε για να καταπολεμήσουμε και εμείς ε, την ε, διαφθορά, την πραγματική διαφθορά. Γιατί μερικές φορές ε, σε αυτή τη σύγχυση που υπάρχει μεταξύ των μηνυμάτων που λαμβάνουμε και των καταγγελιών δημιουργείται μια θολή εικόνα. Καλό θα λοιπόν κάποιος να μας δώσει ένα μήνυμα σαφήνειας και διαφάνειας προκειμένου να διορθωθεί αυτό το πρόβλημα. Τώρα, ε, μιλήσατε για χαρτογράφηση των ε, κινδύνων στις ε, δημόσιες πολιτικές. Αυτό είναι ένα στοιχείο που θα μπορούσε να μας βοηθήσει πολύ. Γιατί το έχουμε συζητήσει και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και με το Ευρωπαϊκό Ελεκτικό Συνέδριο. Το θέμα του σφάλματος, ε, του, του κινδύνου του σφάλματος και πώς θα μπορέσουμε να θεσπίσουμε ένα σύστημα προληπτικό ώστε να θεραπεύουμε, ώστε να προλαμβάνουμε το πρόβλημα και να μην χρειάζεται μετά να επέμβουμε για να το θεραπεύσουμε. Μπορείτε λοιπόν να μας διαφωτίσετε κάπως με βάση και τη δική σας ε, πείρα, γι' αυτό και που πολύ εύστοχα αποκαλέσετε χαρτογράφηση του κινδύνου. Επίσης, εργαστήκατε ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την κατάρτιση των διαφόρων οργανισμών για τους οποίους ασκήσατε έλεγχο. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το θέμα και στο, στη συζήτηση που έχουμε για το μέλλον του Ευρωπαϊκού Ελεκτικού Συνεδρίου, ένα τμήμα της συζήτησης αφορά ακριβώς ε, τα χαρακτηριστικά των υποψηφίων. Είπαμε ότι θα πρέπει να υπάρχει ένα καλό μείγμα μεταξύ των επαγγελματιών, ελεγκτών, ε, και των ε, εμπειρογνωμόνων του ελέγχου που θα προέρχονται από τους πανεπιστημιακούς κύκλους αλλά και ε, θα θέλαμε και εμπειρογνώμονες που θα προέρχονται ίσως και από, το πολιτικό, τον πολιτικό κόσμο γιατί το ελεκτικό συνέδριο ασχολείται και με προγραμματισμό και με αποφάσεις που έχουν ε, μείζωνα πολιτικό αντίκτυπο. Από τη δική σας πείρα και από το έργο που είχατε ώστε να καταστήσετε πιο επαγγελματικό το έργο των ελεκτικών συνεδρίων των διαφόρων φορέων. Πώς πιστεύετε ότι θα συμβάλλετε στη βελτίωση της κατάστασης και στο Ευρωπαϊκό Ελεκτικό Συνέδριο εφόσον εκλεγείτε. Ένα άλλο θέμα που μου προκάλεσε ιδιαίτερα το ενδιαφέρον είναι η ικανότητά σας να εργαστείτε για τη βελτίωση των ελεκτικών συνεδριών σε θέματα όπως είναι ε, θέματα ε, της Βόρειας Αφρικής, του Αραβικού κόσμου, το περιοχές που ενδιαφέρουν ιδιαίτερα και την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί έχετε συνεργασία και με το Ελεκτικό Συνέδριο της Τινησίας. Οπότε με την εμπειρία σας θα μας ανοίξετε και ένα παράθυρο συνεργασίας ε, με τις χώρες αυτές, γιατί υπάρχει και εκεί πραγματικά ανάγκη ελέγχου για χώρες που είναι γειτονικέ. Επίσης, σας ευχαριστώ και για τη θέση σας υπέρ της ανεξαρτησίας, αλλά ταυτόχρονα και υπέρ της επαφής και του μεγαλύτερου ανοίγματο και της συζήτησης με οργανισμούς και θεσμικά όργανα. Γιατί έχουμε ένα Ευρωπαϊκό Ελεκτικό Συνέδριο που βρίσκεται κάπως ε, στην άμυνα θεμητή και φυσιολογική, αλλά όταν λέμε ότι θέλουμε να βελτιώσουμε τη συνεργασία μας ε, και τον κοινό προγραμματισμό μεταξύ του Ευρωπαϊκού ε, Κοινοβουλίου και του Ελεκτικού Συνεδρίου, φυσικά ανακύπτει το ζήτημα της ανεξαρτησίας στο λίγο χρόνο που είχατε στη διάθεσή σας ε, μας είπατε ότι έχετε κάποιες ιδέες για το πώς μπορεί κανείς να διασφαλίσει και να ενισχύσει την ανεξαρτησία του δείχνοντας ένα μεγαλύτερο άνοιγμα και μένοντας ε, ευαίσθητος και ανοιχτός ε, στα αιτήματα των Ευρωπαίων πολιτών. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κυρία Ραμάρκη, έχετε το λόγο. Euh, ευχαριστώ πολύ. Θα απαντήσω ταυτόχρονα στα δύο προβλήματα, εντοπισμό κινδύνων και κίνδυνο, κινδύνων σχετικών με την διαφθορά. Στην αποστολή μας ως ελεγκτών, το πρόκειται στην Εθνική, για την Εθνική Αρχή και για το Ευρωπαϊκό Ελεκτικό Συνέδριο, ε, ε, χειριζόμαστε θέματα που έχουν, ενέχουν κίνδυνο οικονομικό και νομικό πλαίσιο που προκύπτει από αυτά, όπως παράδειγμα οι δημόσιες συμβάσεις ή συμβάσεις εταιρική σχέσεως κτλ. Πρόκειται για υψηλό, αυξημένο δηλαδή κίνδυνο. Οι τοπικές αρχές στη Γαλλία έχουν ε, ποσοστό τριών τετάρτων στις συνολικές επενδύσεις και οι συμβάσει εκχώρησης ε, σε πολλά σε πολλές πτυχές της καθημερινής ζωής. Είδα τα καθαρισμός υδάτων, ε, ίδρευση και το καθεξής ε, ε, έχουν πολύ μεγάλη σημασία για την καθημερινή ζωή του πολίτη. Ο κίνδυνος λοιπόν είναι όντως αυξημένος. Από την έκθεση του Ελεκτικού Συνεδρίου βλέπω ότι οι δημόσιες προμήθειες έχουν περιθώριο σφάλματος υψηλού, γιατί υπάρχει μεγάλος, επειδή υπάρχει μεγάλος κίνδυνος και διαφθοράς και αδυναμία λίγο πολύ ελέγχου του πλαισίου του νομικού. Άρα, οι δράσεις αυτές αναπτύσσονται βέβαια στα κράτη-μέλη και τα κράτη-μέλη έχουν καθήκον να ελέγξουν στο δικό τους πεδίο ερμεδιοτήτων αν υπάρχουν κίνδυνοι, αλλά υπάρχει και η ανάγκη της συνεργασίας μεταξύ των ελεγκτικών αρχών, άρα είναι συνδράμουσα η αρμοδιότητα και επίσης είναι χρήσιμο σε πεδονότερο σε εθνικό αλλά και περιφερειακό οι αρμόδιες αρχές να συνεργάζονται και να ανταλλάσσουν απόψεις προς τις καλύτερες ε, ε μεθόδους για την αντιμετώπιση των κινδύνων τη διαφθορά. Αυτό το έχουμε κάνει ήδη με διάφορα σεμινάρια. Ξέρετε ότι σε ευρωπαϊκό επίπεδο υπάρχει οργάνωση των περιφερειακών αρχών ελέγχου με τα περιφερειακά συνέδρια αλλά και με άλλα χωρών εθνικά συνέδρια Ισπανίας, Γερμανίας, Ρώσιας κλπ. Και εκεί ιδιαίτερη σημασία δίδεται στην αντιμετώπιση ευθόρας στο υλικό το οποίο επεξεργαζόμαστε. Οι δημόσιες αγορές είναι ο κύριος, η κύρια πηγή της διαφθοράς και υπάρχει βέβαια και η σύγκρουση συμφερόντων ή η υπεξαίρεση ε, δημοσίου χρήματος από αυτούς τους δημόσιους λειτουργούς οι οποίοι χρησιμοποιούν τα κρατικά κονδύλια για ίδιο συμφέρον. Έτσι λοιπόν έχουμε συνεργασία και πρέπει να έχουμε συνεργασία με τα κράτη-μέλη τα οποία θα πρέπει να εισαγάγουν στην ένωμη του τάξη το διατακτικό εκείνο που θα είναι παρκές για την διάγνωση και την καταπολέμηση της ε, απάτης από τις εθνικές αρχές, πάντα, όχι σε ευρωπαϊκό επίπεδο, πρέπει να υπάρχει συνεργασία μεταξύ των ελεκτικών ε, θεσμικών οργάνων και σε επίπεδο Επιτροπής Επαφής, αλλά και μέσω εθνικών, ε, ε, μέσω επαγγελματικών οργανώσεων που εκπροσωπούν και επίσης βέβαια χρειάζεται η ύπαρξη των μέσων αυτών των νομικών για την καταπολέμηση της διαφθοράς. Αναφερθήκα ιδιαίτερα στην παρουσία μου στην προβυγγία Άλπης Ροδανός και Ανιακτή, γιατί θεώρησα ότι ήταν η θέση μου αυτή τέτοια που υποχρέωνε να κοιτάξω περιπτώσεις προληπτικά όπου θα μπορούσε να υπάρξει διαφθορά. Γιατί αν κάνουμε έλεγχο με το τυπικό, με το τυπικό μόνο, δεν βρίσκουμε τίποτα. Έλεγχο κάνουμε όταν ξέρουμε που μπορούμε να εντοπίσουμε διαφθορά, όταν είμαστε ήδη υποψιασμένοι από κάποιες καταγγελίες και κάποιες καταγγελίες της Όλαφ εκπλήσουμε που εμφανίζονται ως μη ευσταθείς. Αλλά πρέπει να πω ότι και εγώ πολλές φορές βλέπω ότι οι καταγγελίες που φτάνουν μέχρι εμένα περί τις 80 το έτος, ε, αρκετές από αυτές, κάποιες από αυτές δεν έχουν να κάνουν με την ουσία της διαφθοράς. Μπορεί να μιλάει ένας πολίτης για κάτι που τον ενδιαφέρει, αλλά η διαφθορά, η, η στρέβλωση διαδικασιών για την ανάθεση, η, διείσδυση οργανώσεων μαφιώστικου τύπου σε ορισμένους τομείς ανάθεσης έργου, ε, εγκληματική δηλαδή η δράση, δεν είναι ορατή για τον πολίτη. Αυτά λοιπόν τα οποία αναφέρθηκαν για τον τρόπο με τον οποίο τα εθνικά αλλά και το Ευρωπαϊκό Ελεκτικό Συνέδριο μπορούν να συνεργαστούν στο μέλλον. Φυσικά και χρειάζεται περαιτέρω ανάπτυξη, η απάντηση είναι γνωστή. Στην απάντηση όμως αυτή πρέπει να δώσουμε σάρκα και οστά για την τρίτη σας ερώτηση και την ε, ε, βελτίωση του επαγγελματισμού. Στο ελεκτικό συνέδριο υπάρχει, από ό,τι γνωρίζω, ε, δυνατότητα και μηχανισμός κατάρτισης πολύ αναπτυγμένος, ώστε κανείς να βελτιώσει τις γνώσεις του. Είναι κάτι το οποίο ασφαλώς χρειάζεται για κάθε ελεγκτική αρχή να είναι κανείς δηλαδή πάντοτε ε, με τα μάτια και τα αυτιά ανοιχτά, στις νέες μεθόδους εργασίας, στις νέες τεχνολογίες και αν κανείς δεν ανήκει ήδη στον τομέα έχει να μάθει αρκετά ή πρέπει να στηριχθεί σε εξωτερική υποστήριξη. Αναφερθήκατε στις ευρωπαϊκές εταιρικές σχέσεις με χώρες ε, του Νότου, κυρίως της Αφρικής, Βόρειας Αφρικής. Έχω συνεργαστεί πολύ μαζί τους, διότι η Γαλλία συντονίζει τις δραστηριότητες στο πλαίσιο του γαλλόφωνου κόσμου. όπου είναι πολύ δραστήρια γιατί και προσφέρει υποστήριξη αλλά και ε, συμβουλές ακόμη σε ε, θεσμούς στις χώρες αυτές που ακόμη δεν έχουν εδρεωθεί και δεν έχουν βρει τη θέση τους. Πολλές φορές δυσκολεύονται να βρουν στήριξη, ούτε καν το κοινοβούλιο δεν είναι σε θέση να τα υποστηρίξει. Άρα είναι έναντι της εκτελεστικής εξουσίας που μπορεί ακόμα και να τους απειλήσει, να τους εξαφανίσει, να τους αναδιοργανώσει κατά τρόπο να αποδυναμωθούν και να χάσουν ε, κάθε δυνατότητα λειτουργία, πάρα πολύ δύναμη και εκτεθειμένοι. Ένα ενδιαφέρον κριτήριο της δημοκρατίας είναι το γεγονό της δημοσίευση των εκθέσεων του ελεγκτικού συνεδρίου. Ε, αυτό και μόνο είναι ένας σοβαρός δείκτης. Υπάρχουν χώρες που δημοσιεύουν τις εκθέσεις αναλυτικά, άλλες που δημοσιεύουν τι εκθέσει. συνοπτικά, ενώ άλλε που δεν δημοσιεύουν καθόλου. Και ενδιαφέρον ήταν ότι μόλις ξέσπασε η επανάσταση στην Τινησία, ε, βγήκαν στο διαδίκτυο μέσα σε μέρες οι ε, εκθέσεις του Ελεκτικού Συνεδρίου, ενώ μέχρι τότε μόνο συνοπτικά δημοσιεύονταν από την, ε, την Ισία. Άρα λοιπόν υπάρχει αυτή η ανάγκη και της εδραίωσης της πρακτικής μέσω συνεργασίας, αλλά όχι μόνο με τα δυτικά κράτη, αλλά και μεταξύ του συνεργασία. Εγώ έχω πολύ υποστηρίξει την συνεργασία νότου-νότου, όπως λέμε. Ε, στο Μαρόκο Φερρυπίν υπάρχει ένα σύστημα μεθοδολογία ε, κατάρτισης για το ελεκτικό συνέδριο, ήδη πολύ αναπτυγμένη και στην οποία συμμετέχουν πολλοί συνάδελφοι των ε, μαροκινών συναδέλφων μας από την υποσαχάρια Αφρική αλλά βέβαια είναι πολύ σημαντικός ο ρόλος ε, της Ευρώπης, όχι μόνο ως χρηματοδότη φυσικά, αλλά και για να βοηθήσει αυτά τα μικρά όργανα να αναπτυχθούν, τους θεσμούς αυτούς να αναπτυχθούν, αλλά και να ενσωματωθούν σε ένα δίκτυο που με τις μεγάλες αρχές και της ανεξαρτησίας και της υψηλής, ε, ε, του υψηλού επαγγελματισμού και της διαφύλαξης του ελεκτικού ρόλου πρέπει να τους υποστηρίξει. Και βέβαια όταν ε, κάτι πάει στραβά μπορεί να αποστέλλεται ένα μήνυμα στις τοπικές ε, ή στις εθνικές αρχές για να καταλάβουν ότι δεν επιτρέπεται έτσι. Εγώ το είδα αυτό σε ένα συγκεκριμένο παράδειγμα, όταν παρολίγων να αναδιοργανώσει ο πρόεδρος της Ενεγάλης, μειώνοντας τις εξουσίες του, το ελεγκτικό συνάδριο. Ο εκπρόσωπος λοιπόν του, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Διεθνούς Ταμείου και της Παγκόσμιας Τράπεζας, αντέδρασαν με υποστήριξη ολόκληρο του γαλλόφωνου δικτύου και ιδιαίτερα της Γαλλίας. Η συνεργασία μεταξύ Ελεγκτικού Συνεδρίου και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι για μένα κάτι το φυσιολογικό. Και γιατί η Γαλλία δεν έχει κοινοβουλευτικό σύστημα στον έλεγχο των δημοσιονομικών. Το ελεγκτικό συνέδριο δεν είναι Βέβαια δεν είναι υπηρεσία του Κοινοβουλίου όπως στις ΗΠΑ, αλλά δεν έχει και προνομιούχο δεσμό μέσω ενό γενικού λογιστή όπως συμβαίνει, δημοσιονομικού ελεκτή όπως συμβαίνει στο Ηνωμένο Βασίλειο. Δηλαδή ακολουθεί την ε, μεθοδολογία των ε, κοινοβουλευτικών συστημάτων. Από την αρχή της διαδρομίας μου πάντως από το 1984 ε, βλέπω να ενισχύονται οι δεσμοί μεταξύ ελεκτικού συνεδρίου και κοινοβουλίου αίτημα του ελεγκτικού συνεδρίου, ώστε και το Κοινοβούλιο να αποτελεί φορέα μεταβίβασης των παρατηρήσεων του ελεγκτικού συνεδρίου και ενισχύοντάς να τις μεταδίδει στην εκτελεστική εξουσία και να ε, ενημερώνεται για τις παρατηρήσεις και τους, τις εκθέσεις. Από την δημοσιονομική μεταρρύθμιση στη Γαλλία το 2006 ενισχύθηκε ακόμη περισσότερο αυτή η σχέση γιατί το Κοινοβούλιο είχε και πιο σαφείς ε, εξουσίες για τον έλεγχο και τη διαδικασία του προπολογισμού. Ταυτόχρονα όμως είχε και τη δυνατότητα που είχε και πιο πριν αλλά ενισχύθηκε στην πράξη αυτή η δυνατότητα να ζητεί έρευνες από το ελεκτικό συνέδριο. Έρευνες οι οποίες τώρα αντιστοιχούν στο 15% των δραστηριοτήτων της, ε, του ελεκτικού συνεδρίου με βάση τον προγραμματισμό βεβαίως. Ε, αυτό όμως πάει πολύ καλά και επιτρέπει στο ελεγκτικό συνέδριο να έχει την επικοινωνία του με τις κοινοβουλευτικές αρχές χωρίς να υπάρχει ένας συγκεκριμένο συνομιλητής, αλλά τέσσερις διαφορετικές κοινοβουλευτικές επιτροπές και από τα δύο σώματα, την Ανω και την Κατοβουλή. Φυσικά χρειάζεται ο συντονισμό ώστε να αντιστοιχούν οι έρευνες ε, με τις ανάγκες και αυτό και για το Ευρωπαϊκό Ελεκτικό Συνέδριο στις Ηνωμένες Πολιτείες τους ή άλλως ε, πρέπει και είναι άγραφος νόμος να ε, ικανοποιεί τους όρους της εντολής του το Ελεκτικό Συνέδριο στις έρευνές του, να είναι ανεξάρτητο, να μην μεροληπτεί να εκπληρεί το έργο του γέρος, Όλοι αυτοί οι όροι που ε, ε, πληρούνται εν γέννη. Βέβαια μια έρευνα υπερβολικά επαχθής μπορεί να χρειαστεί περισσότερο χρόνο και να καθυστερήσει, αλλά εν γέννη η συνείδηση και η ανάλυση των ευρωπαϊκών ζητημάτων πιστεύω ότι θα κέρδιζαν και θα αναπτύσσονταν περισσότερο εάν ήταν περισσότερο από τα Εθνικά Ελεκτικά Συνέδρια, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και οι λοιποί φορείς, να διαρευνούν ζητήματα που έχουν να κάνουν με ευρωπαϊκά κονδύλια. Εάν λοιπόν, και όχι γίνει αυτό ήδη σε μια-δύο περιπτώσει, εάν λοιπόν είχε καλύτερη επικοινωνία το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με τα Εθνικά Κοινοβούλια για να προαγάγει τη δουλειά στα διαρθρωτικά ταμεία ή στι ευρωπαϊκέ πολιτικέ, η στις ευρωπαϊκές πολιτικές, η δουλεια των ελεκτικών αρχών θα είχαν ε, μπορέσει να προσανατολιστούν περισσότερο προς τα ευρωπαϊκά θέματα. Σας ευχαριστώ και τώρα να περάσουμε στο δεύτερο γύρο ε, ερωτήσεων. Δεν ξέρω αν υπάρχουν άλλες ερωτήσεις ή κατά πόσο σας έπεισαν ε, πλήρως οι απαντήσεις. Ο κύριος Σουντή, θέλει το λόγο. Ευχαριστώ. Ε, θα ήθελα και εγώ κύριε Λαμάρκα και εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος να σας καλωσορίσω θερμά και να σας ευχηθώ σε την στην Επιτροπή μας. Ε, χαίρομαι γιατί είναι πολύ ποιοτική υποψηφιότητα από την ε, γαλλική κυβέρνηση για, το, για τη θέση του μέλους του Ελεκτικού Συνεδρίου. Θα ήθελα να σας ρωτήσω για το πώς βλέπετε τις ε, σχέσεις μεταξύ Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου και Εθνικών Φορέων Ελέγχου. Ε, είναι ένα θέμα που έθιξε και προσωπικά στην Επιτροπή μας εδώ και πάρα πολύ καιρό. Γιατί θα πρέπει να ισορροπήσουμε την ε, επιθυμία της Επιτροπής να λαμβάνουμε από τι εθνικές κυβερνήσει μια εθνική δήλωση, κάτι που δεν θα λάβουμε ποτέ πιστεύω, και τις χρησιμότητάς της από τους εθνικούς φορείς ελέγχου. Γιατί είναι σημαντικό και το δικό τους ελεγκτικό έργο στην αλυσίδα του ελέγχου, ενώ μια εθνική δήλωση αξιοπιστίας έχει πολύ περιορισμένο τελικά ενδιαφέρον. Ε, σε ό,τι αφορά την κοινή χρήση, την κοινή διαχείριση μάλλον, ποια είναι η γνώμη σας, γιατί σε ό,τι αφορά την κοινή διαχείριση έχουν γίνει πολλά λάθη το Συμβούλιο δεν ενδιαφέρεται και πολύ για το θέμα της απαλλαγής, ενώ ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση το ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει την ιδιαιτερότητα ε, να έχει δύο αρχές αρμόδιες για την νομοθεσία, δύο συνομοθέτες, το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο. Ε, σε κάθε δημοκρατία το κοινοβούλιο έχει και τον πολιτικό έλεγχο και τον δημοσιονομικό. Εμείς είμαστε ουσιαστικά ο βραχίωνας του δημοσιονομικού ελέγχου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Από τις απαντήσεις σας κατάλαβα ότι συμφωνείτε για τις ως προς την χρησιμότητα εθνική φορείς ελέγχου να συμμετέχουν στον έλεγχο της κοινή ε, διαχείρισης, αλλά με σημαντικότερε σημαντικότερες επιφυλάξεις από αυτές που είχε ο κ. Μιλιώνης, που είπε ότι οι εθνικοί ελεγκτικοί φορείς θα πρέπει να ε, επεμβαίνουν στο όνομα και για λογαριασμό του Ευρωπαϊκού Ελεκτικού Συνεδρίου. Κάτι που είναι αδύνατο, γιατί οι εθνικοί ελεκτικοί φορεί εμπίπτουν σε μια εσωτερική ενόμη τάξη, εθνική. Οπότε εμεί, ε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, θα πρέπει να συνεργαζόμαστε με τα εθνικά κοινοβούλια, ώστε με τι κυβερνήσει των κρατών μελών να ε, κινητοποιήσουμε αυτή τη διαδικασία ώστε να ενταχθούν και οι εθνικοί ελεκτικοί φορείς στην ευρωπαϊκή αλυσίδα ελέγχου. Για αυτή την κοινή διαχείριση λοιπόν, ε, θα ήθελα να σας ρωτήσω ε, πιστεύετε ότι η χρησιμότητα των εθνικών ελεκτικών φορέων που θα μπορούσαν να δίνουν όχι στο Ευρωπαϊκό Ελεκτικό Συνέδριο αλλά στην κυβέρνησή τους ε, ε, δηλώσεις ελέγχου για την κοινή διαχείριση έχει νόημα και το Συμβούλιο που δίνει στην διαδικασία απαλλαγής της βεβαιώσεις τα πιστοποιητικά ελέγχου για το σύνολο. Επίσης, σε ό,τι αφορά τον έλεγχο των διακυβερνητικών δράσεων, με την κρίση κυβερνήσεις και αρχή κρατών και κυβερνήσεων ε, συμφώνησαν για πολλές διακυβερνητικές δράσεις χρησιμοποιώντας τους κοινοτικούς μηχανισμούς. Και εκεί έχουμε ακόμη και μεταξύ μας ε, διάσταση απόψεων. Εγώ είμαι κάπως ε, απομονωμένος ό,τι αφορά την απαλλαγή στο Συμβούλιο. Ε, το Ευρωπαϊκό Ελεκτικό Συνέδριο ε, ε, ουσιαστικά τίποτα δεν λέει. 20 γραμμές μόνο παρατηρήσεων για το Συμβούλιο και συστηματικά δύο χρόνια ε, αρνούμαστε την απαλλαγή στο Συμβούλιο χωρίς να ξέρουμε ποιες είναι οι συνέπειες, οι κυρώσεις αυτής της άρνησης της απαλλαγής. Ενώ για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχουμε 200-300 σελίδες παρατηρήσεων και εκεί χορηγούμε την απαλλαγή. Επίσης έχω μια δήλωση από το Συμβούλιο για την δήλωση ε, ε, του, του Συμβουλίου που είναι ε, πραγματικά διανόητη. Δεν ξέρω αν τελικά είναι θετική ή αρνητική η γνώμη του Συμβουλίου σε ό,τι αφορά αυτή τη δήλωση εξοπιστίας. Τώρα, σε ό,τι αφορά την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερική Δράση, μα λέτε έχετε δικαίωμα να ελέγχετε το διοικητικό τμήμα, αλλά όχι το επιχειρησιακό τμήμα των δράσεων τη ΑΕΔ. Όλε αυτέ λοιπόν οι διακυβερνητικέ δράσει από ποιο θα ελέγχονται, από τα Εθνικά Κοινοβούλια, από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, από το Ευρωπαϊκό Ελεκτικό Συνέδριο, από τα Εθνικά Ελεκτικά Συνέδρια, τους Εθνικούς Ελεκτικού Φορείς. Ήμως θα πρέπει όλα αυτά να τα ξανασυζητήσουμε ε, με τι κυβερνήσει. Εμένα με ενδιαφέρει ο έλεγχο αυτών των επιχειρήσεων, ε, των διακυβερνητικών δράσεων, αν ε, όχι από εμά τουλάχιστον από τα Εθνικά Κοινοβούλια. Και πραγματικά είμαστε ε, σοκαρισμένη με την άρνηση των κυβερνήσεων να ελέγξει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τον Ευρωπαϊκό ε, Μηχανισμό ε, Ελληνικής που έχει πρικοδοτηθεί με 700 δισεκατομμύρια ευρώ. Είναι ανήκουστο. 700 δισεκατομμύρια ευρώ που θα τα ελέγχει μόνο ένας ιδιωτικός ελεγκτής. Αν είναι δυνατόν. Το Ευρωπαϊκό Ελεκτικό Συνέδριο τελικά έδειξε, δέχτηκε μία μορφή παρουσίαση, παρατηρητών. Αυτό πραγματικά είναι άλλο αλλοπρόσαλο. Είναι γελίο. Σε τέτοιου είδου ε, διακυβερνητικά όργανα ε, που ελπίζουμε ως ονόπο να γίνουν κοινοτικά, θα πρέπει να εξασφαλίζεται έλεγχος και δημοσιονομικός, ε, δημόσιος, αλλά και πολιτικός ταυτόχρονα. Σας ευχαριστώ πολύ. Αν δεν υπάρχουν άλλες ερωτήσεις, σε αυτή τη φάση θα ήθελα να δώσω το λόγο στην κυρία Δαμάρκη για να κάνει τα καταλητικά τη σχόλια. Το θέμα της ε, μεικτής της κοινή διαχείρισης ε, και του καλύτερου ελέγχου των κοινοτικών ε, δράσεων είναι πολύ περίπλοκα θέματα. Έχουν δοθεί πολλές και διάφορες απαντήσεις και παραμένουν ακόμη πολλά ερωτηματικά. Γιατί και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Ευρωπαϊκό, Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο έχουν δηλώσει ότι διάφορα, διάφοροι μηχανισμοί όπως του ολοκληρωμένου ελέγχου δεν λειτουργούν σωστά, αλλά ούτε και η δήλωση αξιοπιστίας είναι μια ικανοποιητική απάντηση. Οπότε έχουμε περιπτώσεις όπου ε, επιχειρήσει δράσεις που γίνονται σε μια χώρα υπάγονται στον έλεγχο αυτής της χώρας και το ελεκτικό συνέδριο ελέγχει την ε, εφαρμογή ε, ή όχι την των εθνικών ελεγκτικών συστημάτων και των απο... της αποτελεσματικότητας των ε, ελεγκτικών φορέων. Οπότε έχουμε ένα μηχανισμό που από άποψη ελέγχου ε, ε, προσφέρει κάποια επαγγελματικά εχέγγυα. Τώρα, πού έγκυται η δυσκολία. Η δυσκολία έγκυται στο ότι δεν ξέρουμε σε ποιο βαθμό τα κράτη-μέλη είναι ικανά να ελεγχθούν για την εύρυθμη όχι λειτουργία αυτών των μηχανισμών ως προς και δήλωση αξιοπιστίας. Στο μέτρο τώρα που τα, οι ελεκτικοί φορείς ε, δεν είναι εθνικοί και δεν έχουν ε, αρμοδιότητες για τον κοινωτικό προϋπολογισμό, είναι δύσκολο να ενταχθούν σε μια ελεκτική διαδικασία, εκτός και είναι ανεξάρτητα από το Ευρωπαϊκό Ελεκτικό Συνέδριο, γιατί θα είμαστε σε ένα μηχανισμό που ο βασικός ελεκτής θα στηρίζεται στο έργο ενός δευτερεύοντος ε, λογιστού, λογιστού συγγνώμη, ελεγκτού. Και δεν νομίζω ότι μια τέτοια θεσμική διάρθρωση ανταποκρίνεται στη, στα ευρωπαϊκά πρότυπα. Υπάρχει λοιπόν ένα νομικό εδώ σκέλος, αλλά και ένα τεχνικό σκέλος. Την εφαρμογή δηλαδή των διεθνών προδιαγραφών ελέγχου. Εγώ έχω πήρει κυρίως από το Γαλλικό Ελεκτικό Συνέδριο. Εκεί δεν έχουμε, ε, με εξαίρεση την πιστοποίηση των λογαριασμών, που είναι ιδιαίτερη δραστηριότητα, δεν έχουμε ε, την ετήσια βάση, έχουμε περισσότερο πολυετή βάση. Πρόσφατα είχαμε την ε, έκθεση του 2012 με ανάλυση της διαχείρισης του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου στη Γαλλία. Και μάλιστα αυτό έγινε στα πλαίσια ενός εξαετούς προγραμματισμού. Δεν γίνεται με αιτήσια βάση, οπότε υπάρχει ένα πρόβλημα διάρθρωση μεταξύ μιας ε, μεθοδολογίες ετήσιας πιστοποίησης ή ετήσιας απαλλαγής για τον προϋπολογισμό και μίας μεθοδολογίας που έχει πολύ πιο πολυετή βάση και στηρίζεται κυρίως στον έλεγχο των επιδόσεων. Οπότε, στα πλαίσια του ελέγχου επιδόσεων και των ειδικών εκθέσεων και από αυτή την άποψη ίσως θα μπορούσαμε να υιοθετήσουμε και, και την προσέγγιση του Ευρωπαϊκού Ελεκτικού Συνεδρίου ε, για ένα ε, κύκλο, συνολικό κύκλο προγραμματισμού, γιατί το δημοσιονομικό πλαίσιο της Ένωσης ε, προσφέρεται για κάτι τέτοιο, οπότε θα ήταν μια προέκταση των ειδικών αιτήσεων εκθέσεων και θα ήταν ένα συμπλήρωμα της, της απαραίτητης ε, λειτουργίας και της ετήσιας απαλλαγής. Είναι λοιπόν και νομικό και μεθοδολογικό το πρόβλημα, όχι ανεπίλητο, αλλά θα πρέπει να δούμε πού είναι χρησιμότερο ο καθένας. Σε ό,τι αφορά τώρα τις διακυβερνητικέ δράσει και επιχειρήσει. εδώ το διακύβευμα ε, είναι, όπως πολύ σωστά είπατε γιατί αναφερθήκατε στην ΕΙΕΔ, είναι το θέμα του ελέγχου και εκεί υπάρχει πολύ μεγαλύτερη περιπλοκότητα γιατί έχουμε νέα χρηματοδοτικά μέσα και μηχανισμούς. Γιατί έχουμε μια σειρά μηχανισμών, μερικοί αφορούν την Ευρωζώνη, άλλοι την Ευρωζώνη με επιπλέον κάποια μέλη, άλλοι αφορούν το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μερικοί μηχανισμοί είναι διακυβερνητικοί, μερικοί συμπεριλαμβάνονται στην συνθήκη, άλλοι εμ, κανονικά θα έπρεπε να εμπίπτουν στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο, αλλά ακόμη δεν έχουν ενταχθεί. Πρόκειται για ένα περίπλοκο νομικό πλέγμα. Βέβαια, η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, στην κρίση έδρασε άμεσα και αποτελεσματικά. Βλέπουμε λοιπόν όμως ότι όλοι αυτοί οι μηχανισμοί είναι σχετικά νομιόμορφοι, ε, ετερογενείς, ξεφεύγουν από το νομικό πλαίσιο των συνθηκών, διαφεύγουν του κοινοβουλευτικού ελέγχου και του ελέγχου των ε, εθνικών ελεκτών ή του Ευρωπαϊκού Ελεκτικού Συνεδρίου. Ακόμη και ο ρόλος του ελεκτικού συνεδρίου είναι περιορισμένος και πολύ μικρός. Και μάλιστα το, το γερμανικό μέλος του ελεκτικού συνεδρίου συμμετέχει στο ελεκτικό όργανο του Μηχανισμού Σταθερότητας αλλά, όπως είδαμε και σε πολλές χώρες και στη Γαλλία, βλέπουμε ότι είναι πολύ δύσκολο να ενταχθεί το ελεκτικό συνέδριο στον δημοσιονομικό μηχανισμό, γιατί το ελεκτικό συνέδριο ελέγχει την Τράπεζα της Γαλλίας. Υπάρχει αυτή η δυνατότητα, δεν είναι πάντα εύρυθμη κατάσταση, αλλά δεν έχουν όλα, όλοι οι ελεκτικοί φορείς τη δυνατότητα ελέγχου των χρηματοδοτικών φορέων. Έχουμε όμως τώρα κοινωτική αρμοδιότητα για νομισματική πολιτική. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει δυνατότητα και ελέγχου των ε, χρηματοοικονομικών μηχανισμών, των δικτύπου τους, της χρήσης των κονδυλίων και σε συνεργασία με τα κράτη-μέλη θα πρέπει να δούμε πώς αξιοποιούνται αυτά τα κονδύλια. Γιατί με έναν κοινοτικό προϋπολογισμό ετής 140 δις ε, έχουμε 700 δισεκατομμύρια αλλού που κάποια στιγμή θα ενεργοποιηθούν για να χρησιμοποιηθούν στις χώρες. Εγώ ανήκω σε ένα θεσμικό όργανο με ευρύτατες αρμοδιότητες. Ανέκαθεν όμως ε, ε, φροντίσαμε όχι μόνο να εμπεδώσουμε τις αρμοδιότητες μας, αλλά και να τις διευρύνουμε. Γι' αυτό και το Γαλλικό Ελεκτικό Συνέδριο ε, έχει καταφέρει να διευρύνει τις αρμοδιότητες του. Οπότε έχουμε και βελτίωση της ποιότητα, αλλά και τη ε, δημοκρατικότητα του ελέγχου. Πιστεύω ότι ε, θα πρέπει και οι, οι του Ευρωπαϊκού Ελεκτικού Συνεδρίου να είναι πιο ευρειε και η παρουσία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πιο σταθερή και δεδομένη. Αγαπητοί συνάδελφοι, έχουμε αργήσει 40 λεπτά, έχουμε καθυστερήσει. Ε, να δώσουμε τον λόγο στην κυρία Οντή για μια τελική, τελευταία ερώτηση, μια παρατήρηση, ελπίζω. Δεν είναι την ερώτηση. Απλώ θα ήθελα να εκφράσω τη δίπλα μου για την αποχώρηση του Μισελ Κρετάν που ήταν πολύ εξαιρετικό μέλο του συνεδρίου αλλά και του κ. Μπελενκό ο οποίο ήταν ο πρώτο που με μίλησε στι χαρέ του δημοσιονομικού ελέγχου. Ε, ε, Σα ευχαριστώ πάρα πολύ και έτσι μπορούμε να ολοκληρώσουμε την, ακρίωση, ακρόαση τη κυρία Λεμάρκ. Σα ευχαριστώ πολύ. Στο επανειδήν. So, Σας ευχαριστώ πολύ και θα ήθελα να περάσουμε πάρα αυτά ε, στον επόμενο υποψήφιο. Να σας καλέσω στο βήμα. Συνάδελφοι, συνάδελφοι, έχουμε πρόβλημα με το χρόνο. Θα πρέπει να είμαστε λίγο πιο συνοπτικοί, λίγο πιο, περιορισμένοι. Δεν είχα περιορίσει και στις προηγούμενες δύο ακροάσεις ε, τον χρόνο, 10 και 25 πρέπει να έχουμε ολοκληρώσει. 11 ε, έχει πάει η ώρα. Έχουμε καθυστερήσει. Σας παρακαλώ πολύ να μην γίνει βολεί της ακρόασης. Από σας εξαρτάται. Δεν θα ήθελα να ακούσω παράπονα εκ των υστέρων. Κυρίες και κύριοι, σε αυτή την ε, φάση θα ήθελα να καλωσορίσω τον υποψήφιο Ανρι Γκρέτζεν, ο οποίος και προτάθηκε από τις αρχές του Λουξεμβούργου. Κύριε Γκρέτζεν, είσαστε παλιά καραβάνα. Γνωρίζετε πώς κινούνται οι διαδικασίες. Θα ήθελα να σας καλέσω να Απευθύνεται την αρχική σας παρέμβαση ε, σε σχετική συντομία, αν θέλετε. Ίσως να μην ξεπεράσετε τα 10 λεπτά για να μπορέσουμε μετά να ακούσουμε και τις ερωτήσεις. Έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να μην σας ε, πάρω ούτε 10 λεπτά. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, πριν από έξι χρόνια, η δική σα Επιτροπή καταρχά και το Κοινοβούλιο στην Ολομέλειά του εν είχατε την κατοσύνη να γνωμοδοτήσετε θετικά ω προ την υποψηφιότητά μου ω μέλο του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου. Ήταν πολύ σημαντική αυτή η ψηφοφορία για μένα με ε, δεδομένο ότι η καλή συνεργασία μεταξύ του Ελεγκτικού Συνεδρίου και του Κοινοβουλίου αποτελεί τη βάση του συστήματο ελέγχου των δημοσιονομικών τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Από την 1η Ιανουαρίου του 2008 μπόρεσα έτσι να συμβάλλω στην προστασία των δημοσιονομικών συμφερόντων των πολιτών της Ένωσης, στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και τα δημοσιονομικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στη ασφάλιση ότι τα ε, χρήματα αυτά θα αξιοποιούνται κατά τρόπο αποτελεσματικό και χρήσιμο για την υλοποίηση των ευρωπαϊκών στόχων ε, με σεβασμό των κανόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα έξι τελευταία χρόνια ε, το ελεγκτικό συνέδριο μεριμνήσε για την διατύπωση ανεξάρτητων εκθέσεων, γνωμοδοτήσεων και θέσεων με σεβασμό της ανεξαρτησίας και των διεθνών προδιαγραφών δημοσιονομικού ελέγχου, με στόχο να υποστηρίξει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην αναζήτηση προστέμενης αξίας για τα ευρωπαϊκά κονδύλια προς το συμφέρον του Ευρωπαίου πολίτη. Η και η διακυβέρνηση του ελεκτικού συνεδρίου προσαρμόστηκαν η θέσπιση τμήματων επέτρεψε τον εξορθολογισμό της διαδικασίας λήψης των αποφάσεων σύμφωνα με το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο στο μέλλον θα πρέπει πιστεύω να ενισχυθεί ακόμη περισσότερο η υποχρέωση της λογοδοσίας και η υποστήριξη του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου στην εποπτεία της εκτέλεσης του Ευρωπαϊκού Προπολογισμού. Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο θα πρέπει βράχει πρόθεσμα να αναλαμβάνει μέτρα να έχει να αναλαμβάνει μέτρα για την επαλήθευση της λειτουργίας του πολιτού δημοσιονομικού πλησίου και ε, να καταγράφει στην έκθεση, στη δεσία έκθεση της παρατηρήσης του. Επίσης η αξιολόγηση αποδοτικότητας είναι πολύ σημαντική. εμπνεώμενη βέβαια από τις παρατηρήσεις των εμπλεκομένων ε, θα προβούμε τη σχετική μελέτη και πριν ε, κλείσω την εισαγωγική μου παρέμβαση κύριε Πρόεδρε θα ήθελα να ευχαριστήσω τα μέλη της Επιτροπής σας για την εξαίρετη συνεργασία που είχαμε τα έξι τελευταία χρόνια και ιδιαίτερα τους εισηγητές των εκθέσεων ελέγχου και τους εισηγητές για τις εκθέσεις με τους οποίους είχα τη χαρά και τιμή συνεργαστώ. Σας ευχαριστώ πολύ και ελπίζω ότι θα μου επιτρέψετε κύριε Πρόεδρε και κύριοι, βουλευτές να, μου, να, να συνεχίσω αυτή τη τόσο καλή συνεργασία σε μια ενδεχόμενη δεύτερη εντολή. Πρώτη έχει το λόγο η κυρία Γιάλα Σέντερ. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα είμαι πολύ σύντομη. Σας καλωσορίζω λοιπόν και σας, κύριε Γκρέτεν. Σας γνωρίζουμε. Συχνά έχουμε ανταλλάξει απόψεις, αλλά θα ήθελα να σας θέσω παρ' αυτά μια ερώτηση, γιατί είμαι εισηγήτρια και με απασχολούν τα θέματα για το μέλλον του Ελεκτικού Συνεδρίου. Τα πέντε χρόνια λοιπόν που ήσασταν μέλος του Ελεκτικού Συνεδρίου βλέπω ότι ήσασταν υπεύθυνο για τέσσερα, τέσσερις εκθέσεις ε, ελέγχου. Ε, πρόκειται για πολύ περιπλοκές εκθέσεις και οι εκθέσεις ε, αυτές υποβλήθηκαν, τις γνωρίζω. Πείτε μας όμως Πώς προέκυψαν τα αριθμητικά στοιχεία. Δεν γνωρίζουμε επακριβώς τον τρόπο με τον οποίο εργάζεστε. Εξηγήστε μας λοιπόν τον τρόπο εργασίας σας, τον τρόπο εργασίας του ελεκτικού συνεδρίου. Σε ό,τι αφορά την περιφερειακή πολιτική τώρα. Γνωρίζετε ότι τα τελευταία χρόνια Έγινε μια σειρά συζητήσεων επί του θέματος αυτού και σε ό,τι αφορά τα αποτελέσματα που προέκυψαν. Πείτε μας λοιπόν, εξηγήστε μας. Αυτή, αυτά τα αποτελέσματα τα οποία δεν ικανοποιούν, από πού προήλθαν ε, και υπάρχει περιθώριο βελτίωση. Ευχαριστώ. Ποιο θέλει άλλο το λόγο, ο κ. Σοντή. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και ευχαριστώ, κύριε Ποτών, για την ε, Γκρέτον για την παρουσία σας. Είναι άλλε οι ερωτήσει από ό,τι βλέπω σχέση με τα νέα μέλη. Ναι, γιατί πρόκειται για ανανέωση. Όμω, ω Πρόεδρε, θα έπρεπε να διατυπώνουμε τα ίδια ερωτήματα και στου επανερχόμενου υποψηφίου και στου νέου. Για να δούμε. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ευχαριστώ πολύ, κύριε Γκρέτον για τι διευκρινήσει. Από τις 19 Απριλίου του 2012 είσαστε μέλος ε, του ειδικευμένου οργάνου για την δημοσιονομική σταθερότητα. Από το 2013 βλέπω έχετε αναλάβει. Έχουμε ταλαιπωρηθεί αρκετά σε σχέση με την Επιτροπή για, το, για την αντιμετώπιση της παρατυπίας και τη διάκριση της από τη διαφθορά... Γιατί ε, η Επιτροπή που έχει αναλάβει το θέμα αυτό, ε, στις του περιπτώσεις μας έλεγε ότι είναι παρατυπία, ήταν διαφθορά κτλ. Ερωτώ λοιπόν για αυτές τις παρατυπίες. Μπορείτε να μας πείτε δύο λόγια και κυρίως πώς βλέπετε την καταπολέμηση της απάτης. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε κυρία Οντή... και μετά ο κύριος Μούλντερ και η κυρία Γκρέσλα έχουν το λόγο. Σας ευχαριστώ πρόεδρε. Θα ήθελα να ρωτήσω και εγώ το Κατά την περίοδο που ο κύριο Γκέτεν ήταν μέλο ε, του Ανεκτικού Συνεδρίου, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τα Περιφερειακή Επιτροπή, δεν έχουμε δει σημαντική βελτίωση σε ό,τι αφορά τον έλεγχο των ε, δαπανών στις περιφέρειες. Θα μπορούσατε να μας συμβουλέψετε τι θα μπορούσαμε ως Κοινοβούλιο να πράξουμε προκειμένου να βελτιωθεί η κατάσταση αυτή θα πρέπει να επικεντρωθούμε πιο πολύ στην αρμοδιότητα και την ευθύνη των κρατών μελών. Πείτε μας ποιες ιδέες έχετε για το θέμα αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Γκρέσλη έχει το λόγο. Θα ήθελα να συνεχίσω από εκεί που σταμάτησε ο Γιάν. Υπάρχει μια ε, αναθεώρηση από ομοτήμου σε ένα peer review σε ό,τι αφορά την εργασία του Ελεκτικού Συνεδρίου. Πολύ ενδιαφέρον το έγγραφο. Επειδή αναπτύσσει το εξή, ότι θα μπορούσε να διακυβευθεί η ανεξαρτησία του Ελεκτικού Συνεδρίου από τις στενές σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εξηγήστε μας λοιπόν, είναι σημαντικό. Τι γίνεται σε ό,τι αφορά θέματα ανεξαρτησίας, πώς ενδυναμώνετε εσείς δε την ανεξαρτησία αυτή. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Δέσμη ερωτήσεων. Έχετε το λόγο για να απαντήσετε. Θα ήθελα καταρχάς να απαντήσω στην ερώτηση της κυρίας Σαγιάρα Σέντερ. Ο φόρτος εργασίας των διαφόρων μελών του συνεδρίου προχωρεί ανάλογα με, τις, με τη διαθεσιμότητα των ελεγκτών καταρχάς και το ενδιαφέρον των μελών. Πρέπει να πω ότι αυτός ο φόρτος είναι καταμερισμένος δίκαιο. Εγώ ήμουν αρκετά... Είχα, είχα σχετικά λίγη δουλειά, αλλά από την άλλη είμαι και εκφίσως ανυπόμονος και ίσως πίεσα περισσότερο τους ε, συνεργάτες μου και έτσι μπορέσαμε να ολοκληρώσουμε τέσσερις εκθέσεις με άλλη, μία πέμπτη η οποία προχωρεί σιγά σιγά προς την ολοκληρωσή της ε, για τα φυτόρια αυτά επιχειρήσεων τις θερμοκοιτίδες όπως λέμε. η οποία θα ενταχθεί στο κεφάλαιο 5 της θετής έκθεσης. Παραχώρησα το τμήμα αυτό στον κύριο Λαζάρο, το μεταξύ, τώρα λαμβάνει αυτό από το 2013. Έχω ορίστηκα οριστικά κοσμήτορας αυτού του δεύτερου τμήματος από τους συναδέλφους μου εξελέγην. Πολύ σημαντική βέβαια η τιμή που μου έγινε, αλλά από την άλλη δεν μπορώ να κρατήσω όλα τα καθήκοντα που είχα πριν, γιατί θα πρέπει να προεδρεύω των εργασιών του τμήματος αυτού. Ως πρόεδρος τμήματος. Ο κύριος Οντή αναφέρθηκε στις, ε, στην Επιτροπή Παρατυπιών, η οποία στο πλαίσιο του δικαστηρίου εργάζεται κατά περίπτωση Εγώ μια υπόθεση που αντιμετώπισα ήταν ενό εξωτερικού συνεργάτη που ερχόταν να, προσφέρει μαθήματα, να κάνει μαθήματα, μαθήματα τα οποία ακυρώνονταν γιατί ο, το μέρος του συνεδρίου ή οι συνεργάτες του που ήταν να κάνουν μάθημα είχαν ε, κάποιο κόλλημα και έτσι βρεθήκαμε αντιμέτωποι με το ερώτημα εάν θα πρέπει να αποζημιώνεται ο δάσκαλος αυτός ή όχι. Και όπως πρέπει να είναι η γυναίκα του Κέσσερα τίμια αλλά και να φαίνεται τίμια, το ελεκτικό συνέδριο αναζήτησε τις βέλτιστες πρακτικές και λύσεις και διαπιστώσαμε στο τέλος αυτής της μελέτης ότι το σφάλμα, τα λάθη ήταν, ε, εντοπίζονταν σε επίπεδο συνεδρίου και όχι παρόχου των υπηρεσιών αυτών. Για τον κύριο Μιούλτερ, ο οποίος έθεσε ένα ερώτημα λεπτό, διότι το συνέδριο δεν μπορεί να βελτιώσει την αποδοτικότητα. Η Επιτροπή, τα κράτη-μέλη, οι ιδιώτες πρέπει να το πράξουν αυτό. Και για να προσθέσω και στην ερώτηση, στην ερώτηση της κυρίας Γκρέσλε και να απαντήσω μαζί. Εμείς στο συνέδριο παραδείγματι, στο δημοσιονομικό κανονισμό, είχαμε διατυπώσει προτάσεις ώστε να ενισχυθούν οι παρεμβάσεις της Επιτροπής. Αν ένα κράτος μέλος μπορεί ε, ατιμωρητή να αντικαθιστά ένα σχέδιο με ένα άλλο, αν δεν υπάρχουν δηλαδή δημοσιονομικές συνέπειες, η Επιτροπή έχει δεμένα χέρια. Και θα έπρεπε, κατά τη γνώμη μου, να υπάρχουν σαφή κίνητρα ώστε τα κράτη-μέλη να ακολουθούν με προσοχή και να υλοποιούν με ευλάβεια τους φεκέλους για την αιτήσια έκθεση που κατέθεσε μόλις το ελεγκτικό συνέδριο. Καταγράφεται ότι 75% των σφαλμάτων εντοπίζονται σε περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο και το μεγαλύτερο μέρος των σφαλμάτων αυτών θα μπορούσαν σε επίπεδο εθνικό ή περιφερειακό να είχαν εντοπιστεί εάν είχαν κάνει σωστά τη δουλειά τους οι αρμόδιες αρχές. Εμείς ως ελεκτικό συνέδριο απλώς το διαπιστώνουμε αυτό. Δεν αισθανόμαστε την χαρά κάθε χρόνο, εδώ και 20 χρόνια τώρα, να σας ε, επιδίδουμε αρνητικό, αρνητική βεβαίωση. Πολύ θα θέλαμε να μπορούσαμε να πούμε στον Ευρωπαίο φορολογούμενο ότι μπορεί να κοιμάται ήσυχο και ότι το μέλλον του είναι καλύτερα, ότι όλα είναι οργανωμένα τέλεια. Δυστυχώ όμω δεν ισχύει αυτό και όσο δεν υπάρχουν σαφεί και αυστηροί ε, όροι, κυρώσει ουσιαστικά, όσο δεν υπάρχουν αυστηρέ κυρώσει και συγκεκριμένε κυρώσει, δεν μπορεί να βελτιωθεί η κατάσταση. Κυρία Γκρέσλε, εμένα θα μου απαντήσετε. Ναι, με συγχωρείτε κυρία Γκρέσλε. Σας διαβεβαιώ. Ήμουν αρμόδιος για το κεφάλαιο 5, ανάπτυξη περιφερειών, ενέργεια, μεταφορές. Ο Επίτροπος Κάλλας, με τον ε, κύριο Κάλλας, με τον Επίτροπο Κάλλας δεν έχω μιλήσει ποτέ, τουλάχιστον εγώ γνωρίζω, με τον Επίτροπο Έτιγκερ εδώ, δύο φορές μέσα στην Επιτροπή σας, αλλά και να έχω μια επαφή με έναν επίτροπο ή με έναν, ε, ένα μέρος ε, προσωπικού της Επιτροπής, αυτό δεν σημαίνει ότι επηρεάζομαι από αυτούς ε, στην διατύπωση της δρομοδοτησή μου. Ήδη έχουμε αρχίσει την έκθεση για το επόμενο έτος. Έχουμε τους ελεγκτές μας, οι οποίοι έχουν πάει στις διάφορες περιοχές. Ένας ελεγκτής Φερρυπίν που είναι στο... από το Λουξεμβούργο έχει πάει στη Ρουμανία. Ρουμανικά δεν ξέρει. Πρέπει να συνονεθεί στα αγγλικά. Πρέπει να κάνει ερωτήσεις. Συνήθως είναι νεαρός ελεγκτής. Μεταξύ 25 και 34-35 ετών. Ο οποίος συλλέγει πληροφορίες. Τι ερωτήσεις του, οι απαντήσεις δεν θα είναι κατά πάσα πιθανότητα σωστές. Θα χρειαστεί δηλαδή να αναστήσουμε συμπληρωματικές πληροφορίες. Στο πρώτο κομμάτι έχουμε ένα ποσοστό σφάλματος, το οποίο είναι πολύ υψηλό. Και μετά, στο δεύτερο τμήμα, το κατά αντιμολία θα λέγαμε ή κατά παραβολή, επαληθεύονται αυτές οι πληροφορίες και εκεί μειώνεται σημαντικά το ποσοστό του σφάλματος. ενόχληση αυτό να σημαίνει ότι κάνουμε αναθεωρούμε τη δουλειά του ε, ε, ε, ελεγκτή. Απλώς ότι εμείς ως ελεγκτικό συνέδριο κάνουμε πολύ μεγάλη προσοχή τη δουλειά μας. Δεν νομίζω δηλαδή ότι είναι δυνατόν να βρίσκομαι εδώ στην επιτροπή του Κοινοβουλίου και να μου πει ένας βουλευτής ότι έχει έρθει ένας ελεκτής μας σε για να κάνει έλεγχο και έχει κάνει κάτι το οποίο δεν ήταν σωστό, για να το πω έτσι. Δεν το δέχομαι αυτό με τίποτα. Και ξέρετε ότι οι ευρωσκεπτικιστές μόνο το αρνητικό κοιτάνε, δεν κοιτάνε πότε το θετικό. Στην Ευρώπη λοιπόν και φέτος ακόμη είχαμε 4,8% ποστό προσφάλματος, το οποίο όμως μας κάνει να ξεχνάμε ότι το 95% είναι πληρωμές, δαπάνες που έχουν χορηγηθεί σωστά. Εάν λοιπόν μιλάμε μόνο για το κακό, ξεχνάμε να μιλάμε για τα καλά της Ευρώπης. Yeah. Σας ευχαριστώ πολύ. Έχετε και άλλη ερώτηση να κάνετε κυρία Γκρέσλε. Το ερώτημα... Το ερώτημα για το μισογεμάτο και μισό άδειο ποτήρι, εγώ ξέρετε το απαντώ σε εξής, ότι αν είναι μισοάδιο το ποτήρι είναι πιο μεγάλο από ό,τι θα έπρεπε για το peer review. Λέτε ότι δεν χρειάζεται να γίνει συνενετική διαδικασία με τον ενεχόμενο. Είναι μια δύσκολη διαδικασία. Ο δημοσιονομικός κανονισμός το αναφέρει ότι υπάρχει αυτή κατά την παραβολή διαδικασία, όπως προβλέπετε, πολύ ωραία. Αλλά έχουμε την εντύπωση παρόλα αυτά ότι υπάρχει παρόλα αυτά η προσπάθεια για την διαφύλαξη αυτής της συνένεσης. Είναι αυτή η εντύπωση την οποία έχουμε αποκομίσει όλοι όσοι παρακολουθούμε τη δουλειά του ελεκτικού συνεδρίου. Γι' αυτό λοιπόν ε, δεν υπήρξε ζήτημα κριτικής θεώρησης από αυτή την πλευρά, αμφισβήτηση της κριτικής θεώρησης, αλλά ερωτώ ο ρόλος σας σε, αυτήν σε αυτές τις σχέσεις του peer review, πώς τον βλέπετε τον, ρόλο σας. Ευχαριστώ πολύ. Μήπως θέλει και η συγγήτρια ακόμη. Να σας διαβεβαιώσω ότι εμείς ως ελεκτικό συνέδριο ε, ακολουθούμε κατά τη εργασία μας αυστηρά τα, τα διεθνή πρότυπα δηλώσεις της ε, τη της Λίμας ε, της, ε, και τα λοιπά. Αλλά έχουμε και να οικοδόμημα το οποίο δεν ε, μπορεί να συγκριθεί με κανένα άλλο γενικότερα. Να σας διαβεβαιώσω λοιπόν ότι δεν ε, είμαστε ε, ούτε επικοί σε καμία περίπτωση με αυτά που, που ελέγχονται. μιλήσατε για συμφωνίες κτλ. δεν συμφωνώ. Σε ό,τι αφορά το κομμάτι αυτό, το τμήμα αυτό του peer review, εγώ προσωπικά δεν συμφωνώ. Γιατί δεν έχω ζήσει τέτοια πράγματα. Δεν συνάδει με την εμπειρία μου αυτό. Εντάξει, μπορεί η διαδικασία κατά την παραβολή να είναι λίγο πιο μικρή. Για να μην υπάρχει μια προπαρασκευαστική και μια πιο οριστική απόφαση και να μην υπάρχει και follow-up μετά. Αυτό μπορούμε όντω να το συντομεύσουμε ω διάστημα. Δεν νομίζω ότι θα αντιμετώπιζα κάποιο πρόβλημα σε ό,τι αφορά αυτή την πρόταση, αλλά ο κίνδυνο είναι ο εξή. Εκ των υστέρων, σε εθνικό επίπεδο και στο Κοινοβούλιο, θα τεθούν επερωτήματα, θα προκληθούν παρανοήσεις οι οποίες δεν θα έχουν διευκρινιστεί και θα ανακύψουν σε αυτή τη φάση. Αλλά αυτό επαφίεται στο Κοινοβούλιο να το αποφασίσει. Εγώ επαναλαμβάνω ότι δεν έχω πρόβλημα σε ό,τι αφορά την συντόμευση της διαδικασίας κατά την παραβολή, να αλλάξει η διαδικασία αυτή. Αλλά η υπόδειξη στο peer review ότι πηγαίνουμε παραπέρα από ό,τι θα έπρεπε να πηγαίνουμε δεν με βρίσκει σύμφωνο. Η κυρία Γκρέσλα και πάλι. Ναι, συγγνώμη, αλλά Μία μικρή ερώτηση, επιτρέψτε μου ακόμα. Στο έγγραφο αναφέρεται ότι χρειάζεται δύο χρόνια, παίρνει η προκαταρκτική έρευνα. Οι διαδικασίες αυτές είναι μυθικές σε ό,τι αφορά τη διάρκεια τους. Τι κάνετε λοιπόν εσείς, αν μου επιτρέπετε, ε, να σας ρωτήσω για να αλλάξετε αυτές τις διαδικασίες, γιατί όλα τα κράτη-μέλη παραπονιούνται γι' αυτό. Αλλά εγώ θα ήθελα να προωθήσουμε μια αλλαγή επιτέλους. Ρωτώ επίσης, σε μια έκθεση για τη χορηγήση αεροπαλλαγή, ζητήσαμε το χρονοδιάγραμμα για την ε, διαδικασία των ειδικών εκθέσεων να τηρείται το χρονοδιάγραμμα προκειμένου και να καταγράφετε για να δούμε πόσο διαρκούν αυτές οι διαδικασίες. Αν θέλετε λοιπόν να το κάνετε κι εσείς αυτό, ο κύριος Γκρέτεν. Κοιτάξτε. Εγώ μπορώ να σας υποσχεθώ, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο θα τηρήσω τις υποσχέσεις μου. Ξέρετε, είμαστε ένα σώμα 27 μελών η ε, κυρία Αγιάλα Σέντερ υπέδειξε ότι έχω αναλάβει τη σύνταξη πολλών ειδικών εκθέσεων συγκριτικά. Και από πλευράς αριθμού αλλά και από πλευράς δυσκολίας των εκθέσεων. Αυτό φυσικά επηρεάζει και το, την τήρηση του χρονοδιαγράμματος. Ο κανόνας λέει ότι καμία έκθεση, ειδική έκθεση δεν μπορεί να διαρκέσει πάνω από 18 μήνες από τη στιγμή της έναρξης των εργασίων μέχρι τη δημοσίευση της έκθεσης. Αλλά φαντάζομαι ότι και σε αυτό το επίπεδο ενδεχομένως να μπορούν να γίνουν συντομεύσεις. Βλέποντας για παράδειγμα ότι ο ελεγχόμενος έχει δύο μήνες στη διάθεσή του για να τοποθετηθεί, διαπιστώνοντας δε ότι υπάρχουν και μήνες οι οποίοι εξαιρούνται, όπως για παράδειγμα Αύγουστος εκ των πραγμάτων ή τα τέλη του έτους και τα, οι αρχές του έτους. Άρα γνωρίζουμε ότι υπάρχουν αυτές οι καθυστερήσεις. Θα μπορούσαμε, φαντάζομαι, να πούμε ότι, κοιτάξτε, ξέρετε τι ελέγχθηκε, ε, ήσασταν κι εσείς παρόν στον έλεγχο, έχετε 14 ημέρες να ανταποκριθείτε. Εγώ δεν θα είχα πρόβλημα με μια τέτοια πρόταση, αλλά τα άλλα θεσμικά όργανα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για παράδειγμα, θα είχε πρόβλημα θεωρώ. Εγώ προσωπικά δεν θα είχα πρόβλημα. Εμείς ως ηλεκτρικό συνέδριο, το είπα και αυτό εισαγωγικά, ίσως με κάποια σάφια, αλλά εργαζόμαστε στην παρούσα φάση προκειμένου να κάνουμε μία απόπειρα τουλάχιστον να δημοσιεύουμε τις εκθέσεις μας σε πιο σύντομο χρονικό διάστημα και να τις ε, ε, καταρτίζουμε στο μέλλον. Και αυτό είναι η προσωπική μου πεποίθηση. Θα πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη και να εξετάζουμε ε, πιο πολύ τα συμφέροντα και τι επιθυμίε των stakeholders και του Κοινοβουλίου δηλαδή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ λέει ο Πρόεδρος και νομίζω ότι στο σημείο αυτό μπορούμε να ολοκληρώσουμε την ε, ακρόαση. Κύριε Γκρέτεν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ. Και αν μου επιτρέπετε να προσθέσω μία κουβέντα, λέει ο κύριο ε, Γκρέτεν. Ε, κάτι πρόσθετο, εάν παρά, παρελπίδα δεν λάβω τη θετική γνωμοδότηση της Επιτροπής σας και του Κοινοβουλίου, είναι αυτονόητο ότι θα αποσύρω την υποψηφιότητά μου. Θέλω να είναι απόλυτα σαφές αυτό. Γιατί αυτό θα ήταν η απόδειξη ότι η δουλειά που έχω κάνει 7-6 χρόνια δεν ήταν τόσο καλή και ότι δεν έχω την εμπιστοσύνη του Κοινοβουλίου, η οποία είναι όρος εκτερών ουκάνευ για μένα. Και πρέπει να πω ότι εγώ έχω γράψει τον νόμο που ισχύει για το ελεκτικό συνέδριο του Λουξεμβούργου, μέσα στον οποίο ορίζεται ότι τα μέλη του ελεκτικού συνεδρίου ορίζονται από το Εθνικό Κοινοβούλιο και μόνο από αυτό. Δεν θα μπορούσα να κάνω κάτι διαφορετικό δηλαδή. Και καλώς ορίζω τον κύριο Ρίμπιχ που βλέπω εδώ με, με χειροκροτήματα όπως βλέπετε. Καλώς ήρθατε. Και μπορούμε να προχωρήσουμε χωρίς διακοπή στην ακρόαση του υποψηφίου που έχει προτείνει η κυβέρνηση των κατοχώρες για το ελεγκτικό συνέδριο τον κύριο Μπρένιγκ Μάιερ. Μπορείτε να κάνετε την ε, αρχική σας τοποθέτηση, αλλά παρακαλώ με μια κάποια συντομία. Okay. Yeah, yeah. <clears throat> Αγαπητέ Πρόεδρε, αγαπητά μέλη τη Επιτροπή Ελέγχου ε, των Προπολογισμών, θα ήθελα να σα ευχαριστήσω για την ευκαιρία αυτή που μου δίνετε για να παρουσιάσω την υποψηφιότητά μου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ιδιαίτερω στα εξέχοντα μέλη τη Επιτροπή ε, Ελέγχου Προπολογισμού θα παρουσιάσω ε, το βιογραφικό μου στα αγγλικά, θα απαντήσω τις ερωτήσεις στα αγγλικά, εάν χρειαστεί θα απαντήσω στα ολλανδικά σε περίπτωση που χρειαστεί μεγαλύτερη σαφήνεια. Εισαγωγικά λοιπόν θα ήθελα να σας παρουσιάσω κάποιες από τις απόψεις μου σε ό,τι αφορά τον ρόλο του Ευρωπαϊκού Ελεκτικού Συνεδρίου και θα ήθελα να σας παρουσιάσω και τους λόγους για τους οποίους ε, έχω μπει υποψήφιο σε τη θέση αυτή. Η σχέση μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του ολλανδικού Συνοδρίου και των μελών του θεωρώ ότι είναι πάρα πάρα πολύ σημαντική. Η έκθεση δραστηριοτήτων του Ελεκτικού Συνεδρίου θεωρώ ότι μπορεί να βελτιώσει τον δημοκρατικό ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε ό,τι αφορά τον έλεγχο, την άσκηση ελέγχου επί της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αν διοριστώ ως νέο μέλος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, θα δεσμευθώ προκειμένου να προσδώσω νέο νόημα στη συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα άλλα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Και είμαι συνηθισμένος σε διάλογο και επικοινωνία με το Κοινοβούλιο. Είναι σημαντική η σχέση με τα εθνικά ιδρύματα. Και αυτή η διάσταση είναι πολύ σημαντική. Κύριε Πρόεδρε, η ετήσια έκθεση για το 2012 που δημοσιεύτηκε την προηγούμενη Τρίτη στις, ε, περιλαμβάνει 19 αρνητικές δηλώσεις διαβεβαίωσης ε, στην μακριά λυσίδα ε, απογοητευτικών αποτελεσμάτων. Αυτά τα 19 λοιπόν αρνητικά μηνύματα μπορεί να σας φαίνονται κάτι συνθισμένο. αλλά εμένα δεν μου φαίνεται συνθισμένο. Αν ένας πολίτης μου ζητούσε να εξηγήσω πώς είναι δυνατόν να έχουν α, εκδοθεί τέτοια 19 αρνητικά α, μηνύματα, α, εκθέσεις ε, διαβεβαίωσης, ε, που δεν έχουν ωστόσο οδηγήσει σε απαλλαγή τη ε, Επιτροπή. Εγώ θα είχα πολλέ ιστορίε να πω. Αλλά θα έβλεπα ένα, αν θέλετε, μία αμφιβολία στα μάτια του πολίτη. Μπορώ να εξηγήσω με αξιόπιστο τρόπο το γεγονός ότι η νομιμότητα ε, ενός σημαντικού τμήματος ε, των ευρωπαϊκών δαπανών αμφισβητείται και ε, υπάρχει υποψία μην τήρησης των κανόνων για, την, για ανάθεση, για την εκχώρηση των κοντιλίων αυτών. Δεν θα είχε απαντηθεί με σωστό τρόπο και πιστικό τρόπο αυτό το ερώτημα. Η απόδοση ευθυνών στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να υποστηρίζει την νομιμότητα, υποστηρίζοντας την διαφάνεια του προπολογισμού. Πρόκειται για βασικές αρχές οποιασδήποτε δημοκρατίας. Και αυτό με οδηγεί σε μια σημαντική παρατήρηση για την εμπιστοσύνη των πολιτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην περιπλοκότητα της νομοθεσίας. Να ξεκινήσω από τα θέματα εμπιστοσύνης. Ως Ευρωπαίος διομεσο... Εθνικός στην Ολλανδία εργάζομαι... εργάστηκα πολύ σε θέματα που άπτονται της εμπιστοσύνης του πολίτη στη διακυβέρνηση και Είμαι πεπισμένο ότι οι εμπειρίε μου σε εθνικό επίπεδο μπορούν να ωφελήσουν το ευρωπαϊκό επίπεδο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό οι πολίτε να έχουν εμπιστοσύνη στι δημόσιε δαπάνε, στην δημόσια, δημοσιονομική διαχείριση και ότι τα συστήματα απόδοση ευθυνών θα πρέπει να λειτουργούν με αξιόπιστο και αποτελεσματικό τρόπο. Δυστυχώ όμω, στην ετήσια έκθεση τη, το ελεκτικό συνέδριο εξαγάγεται το συμπέρασμα ότι τα συστήματα αυτά εν μέρη μόνο είναι αποτελεσματικά. Θα πρέπει λοιπόν να βελτιωθεί και να ενδυναμωθεί η εμπιστοσύνη των πολιτών στα θεσμικά αυτά όργανα που χειρίζονται τους πόρους του Ευρωπαϊκού. Δεύτερο θέμα, σε ό,τι αφορά την πολυπλοκότητα, μία κορυφαία προτεραιότητα θα πρέπει να είναι να μειωθεί η περιττή περιπλοκότητα της νομοθεσίας και σε ό,τι αφορά την νομοθεσία και σε ό,τι αφορά την δημόσια διοίκηση. Αυτό επιβαρύνει την κοινωνία περιτά. Και γι' αυτό λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσπαθεί να περιορίσει τη γραφειοκρατία. Η ποιότητα των νόμων είναι πάρα πολύ σημαντική γιατί ζούμε σε μια δημοκρατία υπό το κράτο δικαίου και ω εκ τούτου είναι υπό τη ουσία και αξία η νομιμότητα για κάθε χώρα και θεωρώ λοιπόν ότι ένα βασικό καθήκον του Ρεκτικού Συνεδρίου είναι να εντοπίζει του κινδύνους που προκαλούνται από την περιπλοκότητα των πολιτικών και των νόμων. Αυτοί οι κίνδυνοι θεωρώ ότι θα πρέπει να τοποθετηθούν στην κορυφή των προτεραιοτήτων, όχι μόνο για να βελτιώσουμε τη διαφάνεια, αλλά για να περιοριστεί και ο κίνδυνος σφαλμάτων και απάτης. Είμαι πεπισμένο ότι οι ευρωπαϊκές πολιτικές θα πρέπει να είναι διαφανείς και κατανοητές για τους πολίτες στις σύγχρονες κοινωνίες, όπως όμως αυτό δεν είναι δεδομένο. Θα πρέπει λοιπόν αυτή η εμπιστοσύνη να οδηγήσει και σε εμπιστοσύνη στο σύστημα δημόσιας διοίκησης σε ευρωπαϊκό επίπεδο και άρα το νομικό πλαίσιο για τις, ε, τα κονδύλια θα πρέπει να είναι αποτελεσματικό και διαφανές. Θα πρέπει να υπάρχει λοιπόν τέτοια αποδοσή ευθυνών από τις εθνικές κυβερνήσεις, από τα εθνικά Ινστιτούτα από τις Εθνικές Υπηρεσίες Ελέγχου και λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ελεκτικό Συνέδριο μπορεί να βελτιώσει την εμπιστοσύνη των πολιτών και να βελτιώσει το κύρος των θεσμικών οργάνων. Κλείνοντας λοιπόν, ε, προσωπικό μου κίνητρο για την υποβολή της υποψηφιότητάς μου είναι η παρατήρηση ότι η καλύτερη απόδοση ευθυνών θα βοηθήσει, ελπίζουμε, τους πολίτες να πιστέψουν στον ευρωπαϊκό Προπολογισμό και ότι θα πρέπει να γίνουν πιο πολλά για να βελτιωθεί η ποιότητα της νομοθεσίας. Και η υποψηφιότητά μου προκαλείται σε μεγάλο βαθμό από την ε, ειλικρινή μου πεποίθηση ότι χρειαζόμαστε θεσμικά όργανα όπως το Λεκτικό Συνέδριο προκειμένου να υπάρχει ανεξάρτητη ε, εξωτερική ανάλυση και έρευνα που θα έχει τελικά θετική επίδραση στην εμπιστοσύνη από πλευρά των πολιτών αγαπητοί βουλευτές, αγαπητά μέλη της Επιτροπής Ελέγχου του Προπολογισμού. Ανυπομονώ και προσβλέπω στην καλή συνεργασία μαζί σας και θα χαρώ να απαντήσω στις ερωτήσεις σας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε κύριε Μπρένιγκ Μάιερ. Έχουμε τώρα λίγο χρόνο για ερωτήσεις. Πρώτα θα δώσω το λόγο στην εισηγήτριά μας, την κυρία Γιάλα Σέντερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και καλώς ήρθατε κύριε Μπρένιγκ Μάιερ. Είστε... ο υποψήφιος των κάτω χωρών για το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο. Καλώς ήρθατε και πάλι κύριε Μπρένιγκ Μάιερ. Είστε υποψήφιος των κάτω χωρών για το Ευρωπαϊκό Ελεκτικό Συνέδριο. Θα ήθελα να σας ομολογήσω ότι έχω κάποιες απορίες. Βλέπω ότι ως Ολλανδός διαμεσολαβητής ε, ήσταν υποψήφιος ε, το 2011 στις βουλευτικές εκλογές για, για ανανέωση της θητεία θητείας σας. Ανανεώθηκε η θητεία σας. Φαντάζομαι ότι κατεβήκατε στις εκλογές γιατί υπολογίζετε ότι θα μένατε έξι χρόνια στη Βουλή. Βλέπω ότι καταθέσετε υποψηφιότητα και για Ευρωπαίο διαμεσολαβητής. Και μάλιστα Ήσασταν και πρόεδρος ομόφωνα το 2012 του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Διεθνούς Συστήτου Διαμεσολάβησης. Δεν ξέρω ε, πόσα χρόνια θητεία έχετε εκεί. Και η κυβέρνησή σας σας όρισε υποψήφιο για τη θέση του ελεγκτή στο Ευρωπαϊκό Ελεκτικό Συνέδριο. Μήπως θα πρέπει κάποια στιγμή να επιλέξετε γιατί σας ενδιαφέρει το θέμα της εμπιστοσύνης των πολιτών. Βλέπουμε να, υποβάλ, να κατεβαίνει κάποιες εκλογές ε, ε, και ταυτόχρονα μην μπορεί να ολοκληρώσει την ε, θητεία του, ενώ ταυτόχρονα υποβάλλει και άλλου υποψηφιότητες. Βέβαια, ως ελεγκτής θα πρέπει να είστε εμπειρογνώμονας σε θέματα ελέγχου λογαριασμών. Έχετε και εμπειρία ως διαμεσολαβητής. Οπότε, μια ναι, και πρόκειται για δεύτερη υποψηφιότητα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, σε πολύ σημαντικό αξίωμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πώς βλέπετε αυτή την εναλλαγή των υποψηφιότητων. Επίσης, όταν μας μιλήσατε για τις τρεις πιο σημαντικές στιγμές της σταδιοδρομίας σας, είδα ότι ήσταν και δικαστής ε, στο τμήμα φορολογικών υποθέσεων ε, και σε ε, υποθέσεις ε, ισότητας ανδρών γυναικών. Και μάλιστα ο, οι πολιτικοί μερικές φορές ε, αμφισβήτησαν το θέμα της ανεξαρτησίας του δικαστού σε θέματα ισότητας φύλων. Γιατί πιστεύετε, γιατί αυτό μας είπατε, γιατί είπατε ότι οι πολιτικοί φοβούνται κατά κάποιο τρόπο μια τέτοια ανεξαρτησία ή έχουν επιφυλάξει με τέτοια ανεξαρτησία και πώς πιστεύετε ότι εσείς θα την ε, εξασφαλίσετε. Επίσης, ό,τι αφορά ε, τον δεσμευτικό χαρακτήρα του συστήματος ε, κυρώσεων ή αποζημιώσεων σε περίπτωση ανικανότητας για εργασία και σε διενέξει με την κοινωνική ασφάλιση. Είχατε πει ότι η κοινωνική ασφάλιση, το κράτος πρόνοιας έχει κλείσει στις κάτω χώρες. για αυτή ήταν η θέση της κυβέρνησης. Ποια είναι η γνώμη σας σχετικά για το θέμα των δημοσίων υπηρεσιών, το θέμα των δικαιωμάτων του πολίτη σε μια δημόσια υπηρεσία, κοινοφελή υπηρεσία υγείας είναι για μας πολύ σημαντικά θέματα. Αυτά προς το παρόν. Ευχαριστώ πολύ. Ας ακούσουμε όλες τις ερωτήσεις πρώτα. Και έτσι θα δώσω το λόγο στον κύριο Οντί και μετά στον κύριο Κερμπράντη. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Εκ μέρου του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματο, αλλά και προσωπικώ, θα ήθελα να σα καλωσορίσω καταρχά, να σα ευχαριστήσω για τι ευκρινήσει που μα προσφέρατε και να διατυπώσω δύο ερωτήσει. δεν έχετε, από ό,τι βλέπω, κατάρτιση στον δημοσιονομικό έλεγχο ή εμπειρία σχετική. Στο σημείο αυτό της εμπειρίας του δημοσιονομικού έλεγχου μπορείτε να μας ε, διευκρινίσετε ποια στοιχεία θα μας οδηγούσαν στη διαπίστωση ότι θα είστε καλός ως μέλος, κατάλληλος ως μέλος γιατί σας ήταν βέβαια καλός δημοσιολαβητής, αλλά ο δημοσιολαβητής δεν απαραίτητα καλός δημοσιονομικός ελεγκτής. Για το, για το ζήτημα της ανεξαρτησίας μπορείτε να μας προσφέρετε ανε, ε, εγγυήσεις ως προς την ανεξαρτησία σας έναντι της Ολλανδικής κυβέρνησης που σας έχει προτείνει. Μπορείτε να μας καθισχάσετε σχέση με αυτό. Αυτές είναι οι δύο μου ερωτήσεις, Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Γκερμπράντι έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και εγώ θα ήθελα να καλωσορίσω τον κύριο Μπρένιγκ Μέιρ στην Επιτροπή Ελέγχου Προϋπολογισμών. Να κάνω και εγώ κάποιες ερωτήσεις. Συμφωνώ με τον κύριο Ντι. Έχω μία παρατήρηση να κάνω για την ανεξαρτησία. Η ανεξαρτησία είναι αναπόσπαστο μέρος ενός μέλους του ελεκτικού συνεδρίου, αλλά ασφαλώς και ε, ουσιώδους σημασίας για την επιτέλεση των καθοκόντων του διαμεσολαβητή. Αν μπορώ λοιπόν κάτι να επιβεβαίωσω από πλευράς Ολλανδίας είναι ότι όντως ε, ε, είχατε μια ανεξάρτητη θέση ως διαμεσολαβητής και γι' αυτό λοιπόν στη Χάγη να μην τους πειράσει τόσο πολύ που θα φύγετε να πάτε στι Βρυξέλλε. Αυτό είναι όμως προσωπική μου εκτίμηση. Δύο άλλες ερωτήσει έχω να θέσω. Μιλήσατε εκτενώς στην ε, εισαγωγή σας για το γεγονός ότι οι πολίτες θα πρέπει να έχουν καλύτερη επισκόπηση σε ό,τι αφορά θέματα ευρωπαϊκού προϋπολογισμού, προκειμένου να υποστηρίζεται αυτή αυτός πιο ευραίος από τους πολίτες στο λεκτικό συνέδριο στο Λουξεμβούργο απέχεται πολύ από τον πολίτη και διαβάζοντας τις εκθέσεις του λεκτικού συνεδρίου ακόμα και οι πιο ειδικοί, οι πιο μεγάλοι εμπειρογνώμονες δυσκολεύονται να κατανοήσουν ακριβώς το περιεχόμενο των εκθέσεων. Άρα, ποιες ιδέες έχετε συγκεκριμένα για να προσελκύσετε τον πολίτη. Και το δεύτερο θέμα είναι λίγο πιο ευρύως πρόβλημα είναι κάτι το οποίο εδώ και χρόνια επισημαίνω και υπογραμμίζω. Η αποτελεσματικότητα των ευρωπαϊκών ε, κονδυλίων, των ευρωπαϊκών δαπανών που έχει βάζει πολύ νερό. Αν λοιπόν υπάρχει ένα θεσμικό όργανο που μπορεί να προασπίσει αυτά, είναι το ελεκτικό συνέδριο και σε ό,τι αφορά ε, την περιπλοκότητα του θέματος και σε ό,τι αφορά τις εκθέσεις. κοιτώντα λοιπόν την έκθεση για το 2012, την ετήσια έκθεση, περιλαμβάνονται όλα τα σχέδια για την επόμενη επταετή δημοσιονομική περίοδο. Είναι καταστροφική. Πώς θα καταφέρουμε και το χρησιμοποιώ το πρώτο πληθυντικό ε, συνειδητά. Πώς θα τα καταφέρουμε μαζί με το ελεκτικό συνέδριο σε ό,τι αφορά τις εκθέσεις αυτές του ελεκτικού συνεδρίου να μεταφραστούν τα συμπεράσματα των εκθέσεων σε συγκεκριμένες πράξεις. Γιατί κάθε χρόνο μιλάμε για την περιπλοκότητα που είναι πάρα πολύ ψηλή ε, και ότι δεν πετυχαίνουμε τελικά τα αποτελέσματα. Ένα τελευταίο σχόλιο. Αυτό που μου προξενεί πάντα εντύπωση σε ό,τι αφορά το ελεκτικό συνέδριο είναι ότι δεν ε, πρόκειται για τα μεμονωμένα κρατέν μέλη. Θα μπορούσατε λοιπόν να ε, τοποθετηθείτε σε ό,τι αφορά την... το να κατανομωστουν συγκεκριμενα συγκεκριμένα κράτη-μέλη που έχουν προβλήματα. Ευχαριστώ κύριε Κρυπράντη. Ο επόμενος είναι ο κύριος Ρουμπίκ. Ευχαριστώ πολύ πρόεδρε. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω το μέλλον εφόσον λάβετε καθήκοντα στο ελεκτικό συνέδριο. Πώς βλέπετε την κατάσταση των ε, πληρωμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και τους φορολογικούς παραδείσους. Πώς είναι δυνατόν να συμμετέχουν φορολογικοί παράδεισοι σε project και σχέδια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομίζετε ότι αυτό μπορεί να αποτελέσει έργο του ελεκτικού συνεδρίου. Ευχαριστώ πολύ και για να ολοκληρώσουμε το κομμάτι αυτό, κύριος Χάρτονγκ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, αξιότιμε συνάδελφοι. Θεωρώ ότι ένα μέλο του Ελεκτικού Συνεδρίου θα πρέπει να είναι απόλυτα ανεξάρτητο, γιατί θα πρέπει να μην έχει ε, πολιτικό χρώμα και να ασκεί τα καθήκοντά του με αξιοπρεπή τρόπο. Και μου φαίνεται ότι δεν είναι τόσο ανεξάρτητο ο κ. Μπίνκεν Μάιερ. Ε, Όπω φάνηκε ε, στις 20 Οκτωβρίου στο τηλεόραση έκανε την εξή δήλωση. Ε, η πολιτική καιρή εδώ στην Ολλανδία είναι διακριτική, ρατσιστική και δεν μιλάω για ένα πολιτικό κόμμα αλλά για τη γενικότερη πολιτική ε, κουλτούρα στην Χάγη που είναι κατά του εξωτερικού ε, λαϊκισμός, εθνικισμός, πολύ εθνικιστική, πολύ λαϊκιστική είναι η Ολλανδία. Τέλος παράθεσης. Αυτά δήλωσε ο κύριος Μπρινιγκ Μάιερ. Αν λοιπόν τόσο έντονα είναι τα συστήματα του κ. Μπριγμαϊρ για την ε, πολιτική κατάσταση, αναρωτιέμαι κατά πόσον μπορεί να είναι μέλο υποψήφιο από πλευρά τη χώρα μου για το ελεκτικό συνέδριο. Ε, εκφράζει, περιφρονή περιφρονεί τους, ε, το πολιτικό σύστημα και την κουλτούρα στη χώρα μας. Και επίσης δεν ξέρω κατά πόσο τα κίνητρά του είναι αμυγή. Ήταν υποψήφιος προσφάτως για για τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή. Αλλά τώρα παρουσιάζεται εδώ ως υποψήφιος για το ελεγκτικό συνέδριο. Μου φαίνεται ότι μάλλον αναζητά μία θέση και δεν επιθυμεί πραγματικά να εξυπηρετήσει τα συμφέροντα του ευρωπαϊκού πολίτη. Ερωτώ λοιπόν είναι διτεθειμένος χωρίς ε, καμία επιφύλαξη να ζητήσει συγγνώμη και να αποσύρει τη δήλωσή του αυτή που περιφρονεί το Ολλανδικό κράτος. Αν όχι, θα συστήσω και στην εισηγήτρια και στους αξιότιμους συναδέλφους να αποφανθούν αρνητικά για την υποψηφιότητά του. Äh, ευχαριστώ πολύ <clears throat> για την ομοβροντή αυτή ερωτήσεων. Έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε για την ευκαιρία που μου δίνετε να απαντήσω σε όλες ε, αυτές τις εξαιρετικά ενδιαφέρουσες ε, ερωτήσεις και να σας διαφωτίσω για διάφορα θέματα. Η κυρία Σέντερ με ρώτησε τι θα προσφέρω εγώ με τη δική μου πείρα και διαδρομία στο Ευρωπαϊκό Ελεκτικό Συνέδριο. Πώς θα συνεισφέρω. Όντως, ε, δεν έχω πείρα δημοσιονομικού ελεγκτή ούτε στις κατοχώρες ούτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά δεν είναι όλα τα μέλη του ελεγκτικού συνεδρίου που έχουν πείρα δημοσιονομικού ελεγκτή, ούτως ή άλλως. Πάντως, ε, έχω διαδρομία και ως πανεπιστημιακός και ως δικαστής και ως διαμεσολαβητής. Και, όπως βλέπετε, ε, είχα ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα θέματα, το, θέμα των δημοσίων ε, λογαριασμών και ως δικαστής ασχολήθηκα ιδιαίτερα με φορολογικά ζητήματα, με κοινωνικά επιδόματα, συντάξεις και ως ε, πανεπιστημιακός καθηγητής ε, έκανα δημοσιεύσεις ε, για την εισαγωγή του ευρώ, για την Ευρωπαϊκή Νομισματική Ένωση και ανέλησα τις συνέπειες αυτής της νομισματικής ένωσης στην Ευρωπαϊκή Δημοκρατία. Και εγώ δεν ταυτίζομαι με την ιδιότητα του δημοσιονομικού ελεγκτή, αλλά ε, ασχολήθηκα πιο γενικά ε, με πολλά θέματα και ως δικαστής και ως ε, καθηγητής, ως πανεπιστημιακός. Και πολύ σύντομα εξοικειώθηκα με πολύ ε, πολύ γρήγορα εξοικειώθηκα με πολύ περίπλοκα θέματα και έχω προετοιμαστεί για την πιθανότητα ε, συμμετοχή στο Ευρωπαϊκό Ελεκτικό Συνέδριο. Όταν ο Ολλανδό Υπουργό Οικονομικών με ρώτησε αν ενδιαφέρομαι να είμαι υποψήφιο στον κάτω χωρό στο Ελεκτικό Συνέδριο, ανακάλυψα ότι αφενός ε, απαιτείται ένα πολύ βαθύ τεχνικέ γνώσει για τη μεθοδολογία τη δήλωση αξιοπιστία τη ΔΑΣ Απ' την άλλη όμως βλέπουμε ότι ο ρόλος του ελεκτικού συνεδρίου είναι και από άλλες απόψεις ε, σημαντικός και αποτελεσματικός και θα πρέπει να εξοικειώσουμε και τους πολίτες με το ρόλο του δημοσιονομικού ελεγκτή. Γιατί μερικές φορές δεν καταφέρουμε να εξηγήσουμε στους πολίτες ότι η δήλωση του ελεκτικού συνεδρίου για πολλά χρόνια ήταν αρνητική. Τι θα πρέπει λοιπόν να κάνουμε γι' αυτό να προσθέσουμε άλλους 10 ελεκτές στο σύστημα, 50, 100, 200, 200 ή θα πρέπει να θέσουμε με διαφορετικό τρόπο τις ερωτήσεις, πιο εύστοχες ερωτήσεις, ερωτήσεις που ενδιαφέρουν και αγγίζουν περισσότερο τον Ευρωπαίο πολίτη. Εγώ σε αυτό το δεύτερο θα ήθελα να συμβάλλω. Κυρία Σέντερ, είπατε ότι ήμουν υποψήφιος και για τη θέση του Ευρωπαίου Μεσολαβητή και τώρα είμαι υποψήφιος ε, για το ελεκτικό συνέδριο, το Ευρωπαϊκό Ελεκτικό Συνέδριο. Ε, τι θέλετε, μήπω ε, ζητάτε μια καλή θέση. Απλώς, όχι κυρία Σέντερ, δεν ζητώ μια καλή θέση, ένα καλό θόκο. Εγώ ήμουν διαβεσολαβητής και στι κάτω και όταν ο Υπουργό Οικονομικών ε, της Ολλανδία με ρώτησε αν με ενδιαφέρει υποψηφιότητα στο ελεκτικό συνέδριο, πραγματικά έμεινα άναυδο. Εξεπλάγιν που ήρθε σε μένα τον πρώην Ολλανδό διαμεσολαβητή να μου ζητήσει να είμαι υποψήφιο για τη θέση του ελεκτικού συνεδρίου και το ρώτησε γιατί εγώ, γιατί με διαλέξατε. Και μου είπε, καταρχήν ήσασταν ικανός να μετατρέψετε την τελείως άγνωστη ιδιότητα του Ολλανδού διαμεσολαβητή σε ένα πολύ γνωστό θεσμό του συνηγόρου του πολίτη και πια οι Ολλανδοί έχουν μεγάλη εμπιστοσύνη στην εύρυθμη λειτουργία του Ολλανδού διαμεσολαβητή και του ρόλου του. Εγώ πιστεύω ότι και στο Ευρωπαϊκό Ελεκτικό Συνέδριο μπορώ να παίξω αυτό τον ρόλο. Να γεφυρώσω δηλαδή από τη μία την τεχνικό, τεχνικό χαρακτήρα και την περιπλοκότητα των, του ελέγχου των λογαριασμών με το ενδιαφέρον των Ευρωπαίων πολιτών. Και αν ρίξετε μια ματιά στο ανακοινοθέν τύπου ε, του ελεκτικού συνεδρίου, διαρωτάστε πόσοι Ευρωπαίοι πολίτε είναι ικανοί να το καταλάβουν, λιγότερο από 1%. Αλλά και δημοσιογράφου να ρωτήσουμε, καταλαβαίνετε την έκθεση του ελεκτικού συνεδρίου και πάλι ούτε 1% δεν την καταλαβαίνει, των δημοσιογράφων. Κανένα ουσιαστικά δεν καταλαβαίνει τι συμβαίνει. Και στα οικονομικά έχω μάθει ένα δύσκολο μάθημα, ότι κανεί, δεν θα πρέπει κανεί να βάζει την υπογραφή του σε ένα έγγραφο που δεν κατανοεί. Και αυτό είναι πολύ δύσκολο το πρόβλημα. Πώ θα εξηγήσουμε τη λογοδοσία στην Ευρώπη και στου πολίτε. Και αυτό θα ήθελα να κάνω εγώ. Αυτή είναι η δική μου επιθυμία. Πιστεύω ότι απαντώ έτσι και στην, στην ερώτηση του κυρίου Οντί που με ρώτησε τι θα προσθέσω εγώ στη λειτουργία τώρα. Κάτι που αφορά και τις παρατηρήσεις του κυρίου Χάρτονγκ σε ό,τι αφορά τη διακριτική μεταχείριση. Η συνεισφορά μου σε ό,τι αφορά την καταπολέμηση της διακριτικής μεταχείρισης και των διακρίσεων, όχι μόνο στην Ολλανδία, αλλά γενικά, ε, έχει εκτιμηθεί ιδιαίτερω. Γιατί πολλοί πολίτε ήρθαν και μου είπαν «Χαιρόμαστε ιδιαίτερω που θίξετε αυτό το ζήτημα των διακρίσεων». Κύριε Χάρτον, αυτό είναι απόδειξη της ανεξαρτησίας μου της ανεξαρτησίας μου από την ε, Ολλανδική κυβέρνηση και δεν θα αποσύρω την υποψηφιότητά μου επειδή εσείς έχετε διαφορετικές πολιτικές ιδέες. Τώρα έχετε δικαίωμα να πρεσβεύετε τις ιδέες σας. Κύριε ότι με ρωτήσατε αν είμαι ανεξάρτητος. Είμαι πλήρως ανεξάρτητος και είμαι γνωστός στην Ολλανδία για την ανεξαρτησία μου. Ήμουν ανεξάρτητος δικαστής, ανεξάρτητος και ως πανεπιστημιακός, ως ακαδημαϊκός και ως διαμεσολαβητής. Φαίνεται ότι έχω το γονίδιο της ανεξαρτησίας. Απ' την άλλη, με ενδιαφέρει η συνεργασία και σέβομαι τη συνεργασία με την Ολλανδική Βουλή και έχτισα γέφυρες με την Ολλανδική Βουλή. Ρώτησα τους βουλευτές τι πιστεύετε ότι είναι σημαντικό στο έργο του διαμεσολαβητή. Και νομίζω ότι είναι πολύ σημαντική αυτή η ερώτηση και πολύ εύστοχη Πώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τι θεωρεί η Επιτροπή Ελέγχου Περιπολογισμού ότι είναι σημαντικό στο μελλοντικό έργο του Ευρωπαϊκού Ελεκτικού ε, Συνεδρίου και πώ θα το καταστήσουμε πιο αποτελεσματικό και πιο πιστικό. Κύριε Γκερμπράντε. Τονίσατε την ε, σημασία της σχέσης μας με τους Ευρωπαίους πολίτες. Και αυτό το θέμα το ανέπτυξα και εγώ ενδελεχώς, ε, γιατί συμφωνώ μαζί σας. Είναι σημαντική σχέση με τους πολίτες. Η δεύτερη σας ερώτηση αναφέρθηκε στην αποτελεσματικότητα και στο κατά πόσο πιάνουν τόπο τα ευρωπαϊκά κονδύλια και πώς αξιοποιούνται. Αυτό το θέμα με ενδιαφέρει ιδιαίτερος. Στην τηλεόραση πολύ συχνά παρακολουθούμε εκπομπές για ευρωπαϊκά προγράμματα και σχέδια που δυστυχώς δεν εξυπηρέτησαν κανένα σκοπό, ήταν προβληματικά και γι' αυτό προκάλεσαν τον περίγελο. Ο δημοσιονομικός έλεγχος του Ευρωπαϊκού Ελεκτικού Συνεδρίου ασχολείται και με τα θέματα αυτά. Το πόσο αποτελεσματικά είναι τα ευρωπαϊκά προγράμματα. Και εκεί βρίσκεται και ο συνδετικός κρίκος ε, μεταξύ του δημοσιονομικού ελέγχου και της καθημερινότητας των Ευρωπαίων πολιτών. Αυτός ο συνδετικός κρίκος αυτή τη στιγμή είναι κάπως ασθενής. Θα πρέπει να τον ενισχύσουμε. Επίσης, το ίδιο το δημοσιονομικό πλαίσιο δεν είναι και πολύ σαφές. Το αιτιολογικό δεν είναι αρκετά σαφές. Γι' αυτό και ο ρόλος του ηλεκτρικού συνεδρίου θα πρέπει να επικεντρωθεί στο θέμα της αποτελεσματικότητας ε, των ε, ε, δαπανών του επόμενου δημοσιονομικού πλαισίου. Και ο δημοσιονομικός έλεγχος θα πρέπει να επικεντρωθεί σε αυτό, στην αποτελεσματικότητα και στη σωστή εκτέλεση του προπολογισμού. Το πλαίσιο το έχουμε. Θα πρέπει όμως να το εφαρμόσουμε και σωστά για να το εκτελέσουμε με καλό τρόπο. Και εκεί χρειαζόμαστε περισσότερη ακρίβεια, πιο ελέγξιμους και καταμετρήσιμους στόχους ε, της χρηματοδότησης. Τελευταία ερώτηση αφορούσε τους φορολογικούς παραδείσους. Πιστεύω ότι στην Ευρώπη το θέμα των πολιτικών παραδείσων είναι πολιτικό ζήτημα και δεν είναι θέμα του ελεκτικού συνεδρίου θα πρέπει να ξαναεξετάσουμε το θέμα της δίκης φορολόγησης. Εγώ είμαι υπέρ αυτής της αναθεώρησης. Ευχαριστώ, και πολύ. Έχουμε, έχω ακόμα συμπληρωματικές ερωτήσεις. Ο κύριος Χάρτονγκ. Όχι, πρόεδρε, δεν είναι ο κύριος Ωντί. Δεν είναι ερώτηση, είναι παρατήρηση. Ο υποψήφιος μας είπε πολλές φορές ότι 19 αρνητικές ε, δηλώσεις αξιοπιστίας έχουν εμφανιστεί και ότι όλα αυτά είναι και δυσνόητα. Έστω ε, δυσνόητα είναι, αλλά δυσνόητη είναι η διατύπωση του ελεκτικού συνεδρίου. Ενώ ο νόμος λέει ότι πρέπει να υπάρχει μία δήλωση αξιοπιστίας και στο κείμενο, ενώ η πιστοποίηση των λογαριασμών είναι θετική, έχει θετικά στοιχεία, είναι ε, τακτή και τυπική οι λογαριασμοί. Στα έσοδα είναι όλα εντάξει, στο, στις δαπάνες έχουμε μικρό σφάλματα 2-3% και τέλει μετά ακούμε δήλωση αξιοπιστίας αρνητική. Μα όταν τα ακούσει κανείς αυτό που δεν είναι δικό σου, πώς θα καταλάβει. Εχθές δεν μπόρεσαν να με πάρουν και στη συζήτηση και λυπούμε γι' αυτό. Ο κύριος Χάρτον έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Η απάντηση του κ. Μπρένιγκ Μάιερ ε, σημειώνεται ότι αρνείται να αποσύρει τις δηλώσεις του για λόγους σαφήνειας να πω ότι στις δηλώσεις του δεν κρίνατε μόνο το δικό μου κόμμα, το οποίο είναι και δικαίωμά σα, αλλά όλα τα πολιτικά κόμματα της Ολλανδίας και φαίνεται ότι σκέφτεστε ακόμα ε, ως διαμεσολαβητής και όχι ως υποψήφιος ε, για το ελεγκτικό συνέδριο. Και φαίνεται ότι Ξέρετε ότι αυτό το σύστημα είναι πολύ αμφιλεγόμενο και πολύ ακαθόδες στην Ολλανδία. Γι' αυτό λοιπόν ε, διατηρώ τι απεφυλάξει μου να απαντήσω στα Ολλανδικά. Φαντάζομαι ότι ε, εμένετε στην ε, θεώρησή σα αυτή και σα εύχομαι κάθε επιτυχία. Σα ευχαριστώ. Μπορούμε να ολοκληρώσουμε και αυτή την ακρόαση. Κύριε Μπρένινγκ, σα ευχαριστώ θερμά που ήρθατε στην ακρόασή μα. Μέχρι νεοτέρας λοιπόν σε άλλες διαδικασίες. Και έτσι μπορούμε να περάσουμε στον προσεχή υποψήφιο Ja, meine Damen και κύριοι, μετά τη σύντομη αυτή διακοπή, παρακαλώ να καλωσορίσουμε εδώ τον κύριο Owen, εδώ στην Επιτροπή μας. Ε, πρόκειται για τον επίσημο υποψήφιο από το Ηνωμένο Βασίλειο. Είσαστε υποψήφιος λοιπόν για το λεκτικό συνέδριο. Παρακαλώ να μας δώσετε τις εισαγωγικές σας παρατηρήσεις. Έχετε το λόγο κύριε Όουν. Κύριε Πρόεδρε, κύριε και κύριοι της Επιτροπής, σας ευχαριστώ πολύ. Είναι μεγάλη τιμή που βρίσκομαι εδώ. Οι γονεί μου είχαν πολύ αυστηρές αρχές και αξίες ως προς την ευθύνη μας των πολιτών και με ενθάρρυναν να γίνω κι εγώ υπεύθυνο πολίτης. Ε, ήμουν αρκετά χρόνια στο Διοικητικό Συμβούλιο Μεγάλων, ε, μεγάλων Δημόσιων Νοσοκομείων. Προσπαθώ να βελτιώσω τη διακυβέρνηση με μία ε, ουδετερότητα ταυτόχρονα. Το δε, η δεν απογραφία, αντίγραφο μάλλον θα ο μιλητής, του Ντονιτσέτη για την καλή διακυβέρνηση είναι κρεμασμένη σε ένα τοίχο του σπιτιού μου. Τα τελευταία εννέα χρόνια ασχολούμαι με μεταρρυθμίσεις υψηλού κινδύνου, μακροπρόθεσμες μεταρρυθμίσεις, μεταρρυθμίσεις σχετικές με τις συντάξεις, με την γύρανση του πληθυσμού, με την κλιματική αλλαγή, με την ενέργεια και έχω αναλάβει και εποπτεύσει πολλές ανεξάρτητες εκθέσεις ε, αντίστοιχες με αυτές απόδοσεις ή της ε, ε, γενικής εκθέσεως του ελεγκτικού συνεδρίου. Έχω εμπειρία από το δημοσιονομικό έλεγχο, έχω προσωπικώς ελεγχθεί πολλές φορές και έχω υπηρετήσει ως υπεύθυνος για τα λογιστικά και ως εκ έχω κληθεί ενώπιον της Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγχου στη χώρα μου. Έχω συμμετάσχει σε Επιτροπές Δημοσιονομικού Ελέγχου αυτή τη στιγμή στην ε, Εθνική υπηρεσία ελέγχου παγιώνω, εμπεδώνω τις ε, γνώσεις μου. Έχω εμπειρία από μεγάλους οργανισμούς με πάνω από χίλια, χίλια μέλη προσωπικό στο είναι, στην ελεκτική αρχή, αλλά και στους δημόσιους οργανισμούς που έχω εργαστεί νωρίτερα με πάνω από 100.000 ε, προσωπικό. Έχω ε, Μεγάλη πίστη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι βλέπω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και προσθεμένη αξία και εμ, ηγετικό ρόλο στα παγκόσμια πράγματα και αποφασιστικό ρόλο έχετε. Πρόκειται για την μεταρρύθμιση των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, την κλιματική αλλαγή, η άλλα ζητήματα στα οποία έχει συμβάλει και στη βελτίωση των, του, του, πλαισίου στον Ηνωμένο Βασίλειο η Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία τώρα περνάει μια ε, περίοδο αλλαγών, όπως κατέγραψε και ο εισηγητής σας στην έκθεση για το μελλοντικό ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ελπίζω ότι θα μπορέσω ως μέλος του Ελεκτικού Συνεδρίου να ανήκω σε ένα όργανο το οποίο θα κάνει τα εξή πράγματα καλύτερα, ότι θα συνεργάζεται καλύτερα και θα, θα χρησιμοποιεί καλύτερα το ελεκτικό έργο της Επιτροπής και των ανωτάτων ελεκτικών ε, θεσμών των κρατών μελών. Δεύτερον, θα μπορέσει να μετακυλήσει την, ε, την ισορροπία προς περισσότερη αξιολόγηση αποδοτικότητας με εντοπισμό υψηλού κινδύνου περιοχών και καλύτερων αποτελεσμάτων. Και έτσι γιατί και, το οι Ηνωμένε Πολιτείε αλλά και το Γαλλικό Ελεκτικό Συνέδριο έχουν αποδείξει ότι μπορούν πολλά πράγματα να γίνονται και καλύτερα και ταχύτερα. Τρίτον, ελπίζω ότι θα μπορέσει να είναι πολύ πιο υψηλή η επίδραση, η επιρροή του Ελεκτικού Συνεδρίου με ε, την ε, γνώση, τη λογοδοσία και τα προγράμματα διαχείρισης. Θα είναι τιμή για μένα το να υπηρετήσω στο ελεκτικό συνέδριο. Θα είμαι θεματοφύλακα των χρηματοπιστωτικών χρηματο των δημοσιονομικών συμφερόντων των, ε, ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα μεριμνώστε κάθε ε, ευρώ που δαπανάτε για την Ευρωπαϊκή Ένωση να αποδίδει. Και πιστεύω ότι θα μπορέσω και με καλή συνεργασία μαζί αλλά και με καλή διάθεση με την Ένωση, του εθνικού θεσμού, ιδιαίτερα όμω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Επιτροπή σα, να αναλάβω τα καθήκοντά μου. Σα ευχαριστώ πολύ. Είμαι έτοιμο να ακούσω τι ερωτήσει σα. Σας ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Η καλή διάθεση και το χιούμορ που όπως όλοι ξέρουμε δεν κοστίζει τίποτα αλλά βοηθάει πολύ στη βελτίωση της ζωής. είναι πολύ σημαντικό. Ας ακούσουμε πρώτα την εισηγήτρια, κυρία Γιάννα Σέντερ. Ευχαριστώ. Καλώς ήρθατε κύριε Όεν στην Επιτροπή Ελέγχου Προϋπολογισμού ως υποψήφιος της ε, Βρετανικής κυβέρνησης για το Ευρωπαϊκό Ελεκτικό Συνέδριο. Είναι πολύ σημαντικό που αναφέρετε τους γονείς σας ε, που σας ε, εστάλαξαν αυτά τα χαρακτηριστικά και βλέπω ότι είστε εδώ κάνατε ένα στάζι, μια, είχατε μια περίοδο άσκησης στο Βρετανικό Ελεκτικό Συνέδριο. Αυτό βλέπω στο βιογραφικό σας γιατί από την ε, υποψηφιότητά σας βλέπω ότι πήγατε ε, στο Εθνικό σας Ελεκτικό Συνέδριο και κάνετε ένα είδος μαθητείας άσκησης. Γιατί ε, επιδιώξατε αυτή την άσκηση σε ένα βρετανικό θεσμικό όργανο. Μπορείτε να μας το δικαιολογήσετε. Είναι πολύ σημαντική η εμπειρογνωμοσύνη σας ε, και η γνώση ε, για τα οικονομικά θέματα. Στην ερώτηση 4 είδατε ότι αποδίδουμε ιδιαίτερη σημασία στο θέμα της έγκρισης της ε, διαχείρισης, της δημοσιονομικής διαχείρισης και για ιστορικούς λόγους, αλλά και η σύγκριση με τους εθνικούς μηχανισμούς δεν είναι εύκολη. Είπατε ότι στην Βρετανική νομοθεσία δεν εφαρμόζεται ένα, ένα αντίστοιχο δεν γίνεται αντιστοίχη βεβαίωση ε, της δημοσιονομικής διαχείρισης, τότε πώς γίνεται η έγκριση της διαχείρισης, γιατί είπατε ότι ήσταν υπεύθυνο για διαχείριση πολύ μεγάλων ποσών. Είπατε ότι είστε εκτελεστικός διευθυντής του ομίλου της, ε, της Εθνικής Υπηρεσίας Υγείας. Θα ήθελα να μου πείτε ακριβώ ε, ποια είναι τα καθήκοντά σας εσύ και η Εθνική Υπηρεσία Υγείας, το NHS, ε, στο οποίο είστε αντιπρόεδρος με εκτελεστικός διευθυντής, έλαβε, ε, έχει λάβει κοινοτικά κονδύλια. Συμμετείχατε σε πολύ σημαντικά θέματα, όπως είναι η, η διάλυση ενός εργοστασίου αντιμετωπίσατε δυσκολίες σε κοινοβουλευτικό επίπεδο με τα θέματα αυτά γιατί υπήρχε με ένα πρόβλημα, δεν κάνω λάθος τότε, με τη Βουλή και πώς τις ξεπεράσατε. Ευχαριστώ. Κύριο Στόγων έχει Βον. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και κύριε Όν, καλώς ήρθατε στην Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Σας συγχαίρω για την παρουσία σας αυτό, όχι μόνο γιατί είστε ουαλός, όπως εγώ, αλλά φαντάζομαι ότι αυτό θα εξηγεί και την αίσθηση του χιούμορ που έχετε. Το ξέρουν οι συνάδελφοι ότι και εγώ έχω χιούμορ. Τρεις ερωτήσεις. Πρώτον, ανεξαρτησία. Έχουμε συζητήσει το θέμα αυτό με τους άλλους ε, υποψηφίους τη σημασία της ανεξαρτησίας των μελών αλλά και του ελεγκτικού συνεδρίου στο, στο βιογραφικό σας σημείωμα βλέπω ότι έχετε εργαστεί για δεξιάς κυβέρνηση υπουργού. Ε, και ίσως αυτό αποτελέσει λόγο ανησυχίας για την ανεξαρτησία σας. Μπορείτε να μας εξηγήσετε κάτι. Και κάτι ακόμη. Καθώς ήμουν επικεφαλής μιας ε, ε, δημοτικής αρχής, κοινοτικής αρχής καλύτερα, θα ήθελα να ρωτήσω ε, γιατί εγώ πιστεύω ότι η ανταλλαγή των βέλτιστων πρακτικών είναι κάτι το οποίο μπορεί να, στο οποίο θα πρέπει να επενδύσουμε, να διαδίδουμε λέει στους άλλους ότι καλύτερο έχουμε. Εσείς για το ελεκτικό συνέδριο αυτό πώς το βλέπετε. Και επίσης για το 2012 την έκθεση που δημοσιεύτηκε αυτή την εβδομάδα και που θα γνωρίζετε ότι το ποστό σφάλματος έχει αυξηθεί στα 4,8 από 3,9%. Προφανώς κακό δείγμα. Ξέρουμε ότι τα κράτη-μέλη θεωρούν και ισχυρίζονται ότι είναι σφαλμένη αυτή η ένδειξη σφάλματος. Ε, ωστόσο, ξέρουμε ότι ούτε πρόκειται να τα εξυπηρετήσει το να παραμείνει αυτό το σφάλμα. Τι είδου σχόλια θα μπορούσατε να κάνετε για, αυτούς, τους, για αυτή την κατάσταση. Ευχαριστώ κύριος Γκερμπράντη. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ και εσάς κύριε Όουεν για την αρχική σας δήλωση. Νομίζω ότι η υποψηφιότητά σας ήταν εξαιρετική Η μαθητεία σας ήταν ε, εξαιρετική ιδέα. Ελπίζω να το έχουν κάνει κι άλλοι αυτό. το είχε κάνει και η κυρία κάμερα πριν είχε εργαστεί στο Συμβούλιο. Σε ό,τι αφορά τους ελέγχους απόδοσης. Το ρώτησα αυτό και στους άλλους υποψήφιους. Κοιτώντας τις αιτήσιες εκθέσεις, την αιτήσια εκθέση που δημοσιεύθηκε φέτος για το 2012 το όραμα του Ευρωπαϊκού Ελεκτικού Συνεδρίου είναι καταστροφικό σε ό,τι αφορά την επόμενη δημοσιονομική περίοδο μέχρι το 2020. Οι κανόνε είναι πολύ περίπλοκοι φυσικά, αλλά δεν υπάρχουν σχεδόν καθόλου συγκεκριμένοι στόχοι βάσει των οποίων θα μπορέσουμε να προσμετρήσουμε την απόδοση. Θα ήθελα να μας πείτε ότι θέλετε να επικεντρωθείτε πιο πολύ σε θέματα απόδοσης και μπορεί να το δηλώσετε αυτό, αλλά πώς μπορούμε να μεταφράσουμε καλύτερα τις συστάσεις ε, του ελληνικού Συνεδρίου σε πράξη. Αυτό θα πρέπει να μας απασχολήσει και εμάς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όχι απαραίτητα στην Επιτροπή μας, αλλά και σε άλλες επιτροπές. Συχνά δεν ακούμε απαραίτητα το τι λένε οι ειδικέ εκθέσεις και οι άλλες εκθέσεις του Ευρωπαϊκού Ελεκτικού Συνεδρίου. Ίσως λοιπόν θα θέλατε να μοιραστείτε κάποιες σκέψεις μαζί μας για το πώς μπορεί να υπάρξει μεγαλύτερη επιρροή του έργου του Ελεκτικού Συνεδρίου. Ευχαριστώ, ο κύριος Οντή. Ευχαριστώ. Θα ήθελα και εγώ και εκ μέρους του ΕΛΚΑ να ευχαριστήσω και να καλωσορίσω τον κύριο Owen ε, να τον ευχαριστήσω για τις διευκρινήσεις που μας έκανε σε σχέση με τις ερωτήσεις που του υποβάλαμε και γραπτός. Διαπιστώσαμε ότι στα διαδρομή σας ε, ε, εντοπίζετε κυρίως στη δημόσια διοίκηση και ούτε από τις σπουδές σας ούτε από την εμπειρία σας βλέπουμε να έχετε κάποια προσόντα δημοσιονομικού ελεκτή. Μπορείτε λοιπόν να μας καθησυχάσετε ότι έχετε τα προσόντα για να αναλάβετε την ιδιότητα τη θέση του μέλους του Ευρωπαϊκού Ελεκτικού Συνεδρίου. Επίσης, από τη στιγμή που η καριέρα σας ήταν ε, στη δημόσια διοίκηση, σίγουρα στους διορισμούς και στις προαγωγές είχατε κάποια σχέση με την πολιτική εξουσία. Μπορείτε να μας διαβεβαιώσετε για την ανεξαρτησία σας ε, και να συμπληρώσετε την ερώτηση αυτή ως προς την ανεξαρτησία που θα πρέπει να δείξετε απέναντι στην Βρετανική κυβέρνηση. Τέλος, στην τελευταία σας γραπτή απάντηση, εκεί που απαντήσετε αν θα αποσύρατε την υποψηφιότητά της σε περίπτωση που είναι αρνητική γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η απάντηση είναι κάπως συγκεχημένη, δεν είναι και πολύ σαφής. Μπορείτε να μας απαντήσετε κάπως πιο ρητά, γιατί έχουμε μακροχρόνια ε, εμπειρία με τέτοιου είδους ε, αφήσιμες απαντήσεις. Μπορείτε λοιπόν να μας δώσετε μια ξεκάθαρη απάντηση για να ξέρουμε κι εμείς ε, που βρισκόμαστε στο θέμα αυτό. Σας ευχαριστώ και ο Γιάννη Μιλντερ είναι ο τελευταίος εδώ στον κατάλογο μου. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα κι εγώ να μου δώσετε λίγο παραπάνω πληροφορίες για το θέμα που έδειξε ήδη ο κύριος Οντή. Σε περίπτωση αρνητικής γνωμοδότησης από πλευρά μας, αναφέρεται ότι στην ε, περίπτωση αυτή θα εξετάσω σοβαρά το ενδεχόμενο να αποσύρω την υποψηφιότητά μου. Θα πρέπει να διαβουλευτώ με την κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου και θα πρέπει να γνωρίζω τους λόγους που οδήγησαν στην αρνητική γνωμοδότηση από πλευρά τη Επιτροπής Αλέγχου του Προπολογισμού. Η ψηφοφορία, ξέρετε, είναι μυστική. Τι θέλετε να σας εξηγήσω εκ των υστέρων σε περίπτωση απόρριψης πώς και γιατί ψήφισα αυτό που ψήφισα. Και πραγματικά ε, περιμένετε ότι εγώ ή οποιοδήποτε άλλος εδώ στην Επιτροπή θα το κάνω αυτό. Πώς θέλετε δηλαδή να λάβετε τους λόγους για την απόρριψή σας. Πώς θέλετε να γνωρίζετε τους λόγους αυτούς. Αυτή είναι η ερώτησή μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Η κυρία Γκρέσλε, κλείνοντας, ευχαριστώ πάρα πολύ. Είπατε ότι θα διαβουλευτείτε με την κυβέρνησή σας σε περίπτωση μία αποδοχή στις υποψηφιότητά σας. Τι γίνεται σε ό,τι αφορά τις υπόλοιπες διαβουλεύσεις με την κυβέρνησή σας. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ, λέει ο πρόεδρο, Ολόκληρη δέσμη ερωτήσεων. Δεν ζητά κανεί άλλο το λόγο. Να δώσω το λόγο στον κύριο Όουεν για να απαντήσει. Θέλουμε να ακούσουμε τις ευχέστατε απαντήσεις σας. Ε, εγώ έτσι κάνω χιούμορ, συγγνώμη. First of uh, I will begin with report. Θα κάνω ό,τι μπορώ κύριε Πρόεδρε ξεκινώντας με τις ερωτήσεις της συγκεκριτρίας για την ε, δουλειά μου στο NAO. Είχε ιδιαίτερη σημασία όταν διορίστηκα να ε, ενημερωθώ, να εμβαθύνω, να βελτιώσω τις γνώσεις και την εμπειρία μου και ιδιαίτερα είδα και παρακολούθησα με προσοχή το πώς ε, διοικείται ένας ελεκτικός οργανισμός, έχω συμμετάσχει σε σεμινάρια κτλ. Έχω κάνει πέραν της, και μαζί με την γεωργική ομάδα ελέγχους αποδοτικότητας, μαζί με την ε, ομάδα εσόδων, έχω κάνει σεμινάριο για τις μεθοδολογίες, στατιστικές μεθοδολογίες για τη δειγματοληψία μαζί με κάποια μέλη του ελεκτικού συνεδρίου που είχαν έρθει ως επισκέπτες. Έχω λοιπόν μια σειρά από ε, εμπειρία τέτοιου τύπου. Και έχω πρακτικά παραδείγματα για το, για το πώς ε, στην πράξη μπορούμε το ποσοστό του σφάλματος να το μειώσουμε στο 2% ή περισσότερο με τον δημοσιονομικό ελεγχό. Και νομίζω ρωτήσατε γιατί αν είχα πάει στο London Business School, με συγχωρείτε αν δεν κατάλαβα καλά την ερώτηση σας, που σπούδασα στο London Business School. Λοιπόν, επειδή ήμουν στο δημόσιο, ε, θέλησα να μάθω περισσότερα πράγματα για το πώς ε, λειτουργεί το κράτος και όχι μόνο δημοσιονομικά και διαχείριση λογαριασμών, αλλά στρατηγική, μακρο-μικροοικονομία, ε, marketing. Πολλά ήταν τα μαθήματα που διδάχθηκα και τα οποία έχουν σχέση με την δουλειά ενός σύγχρονου λεκτικού οργανισμού και ιδιαίτερα στην, στον έλεγχο αποδοτικότητας που γίνεται μέσα σε ένα κόσμο πλέον πολυτομεακό. Όπως άλλωστε καταγράφονται και στις δικές μας ε, ε, στις δηλώσεις ε, του ECA χρειάζεται κανείς να έχει πολλές δεξιότητες και γνώσεις για την έγκριση κοινοτικών κονδυλίων στα κράτη-μέλη. Το Ηνωμένο Βασίλειο πριν από μερικά χρόνια έκανε ένα πείραμα με τη δημοσίευση δημοσίων λογαριασμών, ελεγμένων ε, λογαριασμών ε, ευρωπαϊκών. Δυστυχώς αυτή η πρακτική όμως σταμάτησε για λόγους τεχνικούς, ε, απουσίας γνώσεων. Αν και έχει δεσμευθεί να ξαναρχίσει σύντομα η κυβέρνηση, ελπίζουμε το 2014 ή 2015 να το δούμε. Εγώ τουλάχιστον αυτό ελπίζω. Ε, και, εκ της, και για την Ένωση πιστεύω θα ήταν κάτι το πολύ θετικό. Βέβαια κάθε Υπουργείο το οποίο διαχειρίζεται ευρωπαϊκά κονδύλια θα πρέπει να εξετάζεται χωριστά ασφαλώς. Δεν είναι το ίδιο με τη διαδικασία της επίσημης έγκρισης των ε, λογαριασμών. Εδώ έχουμε να κάνουμε μια ενοποιημένη έκθεση των ε, δημοσιονομικών, των λογαριασμών του κάθε Υπουργείου και το, ο κάθε ελεγκτής που έχει αναλάβει το κάθε Υπουργείο, όπως άλλωστε είχα εγώ ε, την ευθύνη της ενέργειας και του κλίματος ε, για ένα διάστημα, έχει κάνει χωριστά την αξιολόγησή του και έχει δώσει το πράσινο ή το κόκκινο φως εκ μέρους της Εθνικής Αρχής. Αυτό που έχω να πω εγώ είναι για την περίοδο στην οποία βρισκόμουν επικεφαλής ε, του τομέα ενέργειας και κλίματος. Ε, ε, προχώρησαν σε έλεγχο στη συνέχεια από το νέο αρμόδιο χωρίς κανένα σχόλιο. Επικυρώθηκαν δηλαδή χωρίς κανένα σχόλιο. για το σύστημα υγείας. Το σύστημα υγείας και το έργο που προσφέρει άπτεται της υγείας, της ποιότητας ζωής όλων των πολιτών μας, κυρίως όταν βρίσκονται, ε, όταν έχουν προβλήματα υγείας. Πρέπει λοιπόν και η εκτελεστική εξουσία και ο ελεγκτικός μηχανισμός να ε, προβαίνουν σε μία ε, συνεργασία χωρίς προβλήματα και όταν κάποιος συμμετέχει σε ένα διοικητικό συμβούλιο θα πρέπει να αποζημιώνεται για να μην υπάρχει κίνδυνος ε, ε, διαφθοράς. Αυτό ισχύει για μένα ως προς το μισθό που εισπράττω από το νοσοκομείο, από το νοσοκομιακό σύστημα. Έγινε μια ερώτηση για τον προπολογισμό από το Υπουργείο στο οποίο ήμουν εγώ υπεύθυνο για τον προπολογισμό το σχετικό με τον πυρηνικό αφοπλισμό ο οποίος ε, μας κοστίζει κάποια δισεκατομμύρια κάθε χρόνο σε εγκαταστάσεις όπως αυτές του Σέλαφιλ, παράδειγμα, που έχουμε να κάνουμε και με πολύ ψηλό κίνδυνο και με ε, θέμα ασφάλειας πυρηνικής αλλά και οικονομικής, είναι ένα ζήτημα το οποίο θέλει πολύ προσθερή μελέτη. Άλλωστε χαίρομαι που μπόρεσα να συλλέξω τη σχετική ε, γνώση και ίσως οι γνώσεις μου και από τον τομέα της ε, κλιματικής αλλαγής και της ενέργειας ε, να αποβούν χρήσιμες. Θα ήθελα επίσης να επισημάνω στον κύριο Βόνο ότι είμαι ανεξάρτητος και ουδέτερος. Έχω εργαστεί και για συντηρητική κυβέρνηση και στο, Επιτελείο Υπουργού των Οικονομικών Συντηρητικής Κυβέρνησης και για τους εργατικούς και την κυβέρνηση ε, έχω εργαστεί υπό Υπουργό Εργατικό και ως ειδικό σύμβουλος και ως ε, ε υφυπουργός ε, με τον ε, τωρινό επικεφαλής της αντιπολίτευσης του Ρωμανού Βασίλειο και έχω συνεργαστεί με τους ηγέτες ε, του τωρινού κυβερνητικού συνασπισμού, συντηρητικούς δηλαδή και φιλελευθέρους, χωρίς κανένα μια δυσκολία. Νομίζω ότι αυτό αποδεικνύει την εξαρτησία μου και την, τις υπηρεσίες που μπορώ να προσφέρω σε μια δημόσια υπηρεσία και ακολουθώ, όπως είπα, τις ε, αρχές των διακηρύξεων της Λίμα και του Μεξικού. Με ρωτήσατε επίσης για τη διαδικασία του δημοσιονομικού ελέγχου και την ε, διάχυση των ε, βέλτιστων πρακτικών. Νομίζω ότι θα πρέπει κυρίως με θετικά, αλλά και, και με θετικά κίνητρα, αλλά και με αντικίνητρα να επιδιώκουμε την βελτίωση της ε, απόδοση των λογαριασμών. Θα πρέπει να βοηθήσουμε τους ε, υπαλλήλους, το προσωπικό που διαχειρίζεται τους λογαριασμούς να κάνουν πιο καλή δουλειά. Και στους ανεξάρτητους οργανισμούς στους οποίους έχω εργαστεί είχαμε είχαμε για 20-25 χρόνια ποσοστό χαμηλό, πολύ χαμηλό σφάλματος. Τώρα έχουμε φτάσει στο 1%, 1 περίπου, το οποίο είναι μηδαμινό. Και βέβαια πάντα εξετάζουμε τι είδους βελτιώσεις μπορούν να γίνουν ε, μπορούν να γίνουν σε κάθε περίπτωση. Εγώ νομίζω ότι η ανάλυση των λογαριασμών και ιδιαίτερα σε θέματα, σε μεγάλους κλάδους όπως αυτού ή των ε, δημόσιων λογαριασμών, των δημόσιων προμηθειών, θα πρέπει να αναλύονται κατά από πολύ προσεκτικό και κατά, κατά τμήματα ώστε να εντοπίζονται πολύ πιο συγκεκριμένα τα προβλήματα. Για τον κύριο Κερμπράντη μιλήσατε για τις εκθέσεις αποδοτικότητας. Ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση. οι στόχοι προσδιορισμού για, τους, ε, για το προσωπικό προλαμβάνει αυτό το καθήκον είναι δύσκολη, το ξέρω πολύ καλά και από προσωπική πείρα, αλλά ουσιοδέστατοι. Η παραδείγματι, η αξιολόγηση στην δουλειά της Ένωσης, που πιστεύω ότι αν γίνει σωστά μπορεί να προσφέρει μια πλατφόρμα για καλύτερο, καλύτερη διαχείριση αποδοτικότητας για το μέλλον και ελπίζουμε βελτίωση στις αιτήσιες εκθέσεις των γενικών διευθυντών που θα πρέπει να είναι ε, στηριγμένοι στους στόχους και την αποδοτικότητα. Δουλειά δεν μπορούμε να κάνουμε αν δεν έχουμε μια πλατφόρμα στόχων και δικτών που θα πρέπει να επαληθεύονται και ελπίζω αυτό να βελτιωθεί στο μέλλον αλλά και παρακαλώ και εσείς να επιμένετε γι' αυτό, αλλά χαίρομαι που έχει την μονάδα αξιολόγηση επιπτώσεων τώρα το Κοινοβούλιο που θα κάνει αυτή τη δουλειά. Πώς θα έχουμε καλύτερα αποτελέσματα με βάση την έκθεση της συστάσης κατά της CCA. Νομίζω ότι πρέπει απλώς να επιμείνουμε στο να δοθεί συνέχεια. Έχουν κίνη προτάσεις για την παρακολούθηση των εξελίξεων και σε αυτό θα επιμείνω για τα επόμενα χρόνια. Για να διαπιστώνετε δηλαδή αν έχουν ε, υλοποιηθεί οι συστάσεις ή όχι. Για τις ε, δεξιότητες, της γνώσης κύριε ότι όχι, ξέρετε, έχετε δίκιο σε αυτό, δεν έχω ε, κατάρτιση δημοσιονομικού ελεγκτή. Έχω όμως εμπειρία αρκετή από το δημοσιονομικό έλεγχο και νομίζω ότι μπορώ να έχω αντίληψη. Βέβαια έχω μελετήσει τη, στη ε, London Business School τι ε, τις βασικές αρχές του, των λογιστικών, του δημοσιονομικού ελέγχου. Μπορώ να διαβάσω έναν ισολογισμό ε, και ξέρω τι σημαίνει και το ουσιαστικό στατιστικό σφάλμα και το μηδαμινό σφάλμα και πώς αξιολογούνται οι στατιστικές και όλα αυτά. Και επιπλέον αυτού εγώ εκ είμαι υπέρ της διαβίου μάθησης και από ό,τι φαίνεται το συνέδριο προσφέρεται τις ευκαιρίες για βελτίωση των γνώσεων. Για ήταν εξαρτησία που ε, είχε ρωτήσει ο κύριος Φόν νομίζω ήδη απάντησα. Και κάτι ακόμη για την τελική απάντηση στο ερωτηματολόγιο. Νομίζω ότι είναι σαφής η απάντησή μου. Είναι ουσιώδες η σχέση μεταξύ Κοινοβουλίου και Ελεκτικού Συνεδρίου να είναι αμοιβαία, με αμοιβαίο σεβασμό, αποτελεσματική εάν ε, απορρίψετε την υποψηφιότητά μου, ε, με μεγάλη σοβαρότητα θα εξετάσω εάν θα πρέπει να αποσύρω την υποψηφιότητά μου. Θα πρέπει να διαβουλευθώ με τη Βρετανική κυβέρνηση και αυτό θα πρέπει να σας το εξηγήσω. Και αυτό θα πρέπει να εξηγήσω, να συζητήσω μαζί τους για να μπορέσω να δω πώς θα ανταποκριθώ καλύτερα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μια ερώτηση από τον κύριο Μίλτερ και άλλη μια από τον κύριο Οντί. Και στη συνέχεια θα κλείσουμε στην περίπτωση που θα έχουμε αναταραχές. Παρακαλώ να προσταθείτε. Γιάν. Ναι. Θέλετε να καταλάβετε, λέτε, τους λόγους σε περίπτωση που απορρίψουμε την υποψηφιότητά σας. Πώς, λοιπόν, θέλετε να καταλάβετε αυτό. Θέλετε να σας αποκαλύψουμε τη μυστική ψηφοφορία. Αυτό δεν καταλαβαίνω. Θέλετε να απαντήσετε. Όχι, να ακούσουμε για τον κύριο Οντή, λέει ο Πρόεδρος. Στο ίδιο πνεύμα, να μην παίζουμε τώρα το παιχνίδι της γάτας με το ποντίκι, έχουμε πια αρκετές δυσάρεστες και κουραστικές εμπειρίες. Λοιπόν, ε, πείτε μας ξεκάθαρα, εάν ένα αποσύρετε την υποψηφιότητά σας, αποσύρετε την. Είδαμε με τον... Ε, ε, Κροάτι υποψήφιο και είμαι πολύ χνευρισμένος με τον Κροάτι Πρωθυπουργό, ο οποίος δεν έλαβε στο πνεύμα μιας κοινοτική ε, ε, λογικής και συνεργασίας ε, υπόψη την ψήφο του Κοινοβουλίου και μας επέβαλε τον Κροάτι υποψήφιο παρότι τον είχαμε καταψηφίσει. Και το ίδιο θα κάνει και ο Πρωθυπουργό σας εάν τελικά έρθει αυτή η στιγμή έτσι δεν είναι, θα μας επιβάλλει αν, ακόμα και αν σας έχουμε αποσύρει. Εάν έχετε λάβει αρνητική ψήφο, ε, αποσύρτε την υποψηφιότητά σας. Εάν είναι να αφήσετε την απόφαση στα χέρια του Πρωθυπουργού σας, πείτε μας το έτσι. Ή αποσύρεστε ή αφήνετε την απόφαση στον ε, Πρωθυπουργό για να ξέρουμε τι έχουμε να κάνουμε και τι να περιμένουμε. Okay. Μάλιστα. Δύο ερωτήσεις. Ε, ας ακούσουμε δύο απαντήσεις. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Νομίζω ότι τοποθετήθηκα με σαφήνεια, με ειλικρίνεια και ανοιχτό πνεύμα στην καλύτερη, με την καλύτερη, στην καλύτερη επίπεδο που μπορώ και γραπτά και προφορικά. Αλλά να επεξηγήσω το εξή. Ω δημόσιο ε, υπάλληλο και ω ολεκτής ε, έχει καθήκον κανείς να εξετάσει όλα τα στοιχεία όλα τα δεδομένα που έχει στη διάθεσή του πρωτού λάβει μία απόφαση στη δική μου εμπειρία πλέον των 30 ετών είναι καλύτερο να μην απαντάμε σε υποθετικές ερωτήσεις για το πώς ενδεχομένως να αντιδράσει κανείς σε ένα μελλοντικό ε, σενάριο με κατηγορηματικό τρόπο. Θα προσπαθούσα να μάθω πιο πολλά με οποιοδήποτε τρόπο το κατάφερνα για την απόφαση που θα ε, είχε ληφθεί. Σε περίπτωση που ληφθεί μία τέτοια απόφαση από την Επιτροπή και από την Ολομέλεια και νομίζω ότι αυτό είναι λογικό Δεδομένου και τον τρόπο που λειτουργώ ως δημόσιος υπάλληλος, θεωρώ ότι θα έπαιρνα την απόφαση η οποία θα ήταν δική μου, θα την ελάμβανα στη συγκεκριμένη χρονική συγκυρία βάσει των δεδομένων που θα είχα στη διάθεσή μου τότε. Τώρα, για το λόγο για τον οποίο θα διαβουλευόμουν με την κυβέρνησή μου, κοιτάξτε, είμαι υποψήφιο τη κυβέρνησή μου. Είμαι ευγνώμων για την υποψηφιότητά μου. Θα ήταν λοιπόν, ε, θα ε, συνάδει με τις αξίες μου το να διαβουλευτώ μαζί τους. Σας ευχαριστώ πολύ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Όουεν για την απάντηση στα ερωτήματα αυτά. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω. Θα συνεχίσουμε τις διαδικασίες μας εμείς. Ευχαριστώ πολύ. Κυρίες και κύριοι αγαπητοί συνάδελφοι, έτσι ολοκληρώσαμε την πρωινή μας συνεδρίαση. Να διακόψω τη συνεδρίαση στις 3 το απόγευμα. Συνεχίζουμε 15 και 00. Με την έκθεση Sondergaard συνεχίζουμε για τον σεισμό στην Άκυλα στις 3. Σας ευχαριστώ πολύ. Διακόπτω τη συνεδρίαση.